Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα καταρχήν να κηρύξω την έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Το σημείο 2 ανακοινώσεις έχουμε με εξαίρεση τα μαλτέζικα και τα εστονικά όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Berichte von Delegationsreisen, einmal CBD, äh, COP. Τώρα, ανακοινώσεις äh, για τις αντιπροσωπίες. Έχουμε CPD, ε, και την 18η διάσκεψη των μερών για τις κλιματικές αλλαγές. ΔΟΧΑ. Και η δική μας επιτροπή έχει στείλει αντιπροσωπή εκεί. Και μάλιστα τις εκθέσεις των αντιπροσωπιών αυτών θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, για όποιον ενδιαφέρεται. συνέχεια των ανακοινώσεων. Την επόμενη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί, θα λάβει χώρα μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής με τον Επίτροπο Μπόρκ για το σκάνδαλο του κρέατος αλόγους και το πώς παρισέφησε στην ε, επισητιστική αλυσίδα. Επαναλαμβάνω μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 9 με 10 και μισή. Περνάμε τώρα στο, τελευταίο, στο πρώτο και τελευταίο σημείο της που προβλέπει την δημόσια ακρόαση για τα προϊόντα καπνού. Χαίρομαι γιατί έχουμε πολύ σημαντικούς καλεσμένους, έγκριτους εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους της Προεδρίας, της Ιρλανδικής Προεδρίας, τον James Ράιλι, τον Ιρλανδό Υπουργό και τον Αρμόδιο Επίτροπο για Υγεία και Πολιτική των Καταναλωτών, τον κύριο Τόνιο Μπόρκ. Είναι από τα πιο σημαντικά από τα πιο σημαντικά θέματα που έχουν προκαλέσει σφοδρές συζητήσεις και μάλιστα το Κοινοβούλιο ζήτησε εντόνως να λάβει εμπρόθεσμα το συντομότερο δυνατό την πρόταση αυτή για να έχει το χρόνο να προετοιμάσει τη θέση του, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Έχουμε μαζί μας και την κυρία Λίντα Μακάβαν, που είναι σκιώδη συγγήτρια και εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, ή μάλλον η αρμόδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την παρακολούθηση της οδηγίας αυτής για τα προϊόντα του καπνού. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον ε, Ιρλανδό Υπουργό, ώστε να μην χάνουμε άλλο χρόνο και να πάμε κατευθείαν στη συζήτηση. Και σας Παρακαλώ θερμά να τηρήσουμε όλοι το χρόνο αγόρευσης ώστε να έχουμε ευκαιρία και για συζήτηση, να μπορέσουν να υποβάλουν τις ερωτήσεις του συνάδελφοι και να ακούσουν και τις απαντήσεις. 10 με 12 λεπτά έχουν οι καλεσμένοι μας το χρόνο για να μας παρουσιάσουν τα θέματά τους. It's your turn. Είναι η σειρά σας, λέει ο πρόεδρος στον Υπουργό. Uh, uh, θα ήθελα, λέει ο Γιώργος Υπουργός, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που με προσεκάλεσε να σας μιλήσω και να σας μιλήσω και για την Ιρλανδία και για την Ευρώπη σήμερα για τα προϊόντα καπνού αλλά και τις βλάβες που προκαλούν. Επομένως θα πρέπει να αναλογιστούμε το μέγεθος της βλάβης που προέρχεται από το κάπνισμα, αλλά και την οικονομική ζημία επίσης που βαρύνει την Ευρώπη. 700.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αιτίες από που έχουν σχέση με το κάπνισμα. Μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία. Χειρότερα από παχυσαρκία, ε, από το αλκοόλ και έχουμε ζημιά 5,3 δις ευρώ ετησίως. 8,3 δις ευρώ ε, χάνονται από αυτούς που απουσιάζουν τη δουλειά, αυτούς που παίρνουν πρόορη σύνταξη λόγω του καπνίσματος. Οπότε βλέπουμε πόσο ζημιά προκαλεί παντού και σε όλους το κάπνισμα. Και όλοι γνωρίζουμε ότι η μισοί από τους ε, μακροπρόθεσμα καπνιστές πρόκειται να πεθάνουν και σήμερα με τα στατιστικά του ΠΟΗ έχουμε 100 εκατομμύρια θανάτους έχει προκαλεί στο κάπνισμα στον 20ο αιώνα. Και πάμε για ένα δις τον 21ο αιώνα. Δεν είναι εδώ να επιτρέψουν να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Το Ευρωβαρόμετρο έχει εξηγήσει ότι 60% των Ευρωπαίων καπνίζουν και η Ιρλανδία βρίσκεται στο 29% όσον αφορά τους καπνιστές δηλαδή, όπως είναι ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός. Αυτό είναι απαράδεκτο, η νοικοτήνη είναι πάρα πολύ θυστική ουσία και μόλις εθιστούν σε αυτήν ενήλικοι και έφηβοι είναι παγιδευμένοι 70% των καπνιστών στην Ευρώπη άρχισαν να καπνίζουν όταν ήταν νέοι. Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να είναι λιγότερο ελκυστικό το κάπνισμα στου νέου. Είχαμε 78% των Ιρλανδών που είπαν ότι ξεκίνησαν όταν ήταν κάτω από 18. Τι μπορούμε να κάνουμε επομένω για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ε, κοινωνία για, για αυτή όλη τη ζημιά και οικονομική και άλλο. Πώ θα αποθαρρύνουμε τον κόσμο να καπνίζει. Τότε που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο ήμουν αποφασισμένο να αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Η ιδέα οδηγία για το προϊόντα καπνό είναι η βασική προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Κανένα μέτρο από μόνο του δεν μπορεί να μειώσει τον αριθμό των καπνιστών και των ανηλίκων που να καπνίζουν. Αλλά χρειάζεται συνδυασμό μέτρων, αποτελεσματική νομοθεσία, συνολική υποστήριξη αυτού που προσπαθούν να κόψουν το κάπνισμα και επίση εκστρατείε μέσω των σχολείων και γενικότερα. Επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα πάψει να θεωρείται κάτι το φυσιολογικό. Θεωρείται μη φυσιολογικό στην κοινωνία το κάπνισμα και κατά γνώμη αυτό είναι το κλειδί, ούτως ώστε να λυθεί το πρόβλημα για τις επόμενες γενιές και η προεκτηνομένη οδηγία θα είναι ένα εργαλείο κλειδί για να σταματήσουν είναι το κάπνισμα ή να μην το αρχίσουν. Όπως θα αξίσει ο κύριος Μπόρκ, θέλουμε να γίνει λιγότερο ελκυστικό το κάπνισμα, να αποθαρρύνουμε τον κόσμο το να αρχίζει να καπνίζει ιδίως τους νέους, αυστηρότεροι κανόνες. Και αυτό επίσης θα αφορά και το πώς δεν θα είναι ελκυστικό το άρωμα και η γεύση του καπνού. Όπως ξέρετε, ε, θα πρέπει με την οδηγία να ρυθμίσουμε και τα περιεχόμενα, το, το, το, το περιεχόμενο σε νοικοτήνη, παράνομο εμπόριο, την τυχετοθεσία, το, τη συσκευασία με, με χαρακτηριστικά ασφαλείας, οπότε έτσι θέλουμε να υπάρχει μια συνένεση, να βοηθήσουμε να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη και έτσι να αρχίσουμε τη περίοδο του θέματο που συνεργασία με το Κοινοβούλιο των Ορειτρών Δυνατών. Όπω σα είπα, προσωπικά έχω αναλάβει να αντιμετωπίσω το πρόβλημα, γι' αυτό και θα ήθελα να κάτσουμε και να αναλογιστούμε τι μπορούμε να πετύχουμε, πώ θα φτιάξουμε σε μια κοινωνία ελεύθερη από κάπνισμα χωρίς καπνό και βέβαια αυτό που θέλουμε να έχουμε νομοθεσία όπως έχουμε στη χώρα μας και γι' αυτό και είμαστε από τους πρωταθλητές στον τομέα αυτό και μεταξύ άλλων προσπαθούμε αυτή η πρωτοβουλία του 2004 να επανελθεί το 2007 είχαμε μια νομοθεσία, το 2009 επίσης για τα απαγορεύσεις για, την, για διαφήμιση και επίσης είχαμε και κάποιο μητρό λιανικής πώλησης, απαγόρευση ε, στα, όσον αφορά τις, ε, τις αυτόματες μηχανές πώλησης και επίσης ε, έχουμε για αυτόν τον τρόπο απαγόρευση για πώληση τσιγάρων στους νέους 118 και έτσι να μπορούμε να το αποτρέψουμε τους νέους να αρχίσουν το κάπνισμα και έτσι να μπορούμε συνεχίσουμε την προστασία από την αρχή του αυτού του μήνα. Ε, πακέτα που έχουν λιγότερο από τσιγάρα, Προειδοποιήσει πάνω στο πακέτο. Όλα αυτά θεωρούμε ότι έχουν επιπτώσει θετικές μακρόπονα στους νέους και επίσης σε μια πρόσφατη έρευνα μετρήθηκαν πόσοι νέοι μεταξύ 10 και 17 καμίζουν και το ποστό μειώθηκε από 18% σε 12% το 2010. Παρ' όλα αυτά όμως τα νούμερα είναι εντυπωσιακά ψηλά. Επίσης, τα μέτρα αυτά που έχουμε λάβει διευκολύνθηκαν και από τα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι πάρα πολύ σημαντικό η πολιτική μας σχετική με τον πρόεδρο καπνού καθώς και τον παιδικό πλαίσιο να συνεχίσει και να εξελίσσεται στα πλαίσια της Ένωσης και επίσης μοιρατούμε και άλλα μέτρα ας πούμε, απαγόρευση στα αυτοκίνητα όταν μέσα υπάρχουν ανήλικοι. Επίσης, να προωθούν τσιγάρο και σε άλλες περιοχές όπως σε γήπεδα, πάρκα, ε, επίσης σε, σε, σε περιοχές τέλος πάντων γύρω από το πανεπιστήμιο, φυτικές αισθήσεις, τέλος πάντων ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μία αποτίμηση ότι έχουν πετύχει όλα τα κρατη σε μία σύσκεψη που θα γίνει στο Δουβλίνο τον επόμενο μήνα. Ελπίζω να σας δούμε εκεί και περιμένω πώς και πώς να ακούσω σήμερα τη γνώμη σας και επικοδομητικά να συνεργαστούμε και με την ε, εισηγητρία την Λίντα Μακάβων και να συμφωνηθεί με τους χειώδες εισηγητές σε ένα κείμενο για αυτή την σημαντική οδηγία. Περιμένω να ακούσω και θα πει και ο κύριος Μπόρο και ξέρω και εκείνος έχει δεσμευτεί ε, το εργαλείο δυνατό να κάνει την πορεία για να εγκριθεί αυτό το κείμενο. Γιατί πρέπει να εγκριθεί σύντομα αυτό το κείμενο, μια που κάθε χρόνο πεθαίνουμε με 700.000 συμπολίτε μας. Έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, έχουμε ένα πλαίσιο πολιτικής, το οποίο χρειάζεται ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις ασθένειες που έχουν σχέση με τα προϊόντα καπνού, κυρίες και κύριοι. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι προσπαθούμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, για να προστατεύσουμε τους συμπολίτε μας. Να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από αυτή την δολοφονική συνήθεια. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριε Υπουργέ. Τώρα, Ήρθε να ακούσουμε τον Υπουργό με τον Χαρτοφυλάκιο Υγεία, Κύριε Μπόργκ, έχει το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, Ράιλι, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κύριε και κύριοι. Θα σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για συζήτηση σε μια τέτοια δημόσια ακρόαση την αναθεώρηση τη οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Και γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρέθηκε ε, στο προπύριο αυτής της συζήτησης, ε, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την κοινοτική νομοθεσία των προϊόντων καπνού ε, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι η νομοθεσία αυτός σκοπός. Θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι ώστε να μειώσουμε τον αριθμό των καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να σώσουμε ζωές, ανθρώπινες ζωές. Γνωρίζετε ότι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 700.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από αρρώστιες συναφής με το κάπνισμα. Και ο βασικός στόχος της οδηγίας, πέραν των άλλων θετικών παρενεργειών, θέλουμε να εξασφαλίσουμε, να εξασφαλίσουμε πιο υγιεινή ζωή ε, και μακροβιότητα στους συμπολίτε μας. Αυτό είναι ο στόχος της οδηγίας. Αυτό μου ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό έκανα. Στην ακρόασή μου τον περασμένο Νοέμβριο υποσχέθηκα ότι μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου και το κατάλαβα με την υποστήριξη του κυρίου Μπαρόζο και των υπόλοιπων επιτρόπων στις 19 ε, Δεκεμβρίου, δηλαδή έξι εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι φανταζόμουν να καταθέσω την πρόθεση για την αναθεώρηση της οδηγίας. Ήδη έχει 11 χρόνια ζωής η αρχική οδηγία. Καιρός είναι λοιπόν να την προσαρμόσουμε στις νέες εξελίξεις, στην πραγματικότητα και στις, στα νέα επιστημονικά πορίσματα. Νέα προϊόντα καπνού έχουν ε, εμφανιστεί στην αγορά, μοιάζουν με κραγιόν. Κοιτάξτε. Βλέπετε να μοιάζει αυτό το προϊόν με καπνό, μοιάζει με άρωμα ή μοιάζει με κραγιόν. Ακόμη και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος που ε, έχουμε τη σήμανση του, του προϊόντος ε, είναι διαφορετική. Ένα προϊόν καπνού θα πρέπει να έχει τη γεύση του καπνού και να μην έχει άρωμα γεύση ε, βανίλιας ή άλλου γλυκού. Γιατί λοιπόν λέμε ότι τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να μοιάζουν με καπνό και να έχουν τη γεύση καπνού. Γιατί όπως σωστά είπε ο υπουργό Ράιλι, όλα αυτά τα προϊόντα παράγονται με τρόπο ώστε να είναι ελκυστικά στους νέους. Γιατί γνωρίζουμε ότι συνήθως το κάψιμα το ξεκινάει κανείς ε, όχι στα 50, αλλά πολύ πιο νωρί. κάτω των 25 συνήθω είναι οι καπνιστέ όταν ξεκινά το κάπνισμα, για να μην πω και κάτω τα 18. Και έχουμε και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπω είναι τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα. Ήρθε, είχε δημιουργηθεί ανάγκη να λάβουμε δράση λοιπόν και αυτό κάναμε με την οδηγία. Και εντωμεταξύ και το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα επιμέρου κρατημέλη υπέγραψαν και κύρωσαν την σύμβαση πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης ε, Υγείας για τον έλεγχο του καπνού την σύμβαση SPEC ή FCTC. Κάτι που σημαίνει ότι έχουμε νόμιμη υποχρέωση, ένομη υποχρέωση να, καλύψουμε, να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας για την επισήμανση, συσκευασία, τις, τα αρώματα και τις γεύσεις και τα συστατικά. Γι' αυτό και η πρώτες Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνονται κυρίω στου νέου και νομίζω ότι οι ρυθμιστικέ αρχέ και οι ε, οι νομοθέτες έχουν την ε, υποχρέωση να υποχρεώνουν και να, ε, να προστατεύουν και να αποθαρρύνουν τους νέους να, να ξεκινήσουν το κάπνισμα. Και αν καταφέρουμε την επόμενη πενταετία να μειώσουμε κατά 2%, δηλαδή κατά 1,2 εκατομμύρια τον αριθμό των καπνιστών, θα πρέπει να πράξουμε δύο. Να καταρχήν να πείσουμε τους νέους να μην ξεκινήσουν το κάπνισμα και δεύτερον να πείσουμε αυτούς που έχουν ήδη ξεκινήσει το κάπνισμα να το σταματήσουν. Οι νέοι ξεκινούν το κάπνισμα και θεωρούν ότι είναι cool, ότι είναι μαγκιά και κανείς στη συνέχεια μπορεί να το σταματήσει όποτε θέλει. Και μάλιστα πολλοί από εμά, όσοι ήμασταν πρώην καπνιστές, γνωρίζουν πολύ καλά τι εννοώ. Μετά οι άνθρωποι συνεχίζουν το κάπνισμα γιατί τους γίνεται θυσμός, γιατί μερικές φορές αγνοούμε τον εθιστικό χαρακτήρα και τη φύση του καπνού. Και έτσι δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, λόγω του εθισμού και της εξάρτησης, να σταματήσουν. Οπότε μετά από 30-40 χρόνια μετατρέπεται το κάπνισμα σε καρκίνο, καρδιακές παθήσεις και διάφορα άλλα προβλήματα υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τα 700.000 ε, άτομα που ε, πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο από ασθένειε συναφείς με το κάπνισμα. Είναι δηλαδή σαν κάθε χρόνο να εξολοθρεύεται ο πληθυσμός μιας πόλης σαν τη Φραγκφούρτη το Παλέρμο. Αυτό θέλουμε να ρυθμίσουμε την αγορά του καπνού και των προϊόντων του καπνού για να ξέρουν οι άνθρωποι τι προκαλούν τα προϊόντα αυτά. Αν ε, δει κανεί ένα τέτοιο ροζ πακέτο, ένα τέτοιο πακέτο ωραίο με ε, ροζ ελέφαντες, τόσο ωραίο, με γεύση ή άρωμα φρούτου, μέχρι και πίνα, πίνα γεύση έχουμε. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι πρόκειται για ένα επιβλαβές προϊόν και μάλιστα εθιστικό. Περί αυτού πρόκειται. Τα προϊόντα του καπνού θα πρέπει να έχουν και την εμφάνιση αλλά και τη, γεύση προϊόντων καπνού. Και δεν θα πρέπει να συγκαλύπτονται από εφάνταστες συσκευασίε ή να συγκαλύπτονται από παραπλανητικέ γεύσει. Γιατί γίνονται παραπλανητικά τα προϊόντα. Και περί αυτού πρόκειται. Αυτό το χαρακτήρα έχει η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να ε, εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα καπνού περιλαμβάνουν αρκετέ πληροφορίε για τον αντίκτυπό του στην υγεία, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τεκμηριωμένε επιλογέ και αγορέ. Γιατί πραγματικά μπορεί να, είναι, να σας σοκάρει αυτή η φωτογραφία. Είναι σημαντικό να έχουμε ε, τόσο σοκαριστικές εικονογραφικές προειδοποιήσεις, όπως συμφώνησαν και έχουν κάνει 13 χώρες μέλη. Είναι σημαντικό, παρόλο που είναι συγκλονιστικές τέτοιες εικόνες, αλλά με, και με την, είναι σημαντικό να αναγράφονται στα προϊόντα. Οπότε 75% του κα, αυτού του προϊόντου καπνού, 75% της επιφάνειας της συσκευασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει προειδοποιήσεις, ε, ε, εικονογραφικές προειδοποιήσεις και άλλα. Βέβαια δεν θα πρέπει να υπάρχουν και διαφημιστικά στοιχεία, ούτε ελκυστικές συσκευασίε που να θυμίζουν κραγιόν. Στόχος μας είναι όταν ένας, άνθρωπος, ένας καταναλωτής ε, ε, βλέπει ένα προϊόν καπνού να ξέρει ότι θα είναι επιβλαβές για την υγεία του. Και μετά ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και αποφασίζει αν θέλει να το καταναλώσει ή όχι. Δεν είναι ότι υπαγορεύουμε το κάπνισμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους καπνιστές τι κάνουν. Και βέβαια 30% του πακέτου μένει ελεύθερο για το σήμα, το εμπορικό σήμα της μάρκας του τσιγάρου. Και προαιρετικά μπορούν τα κρατημέλη να έχουν και κενό πακέτο. Συνήθως βέβαια δεν είναι κενό, γιατί περιλαμβάνει και προειδοποιητικά μηνύματα και εικονογραφικές προειδοποίησεις απαγορευτικές. Τώρα Θέλουμε ε, τα προϊόντα καπνού με χαρακτηριστικά αρώματα ή γεύσεις, για παράδειγμα ένα έντονο αρώμα της βανίλιας ή μενθόλης απαγορεύεται. Οτιδήποτε αρώματα γεύσεις ή προσθετικά απαγορεύονται όταν έχουν χαρακτηριστικές γεύσεις, γιατί τέτοιου είδους γεύσεις και αρώματα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους νέους και διευκολύνουν την έναρξη του καπνίσματος. Επίσης, ε, βιταμίνες, καφεΐνη ή παραπλανητικά συστατικά επίσης απαγορεύεται να περιέχονται σε προϊόντα καπνού. Η πρόταση βέβαια δεν ρυθμίζει τα πρόσθετα που είναι απαραίτητα ε, για τη μεταποίηση των προϊόντων καπνού, όπως είναι η ζάχαρη που απαιτείται για να είναι πιο εύγευστος ο καπνός. Μία τέτοια πρόταση δεν κάνει διάκριση μεταξύ επίσης των ποικιλιών του καπνού. Προτείνουμε όμως οποιοδήποτε προϊόν που αυξάνει την τοξικότητα ή την εθιστικότητα να μην ε, επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά. Βέβαια θα χρειαστεί να εντείνουμε το έργο μας στον τομέα αυτό και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τις συζητήσεις για τον εθιστικό χαρακτήρα και την τοξικότητα των προϊόντων καπνού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Επίσης, προτείνουμε να διατηρηθεί η απαγόρευση για τον καπνό που λαμβάνεται από τη μύτη. σνούς γιατί πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε λαμβάνει, η, η Σουηδία είχε ε, λάβει ε, την ε, εξαίρεση για το σνούς υπό τον όρο όμως δεν θα κυκλοφορούσε τέτοιο προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η απαγόρευση ίσχυε πριν την προσχώρηση της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσχυε εδώ και 20 χρόνια. Είχε επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2001 και επίσης ε, επιβεβαιώθηκε και στη συνέχεια από την ομολογία του ΔΕΚ του 2004. Το σνούς δημιουργεί εθισμό, έχει επιβλαβεί αποτελέσματα στην υγεία, ε, πολίτες στη Σουηδία σε πακέτα και γεύσεις που έχουν ως κοινό στόχο τους νέους και έχει τεράστιο ε, δυναμικό παρίσπριση στην αγορά είναι πολύ δελαστικό και το πακέτο και τα ονόματα, όπως το Radical Red, το ριζοσπαστικό κόκκινο. Δεν είναι ότι έχει πολιτική απόχρωση, αλλά είναι ελκυστικό. Ούτε υπάρχουν πορίσματα ή αποδείξει επιστημονικές ότι το ΣΥΝΟΣ βοηθά τον κόσμο να σταματήσει το κάψιμα. Στον Καναδά μειώθηκε κατά 19% το ποσοστό των καπνιστών, 12% στην Καλιφόρνια και 20% στις Ηνωμένε Πολιτείε χωρίς τη χρήση του snus. Τώρα για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η πρότασή μας προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν ένα που ξεπερνούν κατόφλι περιεκτικότητα σε νοικοτήνη χρήζουν άδειε ειδική και κάτω από το κατόφλι αυτό τη περιεκτικότητα σε νοικοτήνη αρκεί η προειδοποίηση της υγείας και όχι η ειδική άδεια. Επίσης, ε, α, απαγορεύεται και προτείνουμε μάλιστα την ε, ενίσχυση των κανόνων συσκευασία και επισήμασης και επίσης μέτρα κατά των παράνομων προϊόντων που περιλαμβάνουν ένα σύστημα εντοπισμού και ένα σύστημα ασφάλειας για το, που περιλαμβάνεται στο ίδιο το προϊόν καπνού. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση δεν επεβαίνουμε στις επιλογές των καταναλωτών, αλλά προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους ευάλωτους, τους νέους, τα παιδιά. Ένα στόχος που θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη νομική βάση της πρότασης. Και με το σχόλιο αυτό θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου για την ταχύρυθμη ε, έγκριση της νομοθετικής αυτής πρότασης στη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα πρώτα στους συντονιστές ή στους εισηγητές για να γίνει συζήτηση και ναι, σκιώδης. Ε, δυστυχώς θα πρέπει να σας περιορίσω σε ένα δίλεπτο γιατί δεν θα λάβουν το λόγο οι άλλοι συνάδελφοι. Γνωρίζω ότι είναι άδικο και είμαι αυστηρός, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ. Η κυρία Μακάβαν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο αλλά και τον Υπουργό που ήρθαν σήμερα να μας επισκεφθούν σήμερα. Σημερινός μου στόχος είναι να ακούσω τους ομιλητές και τους αδέλφους που θα λάβουν το λόγο. Γι' αυτό και σε αυτή τη φάση θα σας τα πω εν συντομία, ότι δηλαδή χαιρετίζω το γεγονό ότι επί τη τραπέζη βρίσκεται αυτή η οδηγία. Όλοι οι συντονιστέ όλων των πολιτικών ομάδων δουλέψαμε σκληρά, ούτω ώστε εγκαίρω να διεκπεριωθεί η οδηγία από το Κοινοβούλιο και ο Υπουργό και ο Επίτροπο εξήγησαν γιατί είναι τόσο σημαντική ε, τούτη η οδηγία. Δεν νομίζω ότι ακόμα και οι πιο φανατικοί καπνιστές θέλουν να γίνουν μάρτυρε όλο ένα και περισσότερων νέων που να καπνίζουν και θέλουμε να σταματήσουν να αρχίζουν από την τρυφερή ηλικία που είπαμε και να έχουμε όλο ένα και λιγότερου καπνιστέ και για μένα τα μέτρα τα οποία προτείνονται από την οδηγία είναι αξιόλογα. Οπότε αυτό που θα επιλέξω είναι να τα προωθήσω ε, από πλευρά πολιτική γωνία δημόσια υγεία και έχουμε διάφορα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και μερικά φρέσκα θέματα. Τα ηλεκτρονικά σιγάρα, ε, το οποίο είναι μόνο το αντιφατικό γεγονό, διαφορετικέ τάσει σε κάθε κράτο μέλο. Θα συζητήσουμε τα θέματα τη συσκευασία, ε, τα θέματα αρώματο και γεύση, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί Πάντως, περιμένω πώς και πώς να γίνει αυτή η συζήτηση και σε υπενθυμίζω σε όλους τους αδέρφους ότι έχουμε σύμβαση πλαίσιο. Το, το ανέφεραν και ο υπουργό και ο Επίτροπος. Και οι εισηγητές δουλεύουν στα πλαίσια αυτής της σύμβασης. Και κάνουμε δημόσιες συναντήσεις με εκπροσώπους της καπνοβιομηχανίας, όπως επιτάσσει σύμβαση πλαίσιο. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους τους βουλευτές. Δημόσιες συναντήσεις. Καταγραφή των όσων λέγονται και διαφάνεια σχέση με το ποιο συναντά ποιον. Γι' αυτό σας περιμένω ανυπόμονα, γίνει η συζήτηση μας προηγούμενους μήνες και οι συνάδελφοι επομένω και αυτοί όλοι να λάβουν υπόψη το πόσο σημαντικό μέτρο αυτό για την δημόσια υγεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, την εισηγήτρια ο κύριος Φλόρενς. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος Κύριε Πίτροπε, ξέρετε εγώ ενδιαφέρομαι και κύριε Προεδρεύον του Συμβουλίου εδώ και χρόνια για τα χημικά που αναμειγνύονται με τον καπνό στα τσιγάρα. Κυκλοφορούν φήμες ότι είναι μέχρι 700 ουσίε, έτσι, χημικές ουσίες. Και εσείς ε, περιοριστήκατε ως προς τα χημικά, στα χαρακτηριστικά αρώματα. Γιατί δεν απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλούστατα κάποιε χημικέ ουσίε που είναι και ε, άκρος και άκρο τοξικέ. Ευχαριστώ κυρία ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με την εισηγήτριά μας την κυρία Μακάβαν και να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και την ίδια ε, για την προσήλωσή της, για το ευήκο και το επικοδομητικό πνεύμα ε, που την χαρακτηρίζει και στη συνεργασία μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό Ράιλι και τον Επίτροπο, ε, με τον Επίτροπο έχουμε Ενεργαστεί πολύ για αυτά τα θέματα και στο παρελθόν με την Ιρλανδία πολύ, με τον Ιρλανδό Επίτροπο αλλά θίξατε το ιερό και όσιο ζήτημα της επικουρικότητας. Ε, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο ε, αυτό όταν υπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι προς έγκριση. Ο Επίτροπος Μπόρτς συνηθίζει να υπενθυμίζει, δεν ξέρω αν το είπε σήμερα, αλλά το έχει πει στο παρελθόν, ότι κανονικά έπρεπε σήμερα να πάρει έγκριση ο καπνός για να κυκλοφορήσει στην αγορά, ε, θα απαγορευόταν τα προϊόντα καπνού, ας πούμε, που αυξάνεται η τοξικότητα, λέτε να απαγορεύσετε, ενός προϊόντος που είναι τοξικό από χέρι. Ε, κανονικά θα πρέπει να είναι πολύ ακραίες ε, οι αποφάσεις σας, ακολουθώντας τα λόγια σας. Ε, εγώ δεν είμαι τόσο ακραία. Κυνηγάμε τώρα το παραμικρό γραμμάριο κρέα αλόγου και βλέπουμε τι γίνεται με τα προϊόντα καπνού. Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι να σκοτώνουμε αδιακρίτω. αυτά. Ήθελα να σα πω ότι θα δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή στα μέτρα που θα καταθέσετε ω προτάσει, να μην μπούμε ακόμα στα τεχνικά ζητήματα. Έχω να κάνω δύο ερωτήσει: μία στον ε, Υπουργό έτσι, γενικότερης πολιτική και στρατηγική ευρύτερα. Κύριε Υπουργέ ε, Ράιλι, εσείς τι περιμένετε Φαντάζομαι ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει πολύ μεγάλους δισταγμού και επιφυλάξει για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως κατατίθεται. Ακούσαμε την πρόταση της Πολωνίας και κάποιων άλλων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει βέβαια ως θεσμικό όργανο σε αυτό το τρίγωνο των θεσμικών οργάνων. Υπάρχουν και τα κράτη-μέλη. Έχετε κάνει τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή και κάτι ακόμα. Ακούσαμε πολλά νούμερα, ε, τελειώνω Πρόεδρε, έχουμε όλοι νούμερα και καταστροφικά στοιχεία για την ε, αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας που είναι δεκαετία, ε, όσο καλύτερος, μάλλον ο καλύτερος νόμος του κόσμου δεν μπορεί να κάνει θαύματα. τι γίνεται με τον Καναδά, με τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, έχουν κάνει καμπάνιες εκστρατείες. Εμείς τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σλούτερς και ο των Πρασίνων. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε. Πάρει πολύ καλά τα είπατε στις προτέσεις σας αυτές. Ε, ε, ε να γίνει δηλαδή αυτό που είπατε ε, υποχρεωτικό όσον αφορά την, την, την, τη συσκευασία. δεν είναι τόσο, τόσο αυτά τα μέτρα. Ε, τόσος κόσμος κινδυνεύει παντού σε όλο τον κόσμο. Επίσης όσον αφορά αυτές τις πρόσθετες ουσίες, όσον αφορά την το να κατονομάζονται, το να δηλώνονται τα αρώματα και οι γέύσει. Συμφωνώ με αυτό, οπότε για να δούμε πω θα μπορούσαμε να πιέσουμε όσο γίνεται περισσότερο προ τα εκεί. Το, για το σνούζ επίση, όσοι δεν είναι Σουηδοί δεν ξέρουν πόσο βαρύνει το θέμα. Είναι βασικό λόγο που προσχωρήσαμε στην Ένωση. Και πάντω ξέρω πολλού Σουηδού που δεν θέλουν να το εξάγουμε. Ε, Υπό οδήποτε μορφή νοικοτήνη είναι κάτι το βλαπτικό. Επίσης, να μην αφήσουμε την αγορά αχαλήνοτη όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, γιατί και εδώ υπάρχει θέμα εθισμού. Άρα, θα πρέπει για ασδήποτε μορφής λήψη νοικοτήνης να διέπεται από νομοθεσία. Τέλος δε, όσον αφορά τη συσκευασία, ναι, για την απαγόρευση των μικρών συσκευασιών, ε, τα, τα άλλα παιχνίδια, τα gimmicks, και τα σχετικά με τη διαφήμιση στα σημεία πώληση, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ δεδομένο. Εάν το αντιμετωπίσετε όλο αυτό, ίσω πάρα πολλέ χιλιάδε θα σωθούν. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσουν να καπνίζουν. Είδατε τι έγινε στην Αυστραλία. Με αυτές τις ε, ελεύθερες τηλεφωνικές γραμμές για του καπνίσματος. Αυτό επομένως είναι καλό και για την υγεία και για την οικονομία το τσιγάρο κάνει κακό στην υγεία και το κακό, και κάνει κακό όμως και στο, και στο γείτονα, κάνει κακό και στο παιδί σου και κάνει κακό και στην οικονομία. Επομένω, οτιδήποτε προσπάθεια για κόψιμο του καπνίσματος είναι καλή επένδυση. Ευχαριστώ Γιάννα Ρόσπαχ, συντονίστρια των ε, συντηρητικών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα τα πω στα δανέζικα. Ευχαριστώ. Άκουσα με προσοχή. Τον κύριο Σλίτερ. Και εμείς Επομένως είναι, είναι πράγμα του διαβόλου η νοικοτήνη και επίσης μπορεί κανείς να οδηγεί να πίνει πολύ με το αυτοκίνητο και είπαμε ότι δεν θα πρέπει να καπνίζει ακόμη και στο αυτοκίνητό του. Όμως, για κοιτάξτε, εσείς προτίθεστε να απεμπολίσετε όλα αυτά τα έσοδα που προέρχονται από το, το προϊόντα του καπνού στη Δανία είναι φοβερή, φανταστική πηγή εσόδων. Εδώ πέρα έχουμε ένα φαρσιασμό, μια, μια υποκρισία που σοβεί. Γιατί ξέρουμε από τη μία πόσο κακό κάνει το κάπνισμα, από την άλλη όμω μεριά είναι πολύτιμα τα έσοδα από τα προϊόντα καπνού και ξέρω τώρα τι κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Και πέραν αυτών επίση, επίτηδε, επίτηδε θέλω είναι προκλητικά. Φυσικά και εγώ θέλω να σωθεί ο κόσμο. Φυσικά και εγώ θέλω να μην καπνίζει ο κόσμος. Όμως, από την άλλη μεριά, έχουμε και το δημοσιονομικό σύμφωνο και έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που ε, περιέχουν νοικοτήνη ε, και ε, δεν είναι και ας μην έχουν καπνό και εγώ είμαι κατά αυτών των προϊόντων όμως αυτό το οποίο θέλω είναι να δούμε τι θα γίνει με την απαγόρευση από την άλλη μεριά όμως όχι μόνο απαγόρευση χρειάζεται και ενημέρωση και νομίζω ότι θα πρέπει ένα ενήλικας να ξέρει αν θέλει ή δεν θέλει καπνό. Να, να αποφασίζει αν θέλει κάτι να κάνει για την υγεία του. Και ξέρουμε ότι είναι αυτό, το ξέρουμε όλοι. Όλοι ξέρουν τι γίνεται, όμω ε, είναι, είναι η δουλειά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει το α ή το β προϊόν. Είναι αυτό ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να απαγορεύσει α πούμε το ενόπνευμα ή οτιδήποτε άλλο. Επομένω, νομίζω θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να προχωρήσουμε. Ο συνάδελφος Ρώση δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και θέλω να σας πω πρώτα πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, νομίζετε ότι είναι σωστό εδώ στο, στην επίσημη έγγραφα της Επιτροπής να έχουμε αυτό εδώ, αυτό το, το, το, το λόγο, αυτό το, τα συνθήματα κατά του καπνίσματος. Εμείς θέλουμε να ακουστούν όλες οι πλευρές. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι δυνατόν στο επίσημο έγγραφο της Επιτροπής μας να έχουμε ένα τέτοιο εξώφυλλο το οποίο αφορά τη μία μόνο πλευρά. Όλοι έχουν δικαιώματα, έχουμε καλέσει κόσμο εδώ. Καλά, ούτε εγώ έχω πότε καπνίσει στη ζωή μου. Αλλά επίση δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να προβούμε σε απαγόρευση. Να προβούμε σε κάποιον να μην καπνίζει, ακριβώ όπω είπε πριν από λίγο η κυρία Ρόσμπαρ με αυτό, με αυτό με προβληματίζει, ότι εάν βάλουμε ένα σωρό περιορισμούς και απαγορεύσεις, γιατί μιλούμε εδώ πέρα για καπνιστές που είναι δεκάδες χιλιάδων. Αν όλους αυτούς τους περιορίσουμε και τους πιέσουμε, ίσως τελικά έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ίσως έτσι έχουμε ξαφνικά λαθρεμπόριο τσιγάρων. Και επομένως δεν θα υπάρχει κανείς έλεγχος στο περιεχόμενο αυτών των λαθρέων τσιγάρων. Άρα, ας πούμε, τα περισσότερα, έρχονται, ξέρω, από την Κίνα. Ποιο ξέρει τι, τι ουσίες, τι πρόσθετα υπάρχουν εκεί μέσα, τι ψεκασμοί έχουν γίνει στη, στα καπνοχώραθα. Σας ρωτώ, κύριε Επίτροπε, ξέρετε ότι 16% των τσιγάρων που κυκλοφορούν σήμερα στην Ευρώπη ε, κυκλοφορούν παράνομα. Ποιο τα ελέγχει αυτά, τι εγγύσει υπάρχουν για την ποιότητά του και Φυσικά συμφωνώ με την ιδέα του να έχουμε ενημερωτικέ εκστρατείε. Θα σα ποτέ μου δεν έχω καπνίσει. Όμω η απαγόρευση είναι παραβίαση προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων. Α, τι γίνεται με τα ενωμένα ποτά. Ας πούμε έχουμε και τα ναρκωτικά που λένε πολλοί συνάδελφοι ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε την κυκλοφορία μερικών αυτών. Άρα θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Ευχαριστώ από την ΚΟΕΣ και όδηση συγγήτρια για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, ναι, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προϊόν το οποίο να κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά και να σκοτώνει έτσι σαν τον καπνό χρησιμοποιούμε ακριβώ όπω προβλέπεται από τον κατασκευαστή του προϊόντο. Οπότε γι' αυτό και μεγάλη μου χαρά άκουσα όσα έχει να μα πει ο Υπουργό ο για την οδηγία για το προϊόντα καπνού που θα είναι υψίστη κορυφαία προτεραιότητα τη Ελλανδική Προεδρία. Κύριε Υπουργέ, σχετικά με αυτό. Για πέστε μας, τι άλλες πρωτοβουλίες έχετε σκεφτεί ούτως ώστε να προωθήσετε το στόχο αυτόν. Είμαι άλλωστε και σε εισηγήτρια και γι' αυτό και με ενδιαφέρει πολύ να παρακολουθήσω τις εξελίξεις. Είμαι και σκιώδης ηγητρευμένος και συμφωνώ με τα όσα είπε η συγγήτρια για το πόσο σημαντική είναι και τι θέματα ρυθμίζει η σύμβαση πλαίσιο. Και φυσικά είναι σωστό να συμμορφωθούμε όλοι. Θα πρέπει επομένως να αναβαθμιστεί, να προσαρμοστεί με τους στόχους μας η δημόσια υγεία αυτή η οδηγία. Και συμφωνούμε με το προηγουμένω σε σχέση με, το, με την υποχρεωτική συσκευασία χωρί τι ενδείξει. Το πακέτο αυτό, mm. Λοιπόν, χωρί φωτογραφίε, χωρί παραστάσει. Θέλουμε επομένω να συνεργαστούμε με του άλλου συζητητέ και να μπορέσουμε κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία να διεκπαιρεωθεί το νομοθέτημα. Βεβαίω και υπάρχουν κάποια προβλήματα θα πρέπει να παρακάμψουμε και πέστε μας σε σχέση με αυτά. Όσο και συζητητρία. Θέλω να κάνω ό,τι πρέπει να το μου για να έχει έσει ο τέλος προσπάθειά μας. Ευχαριστώ. Έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους τώρα για γραμμένο. Θα σας διαβάσω τα ονόματα. Ο κ. Κουμουτσάκος, Λίζε. Σκότα, dann McGuinness, dann Gebrandi, Wilmot, Sanoni, Westlund, Florenz hatten wir schon, Fjellner, Thun und Hohenstein, dann Klaas, Franco und Ayuso. Habe ich jemanden vergessen? Έχασα κανένα όνομα, την Rebecca Harms. Ωραία. Παρακαλώ, ένα λεπτό ερώτηση να κάνετε, αλλιώς δεν θα προκάνουμε και δεν θα ακούσετε απαντήσεις. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Και τώρα ο κύριος Κουμουτσάκοτς, παρακαλώ. Σας βλέπω, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και κύριε Υπουργέ για την ε, πολύ ενημερωτική ε, συζήτηση που ξεκινήσατε. Η πρόκληση της ε, οδηγίας που συζητάμε είναι να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Δηλαδή, να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία ως θεμελιώδη υποχρέωσή μας και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού που είναι επίση θεμελιώδης αρχή της ενιαίας αγοράς, άρα και δική μας αρχή. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε μια συζήτηση με όρους θρησκευτικού φανατισμού για να πετύχουμε ένα καλό νομοθετικό κείμενο. Ακούστηκαν ήδη ορισμένε ορισμένοι προβληματισμοί. Εγώ θα ήθελα να μείνω λιγάκι σε μια συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά, σε μια συγκεκριμένη ρύθμιση που αφορά ε, τις, τα τσιγάρα διαμέτρου μικρότερες από 7,5 mm, τα, τα slim. Αν πρόθεση της οδηγίας είναι να αποτρέψουμε νέους να μπουν στο κάπνισμα και έχουμε μάλιστα εξαιρέσει ορισμέ, μια αλφα κατηγορία, αναρωτιέμαι γιατί δεν εξαιρούμε αυτά τα τσιγάρα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μικρά παιδιά να καπνίζουν slim και εν πάση περιπτώσει, με το να αποτρέψουμε τα σλίμ από κάποιον ήδη καπνιστή, δεν θα τον ρίξουμε στα τσιγάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γκροστέτ. Παρακαλώ. Ένα λεπτό έχετε. Κυρία Γκροστέτ. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομά μου, γι' αυτό ε, πάρα πολύ γρήγορα. για το ηλεκτρονικό σιγαρέτο που είναι τώρα ένα προϊόν για να μπαίνει κανείς στο κάπνισμα, στα τσιγάρα. Και μάλιστα τα αγοράζουν και οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες. Βάζετε ένα κατώτατο κατόφλι για συγκέντρωση νικοτίνης αλλά ε, ε, μάλλον ένα ανώτατο όριο εννοεί η ομιλήτρια, αλλά το υπερβαίνουν κατά πολύ τα τσιγάρα. Για τα αρώματα τώρα, δημιουργούνται καινούργια αρώματα για να προσελκύονται οι νέοι να μπαίνουν στο κάπνισμα. Το μεντόλ ε, λέει δεν είναι ενδιαφέρον για τους νέους ως άρωμα. Ισχύει αυτό. Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για αυτά τα θέματα. Γιατί τα ε, σιγαρέτα μεντόλ μπορούμε να τα διατηρήσουμε, γιατί δεν προσελκύουν και πάρα πολλού νέου. Ευχαριστώ. Πέτρα Λίζε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και οι δύο ήρθατε στο ΕΛΚ και δεσμευτήκατε για την προστασία της δημόσιας υγείας και εγώ συμφωνώ με τα βασικά στοιχεία της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό είναι όμως που έχουμε τώρα πολύ χρόνο να τα συζητήσουμε όλα διεξοδικά. Δύο ερωτήσεις έχω. Θα ήσασταν πρόθυμοι να διευκρινίσετε και να συγκεκριμενοποιήσετε την πρόταση ε, για τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα και μάλιστα τους κινδύνους για τα παιδιά. Γνωρίζουν οι πάντες, ε, οι καπνιστές, ότι το κάπνισμα βλάπτει τη δική τους υγεία, αλλά δεν έχουμε μάλλον καταλάβει πόσο βλαβερό είναι για τα παιδιά. Και προ το παρόν προβλέπεται αυτό στην επιτροπολογία, αλλά μήπω θα μπορούσαμε με τη συναπόφαση να βάλουμε μια ειδική ε, προειδοποίηση. Και το τελευταίο, το δεύτερο ρωτάω αυτό που ρώτησε και η κυρία Γκροστέτ για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ακούω πολλούς πολίτες ότι καπνίζουν τέτοια τσιγάρα για να μην καπνίζουν κανονικά. αυτό είναι μείωση του κινδύνου. Θα μπορούσαμε να το δούμε ως τέτοια, harm reduction. Ευχαριστώ κύριο Σκότα για ένα λεπτό. Κύριε Σκότα, για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Συμφωνώ γενικά με τον απότερο στόχο της πρότασης, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση οι καταναλωτές το πόσο τους βλάπτει την υγεία ο καπνός, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τις οικονομικές πραγματικότητες ε, στο κλάδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται λόγος για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για διατήρηση θέσεων απασχόλησης, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις απομιμήσεις κτλ. Καλό είναι να θέλουμε να μειώσουμε τους καπνιστές στην Ευρώπη, αλλά δεν θα πρέπει να μειωθούν οι θέσεις απασχόλησης, εργασίας. Ε, καλό το γενικό πακέτο, αλλά το γενικό πακέτο χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ε, μπορεί εύκολα να αντιγραφεί. Άρα θα αυξηθεί έτσι το λαθρεμπόριο τσιγάρων και θα έχει και επιβάρηση αυτό δημοσιονομική ως προς τα έσοδα των κρατών. Δηλαδή, θα χάσουν τη δουλειά τους και εκείνοι που εργάζονται νόμιμα, θα αυξηθούν οι κίνδυνοι για την παρανομία και το λαθρεμπόριο. Αυτό είναι κοινοτικοί κανόνες. Είναι προτεραιότητα της Ένωσης να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο τσιγάρο. Η ε, κυρία Μαγκίνες, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Προεδρία και τον Επίτροπο για τα όσα μας είπαν. Νομίζω θα ήταν ανισχυτικό εάν αποφασίζαμε ε, όπως προτείνει ο κύριος Ρώση και κάποιοι άλλοι, ε, γιατί ανησυχούν για τα οικονομικά και τις ε, απώλειες θέσεων εργασίας, να σταματήσουμε δηλαδή να προστατεύουμε τα παιδιά μας από αυτό ε, το θάνατο. Ξέρουμε ότι τα τσιγάρα σκοτώνουν. Ξέρουμε όσοι έχουμε παιδιά ότι δεν θέλουμε να αρχίσουν να καπνίζουμε και έχουμε καθήκον να νομοθετήσουμε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και το λαθρεμπόριο, αλλά μην πούμε ότι δεν μπορούμε να λάβουμε καμία δράση για να αποτρέπουμε ε, κάποιον να μπει στο κάπνισμα για να μην χαθούν θέσεις εργασίας στον κλάδο. Έχει δίκιο η κυρία Μακάβαν να μιλά για τις δραστηριότητε ομάδων πίεσης και λόμπι που θέλουν να συνεχίσει ε, να ισχύει το κάπνισμα. Προσοχή. Ευχαριστώ κύριο Γκερμπράντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τις προτάσεις που κάνετε. Εγώ είμαι πολύ ε, υπέρθερμος ε, υποστηρικτής ε, και αλλάζει και η κοινωνία προς την κατεύθυνση αυτή για την απαγόρευση του καπνού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύετε ότι μπορεί να επιβάλλει πολύ αυστηρά μέτρα κατά του καπνίσματος και από την άλλη να συνεχίσει να επιδοτεί την παραγωγή καπνού και τις καλλιεργείες. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, το υπερασπίσει το ίδιο σώμα ε, επιτρόπων, δηλαδή και τη μία και την άλλη πρόταση. Ευχαριστώ κυρία Γουίλμα. Ε, Ευχαριστώ. Χαιρετίζω την πρόταση, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Θέλω προ... τυποποιημένα πακέτα και συσκευασίε για την απαγόρευση. Νομίζω ότι είναι ε, η μοναδική ευκαιρία που έχουν, ε, δεν είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουν ε, οι καπνοβιομήχανοι. Προτιμώ α, πακέτα χωρίς χαρακτηριστικά, όπως έχουν και στην Αυστραλία. Τώρα, για τα αρώματα και γεύσεις. θα πρέπει να υπάρχει αποκλειστική απαγόρευση για όλες τις γεύσεις, ακόμη και τη ζάχαρη. Να μην είναι εύγευστος ο καπνός. Ε, επίσης, από τη μια επιδοτούμε τον καπνό και από την άλλη έχουμε αυτό αυτόν τον προβληματισμό υγείας. Μερικές φορές είμαστε αντιφατικοί. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να δουλεύουν σε ένα περιβάλλον χωρίς καπνό. Δεν είναι πρόβλημα της Κομισιόν, του Κοινοβουλίου είναι, γιατί ακόμη έχουμε προβουλευτές που υποβάλλουν τους εργαζόμενους ε, στο Κοινοβούλιο σε έκθεση στον καπνό, στα μπαρ και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και πραγματικά αυτό είναι ντροπή. Έσχος. Ευχαριστώ, όλοι, κύριε κύριο Ζανώνη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Υπουργό και τον Επίτροπο. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ακολουθεί τη σωστή πορεία. 700.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους πρόωρα, μάλιστα, και είναι υπερβολικό αυτό ο αριθμός θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να σώσουμε τα παιδιά μας, αλλά να αναλάβουμε δράση για να σώσουμε όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους καπνιστές, αλλά και τους παθητικούς καπνιστές. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τεράστιες εκστρατείες ενημέρωσης και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση και στα σχόλια ενημερωτικές εκστρατείες μεγάλης εμβέλειας γιατί θα πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες για τους κινδύνους. Επίσης, ποια είναι η γνώμη σας ως προς την ανάγκη μιας μεγάλης ενημερωτικής εκστρατείας και για το παθητικό κάπνισμα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι από αυτά που προτείνει η αναθεώρηση της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βέστλουντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση μου είναι απλούστατη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, σέβεται την εξαίρεση που είχε λάβει με την ενταξιακή τη συνθήκη η Σουηδία για το σνούς. Γιατί αν και τα προσθετικά στο σνούς, θα απαγορεύσετε ουσιαστικά ε, de facto την ε, παραγωγή και την εμπορία σνούς. Άρα παρακάμπτεται την σουηδική εξαίρεση με τον τρόπο αυτό. ούτε θα ενθαρρυνθούν οι χρήστες με το snooze. Είναι πολύ διαφορετικές ε, οι, απο... οι πληροφορίες που έχουμε εμείς. Δεν υπάρχουν καν τέτοια πορίσματα επιστημονικά. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Βέστροντ. Εντάξει, θέλετε να κρατήσετε την απαγόρευση για το snooze. Λέτε ότι δεν είναι καλό, ότι προτιμάτε να καταργηθεί πλήρως ο, κα... ο καπνός, αλλά είναι το λιγότερο επιβλαβές ε, ε, προϊόν και είναι το μόνο που απαγορεύεται η Επιτροπή αναγνώρισε ότι 100 με 1000 φορές είναι λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα το σνούς. Φανταστείτε ε, να, να απαγορεύουμε το γαλλικό κρασί και να επιτρέπουμε τη βότκα, τέτοια διαφορά ε, έχουμε. Άλλωστε ε, υπάρχει η δυνατότητα αγοράσης μαροκινού καπνού μάτλα που μοιάζει πάρα πολύ ύποπτα με το σνούς και μάλιστα και στο Βέλγιο κυκλοφορεί. Αν είναι να ε, ρυθμίσετε όλα τα προϊόντα, τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, θα πρέπει να το κάνετε. Για όλα όμως, όχι μόνο για μερικά. Γιατί είπατε Νέα Ζηλανδία, Καλιφόρνια, Καναδάς. Εντάξει, ωραία, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Κοιτάξτε την Ορβηγία και τη Σουηδία. Θα δείτε ότι έχουν τα καλύτερα στατιστικά του κόσμου ε, σε ό,τι αφορά τη μείωση του καπνίσματος. Και επιτρέπεται και την ε, δυνατότητα επιλογής. Οι χώρες αυτές δεν απαγόρευσαν το σνούς. Ευχαριστώ κυρία Τούν. Ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται ανάληψη δράσης προκειμένου να σώσουμε την υγεία των συμπολιτών μας και να αποτρέψουμε τους νέους να αρχίσουν το κάπνισμα στην Κρακοβία έχω εκατοντάδε νέους που έρχονται και παραπονιούνται γιατί εμποδίζουμε την ιδιωτική του ζωή, ε, την ιδιωτική του ζωή, γιατί αυτοί μόνο στα μπαλκόνια λεκαπνίζουν και απαγορεύουμε τη μεθόλη, τη βανίλια, ε, το αλκοόλ, ε, την ζάχαρη, ότι παρεβαίνουμε στη ζωή τους. Αντί για τις απαγορεύσεις, δεν είναι καλύτερο να επικεντρωθούμε στην καλύτερη διαπαιδαγώγηση των νέων αυτών. Ευχαριστώ κύριε Κλάς. Ευχαριστώ. Ακριβώς εκεί θέλω και εγώ να συνεχίσω. Θα πρέπει να ενημερώνουμε, να μορφώνουμε τα παιδιά μας και μετά ο καθένας να αποφασίζει από μόνος του. Ξέρουμε από την εμπειρία ότι το απαγορευμένο είναι γλυκό και τραβάει. Και ε, όταν κάτι το απαγορεύεις είναι ελκυστικό. Λοιπόν, ε, υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν από αρρώστιες που προκαλούνται από το κάπνισμα. Όταν το πακέτο είναι ίδιο για όλους, πώς ε, θα καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο. Και 1,5 εκατομμύριο είναι οι εργαζόμενοι. Έχουμε έσοδα από φόρους. Όλα αυτά είναι βρώμικα λεφτά. Μα ε, είναι νόμιμο προϊόν ο καπνός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, λέει ο κύριος Φραγκό. Ε, Κύριε Επίτροπε, δύο λόγια μόνο, γιατί κάποιοι συνάδελφοι πήραν πάρα πολύ κατηγορηματικές ε, και ακραίες θέσεις, άλλοι ήταν πιο μετρημένοι. Ε, εγώ δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, το έχω ξαναπεί. Ε, είναι σαφές ότι είναι δακτυλοδεικτούμενο σήμερα ο καπνός μαζί με το ινόπνευμα, το γάλα, το γελαδινό, το κρέας. Τίποτα δεν θα καταναλώνουμε πια στην Ευρώπη. Βεβαίως ε, να καταπολεμήσουμε το κάπνισμα στους νέους, αλλά ε, για τα υπόλοιπα α ενημερώνουμε τους πολίτε και ο καθένα ας αναλαμβάνει τι ευθύνε του. Οι ίδιοι που θέλουν οπωσδήποτε να απαγορεύσουν ε, το καπνισμά και τον καπνό ζητούν νομιμοποίηση της κανάβεως. Το είπε για τη Μεθόλη προηγουμένως μία συνάδελφος. Δεν έχουμε αντικειμενικά επιστημονικά στοιχεία και κατανοώ και τους Πολωνούς συναδέλφους. Προσωπικά θα ήμουν πολύ πιο συγκρατημένος. Ευχαριστώ η κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ. Όντως, είναι επιβλαβής ο καπνός για την υγεία, αλλά είναι καλός ε, για τον ε, δημόσιο κορβανά, που 10 δισεκατομμύρια υπολόγισε ο, η Όλαφ ε, της απώλειας. Το άρθρο 14 της οδηγίας δεν ευθυγραμμίζεται με το πρωτόκολλο για την απάλληψη του λαθρεμπορίου προϊόντο καπνού που υιοθετήθηκε το 2012 στη Σεούλ και έχει υπογραφεί από 26 από τις 27 χώρες μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο δηλαδή. Από όλες οι υπόλοιπες έχει κυρωθεί. Η οδηγία στο άρθρο 14 έχει την ευκαιρία να διορθώσει αυτό το πρόβλημα. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνεί με την ιδέα ότι χρειαζόμαστε έναν ενιαίο ε, και ε, ασφαλή κώδικα που θα ενεργοποιείται και θα ελέγχετε από τις διοικήσεις με πλήρη ενημέρωση ώστε να παρακολουθείτε ε, η κυκλοφορία των προϊόντων καπνού σε πραγματικό χρόνο γνωρίζοντα ανα πάσα στιγμή τη νομική κατάσταση και αποθηκεύοντας όλες αυτές τις πληροφορίες για πιθανούς ελέγχους διοικητικούς στη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δεχθεί τροπολογίες για το άρθρο 14 για να ελέγξουμε καλύτερα την απάτη από λαθρεμπόριο προϊόντο καπνού. Η Ρεμπέκα Χάρνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πίτροπε, η δική μου πολιτική ομάδα καλωσορίζει και χαιρετίζει τις προτάσεις σας και λέμε και επιτέλους Εμείς δεν αμφισβητούμε τις αναλύσεις σας για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού, αλλά μετά τη συζήτηση αυτή θα παρακαλούσα και εσείς και η Επιτροπή ε, να κοιτάξει πώς έχουν τα συμφέροντα που κρύβεται από πίσω και είναι πάρα πολύ ισχυρή και πάρα πολύ πλούσια βιομηχανία που στεναρά καταπολεμά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη νιώθουμε αυτή την εξουσία και αυτή θα πρέπει να συνδέεται με τεράστια κέρδη μάλλον. Γιατί η ποσότητα ταμπάκου και ε, καπνού δηλαδή και η ποσότητα ε, των υπολείπων ουσιών που περιέχονται σε ένα τσιγάρο είναι ε, πάρα πολύ δυσανάλογη με το κέρδος που αποκομίζουν οι κατασκευαστές. Πρέπει να καταλάβουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Και ένα άλλο που είπε ο κύριος ε, Λίζε, εάν το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να διώξει τον κόσμο από το πραγματικό καπνό, γιατί θα πρέπει να τους δυσκολέψουμε τη ζωή να ακριβίνει αυτό το τσιγάρο. Σας ευχαριστώ για το ένα λεπτό που τηρήσατε και τώρα ερχόμαστε στις απαντήσεις και θα Ήθελα να πω ότι και αυτή η τελευταία ερώτηση ήθελα να την υπογραμμίσω γιατί την έθεσαν και άλλοι συνάδελφοι για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Έχω πάρει πάρα πολλές επιστολές από πρώην καπνιστές για το ηλεκτρονικό τσιγάρο όπου λέγουν ότι πραγματικά με βοήθησε να κόψω το τσιγάρο. Και αρχίζουν στα 26, 24 μιλιγκράμμ ε, και μετά μειώνεται η νοικοτήνη, αλλά στα 4 μιλιγκράμμ που προτείνει τώρα η οδηγία είναι κοντά στην απαγόρευση. Δεν είναι φάρμακο η νοικοτήνη, αλλά λέτε να πωλείτε στα φαρμακεία ως φάρμακο. Ε, μπορείτε να μας βοηθήσετε, ε, τι επιχειρήματα είναι αυτά για να καταλάβουμε την επιχειρηματολογία σας. Ε, είναι πολύ δυσνόητη και δημιούργησε και τεράστια δυσφορία. Ε, θέλω να δώσω πρώτα το λόγο στον Υπουργό Υγεία ε, της Ιλλανδικής Προεδρία για να απαντήσει και μετά στον Επίτροπο. Ε, Ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Όντως, ένα θέμα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τις χώρες που παράγουν καπνό Πάντως ήθελα να ευχαριστήσω τη Λίντα Μακάβαν για την υποστήριξή τη, τον Καρλ Χάινς Φλόρεντ που είναι υπέρ τη ε, κατάργηση των τοξικών προσθετικών ουσιών. Θα αφήσω την Κομισιό να απαντήσει, αλλά μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για μια ε, οδηγία που είναι συμβαστική λύση. Δεν είναι αρκετά φιλόδοξη για πολλού και για μένα το ίδιο, αλλά προτιμώ να είμαι ρεαλιστή, πραγματιστής, ε, να λαμβάνω υπόψη το εφικτό. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε θα πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί. Φυσικά θα προτιμούσα κάτι πιο φιλόδοξο, αλλά προτιμώ να ε, ε, επιλέξουμε κάτι εφικτό. Έχουμε 700.000 συμπολίτε μας που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Θα πρέπει να ε, δράσουμε άμεσα. Με εντυπωσίασε η δήλωση της, ε, Ιταλής, ε, της Πολωνέζας Υπουργού ότι 90.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ε, το χρόνο στην Πολωνία από ασθένειες συναφής με το κάπνισμα. Είναι τεράστιος αυτός ο φόρος ζωής. Πρέπει να δημιουργηθεί μια οικονομία και πέρα του καπνού. Αυτή η πρωτοβουλία βέβαια θα χρειαστεί χρόνια για να λειτουργήσει, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε την κατάσταση και θα πρέπει να βοηθήσουμε ακόμα και τις οικονομίες που είναι εξαρτημένες από τον καπνό να απεξαρτηθούν. Δεν νομίζω ότι είναι επιλογή σωστή αυτή να ε, μην επιλέγουμε τη ζωή του συμπολίτη από τα συμφέρον των, της καπνοβιομηχανίας. Για το, τη συσκευασία και την επισήμαση συμφωνώ με την πρόταση, αλλά αν θέλουμε συμβαστική λύση νομίζω ότι η οδηγία τη δίνει. Δεν θέλουμε να καταργήσουμε το κάπνισμα στα αυτοκίνητα. Μόνο όταν ε, στα αυτοκίνητα ε, υπάρχουν και παιδιά δεν θα πρέπει να τα υποχρεώνουμε να εγκλωβίζονται σε ένα μικρό χώρο με μια τέτοια καρκινογόνο ουσία όπως είναι ο καπνός. Για τα παιδιά ενδιαφερόμαστε περισσότερο. Οι ενήλικες έχουν την ελευθερία επιλογής. Δεν ε, πειράζουμε την ιδιωτική του σφαίρα. Αλλά δεν θα πρέπει στη, ασκώντας αυτό το, την κακή του συνήθεια να επηρεάζουν και άλλους. Και μάλιστα ιδιαίτερα παιδιά που δεν έχουν την ε, νόμη ηλικία και τη δικαιοπρακτική βούληση να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Οπότε έχουν καμία επιλογή τα παιδιά και τους δημιουργούμε εθισμό χωρίς να τα έχουμε ρωτήσει, χωρίς να έχουν καμία επιλογή. Θέλουμε να τα προστατεύσουμε. Ούτε απαγορεύουμε το κάπνισμα, κύριε Ρώση, ούτε είμαστε α, ε, αντικαπνιστές. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους καπνιστές. Είμαστε ε, κατά του καπνίσματος ή κατά των καπνιστών. Τώρα για την εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι όντω πρόβλημα δεν παρεμβαίνουμε στα δικαιώματα των ανθρώπων. Περιχαρακώνουμε και προστατεύουμε τα δικαιώματα κάποιων πιο ευάλωτων, όπως είναι τα παιδιά. Και ευχαριστώ και την κυρία Άντερσον για την υποστήριξή της. Αναφέρθηκε σε πολλές πρωτοβουλίες που χρειάζονται για να ενισχυθεί η κατάσταση. Θα... Ε, έχουμε προγραμματίσει άλλες 10 συναντήσεις για το θέμα αυτό στη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας και την επόμενη εβδομάδα θα συναντήσω πολλούς υπουργού Υγεία. και θα αξιοποιήσω κάθε ευκαιρία διαβουλεύσεων για να θαρρύνω και τους υπόλοιπους υπουργού ε, να φροντίσουν να υποστηρίξουν οι κυβερνήσει στην πρόταση. Γιατί υπάρχει καλύτερος τρόπος ε, για την πρόοδο μιας οικονομίας από την πώληση μιας καρκινογόνου ουσίας. Αναφέρθηκαν ε, τα σε αυτά τα λεπτά πουράκια Μα δεν. Εκεί είπατε ότι δεν στοχεύουν στου νέου. Μα αντίθετα, στου νέου κυρίω στοχεύουν. Είναι πολύ ελκυστική αυτή η συσκευασία και το, έχει και ακόμη και ωραία ονομασία από ένα γνωστό περιοδικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό θέλουμε εμεί. Αυτό θέλουμε να καταλάβουν όταν ανοίγουν ένα πακέτο τσιγάρων. Να, να ξέρουν τι θα του προκαλέσει την υγεία του. Είναι, δεν είναι σωστό να μην τους προστατεύσουμε. Πίτερ Λίζε μίλησε για τα αρώματα, τις γεύσεις, τα προσθετικά. Αναφέρθηκα πριν στο παθητικό κάπνισμα. Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερες προειδοποιήσεις ε, για το κάπνισμα και για το παθητικό κάπνισμα. Κάποιος άλλος μίλησε πάλι για τα αρώματα και γεύσεις και τα πρόσθετα και υποστήριξε την πρόταση. Ε, είπατε ότι μάλλον δεν έχουμε εμεί τα στοιχεία κατά των αρωμάτων και γεύσεων. Εμείς δεν τα έχουμε, αλλά σίγουρα τα έχουν οι εταιρείες παραγωγής ε, σιγαρέτων και αυτό ακριβώς κάνουν. Κύριε Σκότα. Το θέμα της απάτης και των οικονομικών συνεπειών. Έχουμε 20 δισεκατομμύρια τζίρο από το καπνό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξοδεύουμε 23 δις ε, για την υγεία και χάνουμε ε, επίσης ένα ποσό από τις ε, αρρώστιες, τις αναρωτικές άδειες και τις προώρες δεξιοδοτήσεις. Οπότε ποιος βγαίνει χαμένος. Ποιος θέλει εδώ να μιλάει στα παιδιά του σε 20-30 χρόνια και να ακούει από τα παιδιά κατηγορία ότι παρόλο που ήξερε δεν ανέλαβες δράση. Γιατί α, θα δείτε ότι κάποιο που αγαπάτε ε, και σας είναι πολύ οικείος, ε, ε, κοίτατε σε ένα κρεβάτι και είναι άρρωστος από καρκίνο ή άλλη αρρώστια που συνδέεται με το κάπνισμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, τον εντοπισμό και τις διαδικασίες ασφάλειας, συμφωνώ. Και επίση, όπω είπα και στην αρχή, συμφωνώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να κάνουμε ότι είναι εφικτό και να δεχτούμε ότι έστω και αυτό το βήμα είναι σημαντικό βήμα πρόοδο. Μακάρι να ήμασταν πιο φιλόδοξοι, μακάρι να είμαστε πιο απαιτητικοί, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και έχετε δίκιο. Ο καπνός περισσότερες φορές ε, έχει δυσάρεστη γεύση, γι' αυτό και το μήνυμα του σώματος είναι μην καπνίζεις, δεν σου κάνει καλό. Και κάποιο άλλο είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Και η κυρία Γουάστραντ είπε γιατί δεν, ε, απαγορεύεται και το σνου, δεν αποκλείεται το σνου από την οδηγία. Κάποιο είπε ότι είναι λιγότερο επιβλαβέ. Όπω είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουν σνου ούτε στον Καναδά ούτε στην Καλιφόρνια και κατάφεραν παρόλα αυτά να μειώσουν το κάπνισμα. Έτσι δείχνουν οι στατιστικέ. Και η ιδέα ότι κάτι είναι λιγότερο επιβλαβέ από κάτι άλλο και άρα θα πρέπει να ενθαρρύνεται, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν νομίζω ότι εδώ θα, θα κανένα κανένας ε, να χρησιμοποιεί λιγότερο ασφαλή λάστιχα από περισσότερο ασφαλή μόνο και μόνο επειδή είναι λιγότερο ασφαλή. Πιστεύω ότι το κάθε κράτο μέρο έχει κάποιο περιθώρια λιγμών και κάθε ο άνθρωπος μάλλον έχει δυνατότητα ελευθερίας επιλογής, αλλά δεν πρέπει στην άσκηση των δικών του συνήθειών να συμπαρασύρει και άλλους και να τους εκθέτει σε κίνδυνο. Τα παιδιά δεν έχουν δυνατότητα επιλογής και μετά εξαρτώνται, αποκτούν εθισμό. Είναι όμω αργά πια. Τώρα, παρά τις προσπάθειες, ε, δεν είναι επιδοτήσεις ε, ε, τεράστιο για τον καπνό. Δεν ζητήθηκε άλλωστε να νομιμοποιηθεί η κάναβης. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλός ο καπνός λοιπόν. Και πολλοί μίλησαν για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τη γεωργία και τις επιδοτήσεις. Ναι, θα πρέπει ε, να ρυθμίσουμε την κατάσταση και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να είναι βοήθεια για όσους θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα. Αλλά το καλύτερο είναι να ζητήσει κανείς μια επαγγελματική συμβουλή για να βοηθηθεί. Αυτά και αν ανακαλυφθεί ένα νέο φάρμακο στην Ευρώπη που μπορεί να σώσει 100.000 ε, ζωές το χρόνο, όλοι θα ζητούσαν απαιτητικά να υιοθετηθεί. Έχουμε εδώ μια πρωτοβουλία που μπορεί 700.000 ζωές το χρόνο. Αυτό δεν σας λέει τίποτα. Επαναλαμβάνω, αφισβήτα, αν ε, ανακάλυπτα με ένα φάρμακο που θα έσωσε 100.000 φορές το χρόνο, αμέσως θα το νομοποιούσαμε. Δεν μπορείτε να ε, έχετε την επιλογή να, και παρόλα αυτά να θέλετε να γίνετε το παιδί καπνιστή. Σίγουρα ο καθένα θα πρέπει να κάνει τι επιλογέ του, αλλά δεν θα πρέπει να βλάπτει άλλου κατά την άσκηση αυτών των επιλογών, ιδιαίτερα ανηλίκου. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μας βοηθήσει, βοηθήσει να την προωθήσουμε, ώστε να μπορούμε να κοιτάζουμε στο παρελθόν με κάποια περηφάνεια και να λέμε, εάν μη τι άλλο, υιοθετήσαμε μια πρωτοβουλία που με κάθε χρόνο έσωσε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ζωές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Ε, ήταν πολύ εντυπωσιακά αυτά που μας είπατε και απαντητικά στις ερωτήσεις και τελικά το συμπέρασμα και η κεντρική ιδέα ε, είναι αυτό που μας είπατε. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον Επίτροπο να απαντήσει σε ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε εκείνον από πλευρά των συναδέλφων. Παρακαλώ κύριε Μπόρους, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πραγματικά ζωηρή συζήτηση και μου άρεσε με αντικρώμενες απόψεις. Είπαν και κάποιοι ότι η οδηγία δεν πηγαίνει αρκετά μακριά και ορισμένοι θεωρούν ότι το παρακάνουμε. Λοιπόν, και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μάλλον είμαστε στη σωστή οδό. Και όπως είπε και ο Υπουργός, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Προσπαθούμε να προτείνουμε κάτι το οποίο θα έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη συνένεση, παρά να προχωρήσουμε με υπερβολική ταχύτητα ή με υπερβολική βραδίτιδα και να διαφωνήσουν οι πάντες. Έχω πάει και σε άλλο συμβούλιο ανταγωνιστικότητας Έχω έρθει στην Επιτροπή Γεωργίας ε, που με ρώτησαν και για το κάπνισμα και την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Ήρθα εδώ σήμερα, έχω συναντηθεί με βουλευτές, ευρωβουλευτές, ξέρω τις διάφορες απόψεις. Ε, προσοχή όμως ε, με διάφορα επιχειρήματα. Για παράδειγμα, εάν υπεριθμίσουμε λέγουν τον καπνό και τα προϊόντα του, αυτό θα έχει δημοσιονομικές συνέπειες για τα έσοδα των κρατών. Άρα Δηλαδή τι, να προωθήσουμε το καπνό για να γεμίσουν ε, τα κρατικά ταμεία. Ή... Άλλοι λέγουν ότι αν ρυθμίσουμε αυτά τα προϊόντα καπνού και επιτύχουμε μάλιστα και μειωθεί ο αριθμός των καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη πενταετία, ο στόχος μας είναι να μειωθεί κατά 1,2 εκατομμύρια, αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας. Άρα να προωθούμε, να διαφημίζουμε τον καπνό, να αυξηθούν οι καπνιστές και να μην έχουμε πρόβλημα ανεργίας. Και μάλιστα αύξηση θέση ανεργασία. Προσοχή σε αυτά τα επιχειρήματα, διότι προβάλλονται καμιά φορά με σθένος και με ζέση και σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι και πάρα πολύ ελκυστικά επιχειρήματα. Εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα. Υποθέτω ότι η απάντηση είναι καταφατική. Πράγμα που εξηγεί ε, γιατί σε αυτό το κείμενο το κοινοβουλευτικό έχουμε το σήμα απαγορεύεται το κάπνισμα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε χρέος ε, να μην προωθούμε το κάπνισμα και να το κάνουμε όσο γίνεται λιγότερο ελκυστικό. Βέβαια μπορεί να διαφωνούμε ως προς τα μέσα που θα ακολουθήσουμε για το στόχο μας, αλλά ο στόχος είναι σαφέστατος, έτσι δεν είναι. Θα το γυρίσω στα Ιταλικά τώρα για να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που έκαναν ορισμένοι Ιταλοί συνάδελφοι. Αυτό το θέμα της ελευθερίας επιλογής, τι κάνουμε δηλαδή εδώ. Γίνεται μια συζήτηση γενικότερη ε, για διάφορα σημεία, ας πούμε αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναγραφή ε, σε κάποια ε, πακέτα ή να έχουμε ειδικέ τιμές ε, όπως έχουμε κοινέ τιμές για το ενόπνευμα για τους οδηγούς. Αν κάποιος έχει ένα τροχαίο δυστύχημα να τον αφήσουμε να αποφασίζει ελεύθερα αν θα σκοτωθεί όχι. Στην ε, οδική ε, ασφάλεια έχουμε κάποιες ρυθμίσεις για να προστατεύουμε γενικότερα ε, τον πληθυσμό. Ας πούμε υπάρχουν δύο τάξεις για τα κράνη των μοτοσυκλητιστών. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα και σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν κανόνες, διότι τελικά τα θύματα των τροχαίων τα πληρώνει το κοινωνικό σύνολο, οι πολίτες. Δεν έχουμε πει ότι απαγορεύεται γενικά το κάπνισμα για όλους. Δεν είναι ε, όπως υπό το απαγόρευση, αν θυμάστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τότε είχε αλλάξει το Σύνταγμα και απαγορεύθηκε στι Ηνωμένε Πολιτείε συνολικά η παραγωγή και πώληση εινοπνεύματος. Δεν λέμε εμεί αυτό το πράγμα, λέμε ότι ε, επιτρέπεται το κάπνισμα ελεύθερα, αλλά να είναι λιγότερο ελκυστικό, να μην προσελκύονται νέοι καπνιστές. Αυτό είναι θεμητό. Και τελικά ε, και το ε, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει λάβει αντίστοιχε αποφάσεις. Η ελευθερία επιλογής παραμένει. Ο καθένας μπορεί να αποφασίζει ελεύθερα αν θέλει να καπνίζει ή όχι. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να εθαρρύνουμε τους νέους να αρχίζουν να καπνίζουν. Είναι σημαντικό να εγκρίνουμε εμείς Εμεί δεν είμαστε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί δικαίωμα πρωτοβουλία έχουμε, αλλά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνουν κατά τη διάρκεια της παρούς ε, κοινοβουλευτική θητεία. διότι σε αντίθετη περίπτωση <coughs> μετά θα πρέπει να εκλεγεί νέο κοινοβούλιο, να ορίσει νέους εισηγητές, να αρχίσει από την αρχή η συζήτηση και θα παραταθεί η όλη προσπάθεια. Λοιπόν, ακόμα και αν ε, εγκρίνουμε κατά την παρούσα θητεία όλα αυτά τα πακέτα που σας έδειξα θα αντικατασταθούν το νωρίτερο σε 3,5 χρόνια, ίσως και 4. Λοιπόν, αν συνεχίσουμε αυτές τις χρονοτριβές και τις καθυστερήσεις, αφού τόσα χρόνια επιμένει το Κοινοβούλιο να αναθεωρηθεί η οδηγία για τα προϊόντα καπνού, τι σημαίνει αυτό. Ότι θα πλουτίσει ακόμα περισσότερο η καπνοβιομηχανία. Βέβαια μπορεί κάποιο να έρθει να σας πει εδώ ή εκτός κοινοβουλίου ότι η οδηγία αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα ε, στην κατανάλωση προϊόντων καπνού. Αν ισχύει αυτό, ε, τότε γιατί να ανησυχούμε πώς καθούν θέσεις εργασίας ή χρήματα από τα κρατικά ταμεία. Αυτά τα επιχειρήματα προβάλλονται διότι πραγματικά θα κάνει τη διαφορά αυτή η οδηγία. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Και ακριβώς επειδή θα αλλάξουν τα πράγματα, προβάλλονται αυτά τα επιχειρήματα για τις οικονομικές συνέπειες, τη ε, της μείωσης της κατανάλωσης προϊόντων ε, καπνού και της μείωσης των καπνιστών. Και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Έτσι ένα ακόμα επιχείρημα στη συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι γεγονός ότι αν μειωθεί ο αριθμός των καπνιστών θα υπάρξουν οικονομικές συνέπειες, αλλά δεν θα είναι όλες αρνητικές. Ορισμένες μπορεί να είναι ακόμα πιο θετικές και περισσότερες από τις αρνητικές, διότι αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τα κρατη θα εξοικονομήσουν χρήματα από τα δημόσια ταμεία, από τα ταμεία υγείας ας πούμε, αλλά και αυτοί που θα σταματήσουν το καπνισμά θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά αλλού σε άλλου κλάδου τη οικονομία που δεν θα τα δίνουν πια για τσιγάρα και θα δημιουργηθούν αλλού θέσεις εργασία. Δεν θέλω να σα κουράσω με στατιστικέ. Ο Υπουργό, πολύ ωραία εξήγησε ότι ε, το εισόδημα ε, του συνόλου της καπνοβιομηχανίας που είναι 20 δις είναι πολύ λιγότερο από αυτό που δαπανούν τα κράτη και επενδύουν ε, για την θεραπεία των ασθενειών που προκύπτουν από το κάπνισμα και ε, των ε, απολειών στην οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι όταν κάτι το απαγορεύεις είναι πιο γλυκό και πιο ε, ελκυστικό. Είναι γεγονό αυτό. Μερικά από τα καλύτερα πράγματα στη ζωή είναι απαγορευμένα. Αλλά το να λε ότι θα αυξηθεί το λαθρεμπόριο και η τσιγάρα μαϊμού είναι λάθο επιχείρημα. Διότι για πρώτη φορά ε, με τρόπο μάλιστα δεσμευτικό βάζουμε και ένα στοιχείο ασφαλείας, ένα χαρακτηριστικό και ένα χαρακτηριστικό ανείχνευσης στα προϊόντα καπνού. Για πρώτη φορά θα επιβληθεί αυτό δια νόμου. Όχι για να προστατευθούν τα κρατικά ταμεία, αλλά κυρίως για να μην επιτρέπουμε σε άλλα προϊόντα καπνού που δεν συμμορφώνονται με την κοινωτική νομοθεσία να ε, εισάγονται στην αγορά μας. Βέβαια, όσοι εξάγουν τσιγάρα και τέτοια προϊόντα ε, εκτός ένωσης δεν δεσμεύονται αυτούς τους κανόνες. Ε, αυτά ισχύουν μόνο για όσα τσιγάρα και προϊόντα καπνού κυκλοφορούν εντός της ενώσεως. Τώρα, τα αρώματα και οι γεύσεις. Ε, ναι, είναι γεγονός ότι και οι ουσίες αυτές και ο τρόπος με τον οποίο τα τσιγάρα τα ίδια παράγονται και εμφανίζονται ως προϊόντα καπνού επηρεάζουν τις αποφάσεις που παίρνουν κυρίως οι νέοι όταν αποφασίζουν να μπουν στο κάπνισμα. Γι' αυτό λοιπόν και το ρυθμίζουμε. Τι θα πρέπει τώρα να απαγορεύσουμε όλες τις προσθετικές ουσίες, όλες τις γεύσεις. Ο κανόνας της αναλογικότητας μας λέγει ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε τα, τις χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα. Υπάρχει ορισμός αντίστοιχα στην οδηγία. Σε ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων που θα επιτηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη θα αποφασίζεται τι εστί χαρακτηριστική γεύση ή άρωμα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα αυξηθούν ούτε οι απομιμήσεις ούτε το λαθρεμπόριο. Ε, γιατί έχουμε αυτά τα στοιχεία, τα νέα που επιβάλλουμε. Για το ηλεκτρονικό τσιγάρο τώρα. Είναι σαφής ο κανόνας. Πρώτον, δεν θα πρέπει να προωθείτε, γιατί αν και ακόμα και ορισμένοι θεωρούν ότι είναι λιγότερο βλαβερά, δημιουργούν μια εσφαλμένη αίσθηση ασφαλείας. Ορισμένοι που καπνίζουν αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θεωρούν ότι σταμάτησαν να καπνίζουν γιατί δεν βγαίνει καπνός. Ε, παρόλα αυτά ε, προκαλούν την ίδια βλάβη ε, στον εαυτό τους, δίνουν αυτή την εσφαλμένα αυλαβή αίσθηση και εγώ ε, θεωρώ ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα προκαλούν εξίσου εθισμό και οδηγούν σε κατανάλωση νοικοτήνης και επίσης μπαίνουν στην ίδια κατηγορία. Είναι προϊόν καπνού. Κάτω από ένα κατόφλι ή πέρα από ένα κατόφλι που ήδη υπάρχει σε άλλα προϊόντα καπνού χρειάζεται έγκριση το προϊόν και χαίρομαι για τα σχόλια που έκανε ο αξιότιμος κύριος Τζανόνι και ο Πέτερ Λίζε για αυτό το θέμα του παθητικού καπνίσματος. Νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόνοια, αλλά να το ξανακοιτάξουμε ε, για το πώς θα βοθαρίνουμε το παθητικό καπνίσμα. Στις εικόνες, στις προειδοποιητικές ή και στο κείμενο το προειδοποιητικό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το παθητικό κάπνισμα για το σνούς. Ξέρω απ' και ανακατοτά όλα τα επιχειρήματα υπέρ του καπνού αυτού. Ακόμα και στο έντυπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρχε ειδική ε, για την άρση της απαγόρευσης. Εγώ δεν θα προβάλλω μόνο τα νομικίστικα ε, επιχειρήματα που είναι και από μόνα τους πάρα πολύ ισχυρά όταν σου δίνω κάτι με αντάλλαγμα κάτι άλλο, δεν μπορείς να καταργήσεις το ένα και να κρατήσεις το αντάλλαγμα. Η απαγόρευση του σνούς υπήρχε πριν ενταχθεί στην Ένωση η Σουηδία. Δηλαδή τεχνικά όταν προσχώρησε θα έπρεπε να είχε απαγορεύσει και στο εσωτερικό της χώρας την κυκλοφορία. Αλλά για πολιτικούς λόγους έγινε αυτή η παραχώρηση υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σνούς. Και να απαγορεύονται οι χαρακτηριστικές ε, αρωματικές ουσίες και γεύσεις, ε, αυτό θα περιορίζει μόνο στο 10% του σνούς. Γιατί τόσο είναι το ποσοστό. Και από εκεί και πέρα, ποιους μπορούμε να απαγορεύσουμε αυτές τις ουσίες, τις γεύσεις, τις χαρακτηριστικές και τα αρώματα για καπνό ε, που ε, χρησιμοποιείται όχι από τη μύτη αλλά στη μάσηση και να επιτρέψουμε για το σνούς. Ε, αυτά είναι ζητήματα που θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι γιατί θεωρώ ότι η πρόταση είναι και ισόρροπη και λογική. Δεν οδηγεί σε ένα κράτος νταντά, ούτε θέλουμε να νταντεύουμε τον κόσμο με τρόπο έτσι φόντα ε, Είναι ε, ισορροπημένη προσέγγιση, ούτε το παρακάνουμε. Πηγαίνουμε όσο χρειάζεται για να φτάσουμε σε ένα στόχο που σας ανέφερα και στην αρχή ε, της μείωση του αριθμού των καπνιστών στην Ένωση την επόμενη πενταετία κατά 2%. Thank you very Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρότα. Ευχαριστούμε για τόσα μας είπατε. Για την δευτερολογία σας όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σαφή, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση και τώρα θα πάμε στο δεύτερο πάνελ που έχουμε. Κύριε Μπετλέτη. Και εκτό από την κυρία Μπρετελέτη, η οποία ασχολείται με αυτή την εταιρική σχέση κατά του καπνίσματο, έχουμε τον κύριο ε, Ρέλινγκ, ο οποίο ε, προέρχεται από την ε, Συνομοσπονδία των Καπνοβιομηχανιών. Κύριε Μπρετελέτη, πρώτη. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Καλησπέρα σα, αγαπητοί ευρωβουλευτέ. Σήμερα δεν πρόκειται να κάνω μια εισήγηση της, του, του φορέα μα και του φορεί με οποίου συνεργαζόμαστε κατά του καπνίσματο. Όμω αυτό που θέλω είναι να σα πω ότι Εκπροσωπούμε και χιλιάδε ε, νοσηλευτριών, νοσηλευτών, γιατρών και ασθενών οι οποίοι πέρασαν πάρα πολλά οδυνηρά και πόδινα χρόνια ε, οι οποίοι προχωρούνται από αναπνευστικέ ασθένειε, καρκίνο, ε, καρδιολογικέ παθήσει. Και το πρώτο που θέλω να σα πω είναι κάτι το οποίο αφορά την πρώτη ευρωπαϊκή τροπή. Είναι εξισορροπημένη, είναι αξιόλογη και ιδιαίτερω μα χαροποιεί το ότι τα κράτη-μέλη έχουν τώρα την ευκαιρία να έχουν αυτή, αυτή τη συσκευασία χωρί ενδείξει και παραστάσεις και αυτό να γίνει σύμφωνα με την πρόταση υποχρεωτικό. Δεύτερον, πριν δούμε ακριβώ τι επιπτώσει στην οικονομία, κάτι το οποίο έχει φέρει επιχειρήματα για τον δύο αντιμαχωμένων πλευρών, πρώτα-πρώτα. Ε, αυτό να δούμε, να δούμε μισό και να αναλογιστούμε τι γεγονότα και ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο που οδήγησαν ε, τα τελευταία 45 χρόνια στην ε, νομοθεσία κατά του καπνίσματος και στην αναθεώρηση αυτής. Είχαμε μέσα αυτή την απόφαση της κυβέρνησης της για την συσκευασία. Να σας πω μια ιστορία. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ αυτό και σύγκριση με την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιαδιώτη αποφάσισαν οι, οι καπνοβιομηχανίες να αντεπιτεθούν από την Ουρουάη στην Αυστραλία μέχρι την Νορβηγία. Ο, ο Γολιάθ φαινόμενο της δικαιοσύνης, χώρες που προέβησαν σε απαγορεύσεις για να σώσουν τους νέους από το κάρνισμα. Και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Γολιάθ επιτέθηκε διότι προσπάθησε να να, να φημώσει την δημόσια διαβούλευση η οποία ανερχόταν σε 85.000 ε, ε, συμβολές και τελικά πώς έβγαιναν στα δικαστήρια κατά τον κύριο Ντάλη. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Απλώς θα σας πω τα εξή. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κοινοβιομηχανία επιτέθηκε στον υπεύθυνο για την υγεία της Επιτροπής. Βεβαίως θα δικαιωθεί, θα αναδειχθεί του και σήμερα, τη μέρα αυτή της, ε, α, ε, ακρόασης, θα δώσουμε το λόγο και την σκητάλη στους ευρωγνώμονες που μετά το λόγο, γιατί το βασικό όπλο αυτού του Γολιάθ είναι τα ψέματα και κάποιοι μύθοι για να δημιουργήσουν φόβο και αμφιβολίες στο μυαλό μας. Για να δούμε συγκεκριμένα τι επικαλούνται. Πρώτος μύθος δεν έχει ακουστεί η φωνή τους. Είμαστε σαφείς κυρίε και κύριοι. Ο βασικός που το επικαλούνται αυτό ποιος είναι. Δεν τους αρέσει το περιεχόμενο της πρότασης. Δεύτερον, παρά τους ισχυρισμού τους, κανείς δεν λέει ότι θα πρέπει να μην ληφθεί υπόψη η καπνοβιομηχανία. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει ένα τοπίο διαφάνεια και ίσους όρους. Όταν ήρθε η ώρα της συνάντησης επίσης, η προσβασιμότητα σε κάποια έγγραφα έχει καταδείξει ότι είχε πρόσβαση στο γραφείο του Επιτρόπου, την οδηγία για τα προϊόντα καπνού α, τα έχει, την οδηγία την έχει δει, έχει συμβάλει στην ε, δημιουργία της και επομένως όπου και που δεν έχουν προσβασιμότητα. Και ο Τόμα Τζέφερσον τι έλεγε, δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο παρά η ίση μεταχείριση των όσων δεν είναι ίση. Άλλος μύθος, ότι η οδηγία και τα μέτρα της πρόκειται να δημιουργήσουν ένα παράλληλο παράνομο εμπόριο και λαθρεμπόριο. Τι γίνεται, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για το ότι οι κρατοβιομηχανίες για δικό του συμφέρον έχουν ε, δημιουργήσει τέτοιες, τέτοιες παράνομη διακίνηση. Και τώρα έχουν ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αυτό. δεύτερο, αυτό το παράνομο εμπόριο, τι είναι, δεν, δεν μας δίνουν ορισμό, τι εννοούν. Να σας πω. Έχουμε λαθρεμπόριο, απομίμηση, ε, και άλλες μορφές. Επομένως, γιατί μας λένε ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Τρίτος μύθος. Δεν προσάγουν τίποτε στοιχεία. Θα σας τα εξηγήσουν καλύτερα οι μυρογνώμονες. Το ότι ισχύει δεν ισχύει εδώ απλώς. Πρέπει να δούμε ότι έχουμε 1096 σελίδες στοιχείων που κατατείνουν στα όσα προτείνει η οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Άρα, ποιο είναι το ζούμε ποια είναι η ουσία. Ότι δεν είναι ειδική της καπνοβιομηχανίας στο ε, αυτό θα τον αποδείξω. Άλλος μύθος. Ότι αυτοί οι πρόταση πρόκειται να παραβλέψουν την οικονομία. Όπως είπατε κύριε Μπόλ, δεν είναι λογικό αυτό. Ή θα πρέπει να πούνε ότι τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και θα παραβλάψουν την οικονομία ή να πούν δεν είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα. Οπότε αφού δεν είναι αποτελεσματικά, πώ θα βλάψουν την οικονομία στα γαλλικά τώρα. Να, είναι το φίδι που τρώει την ουρά του. Κάνει πραγματικότητα τώρα. Το κάπνισμα είναι εθιστικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κόψει κανείς. Το πιο σωστό είναι να μην αρχίσει κανείς να καπνίζει και ξέρουμε ότι το 75% των καπνιστών αρχίζουν πριν τα 18 και 94% πριν τα 25. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 80 εκατομμύρια ανηλίκους, 80 εκατομμύρια νέους και οι κόρη μου βρίσκεται εδώ στην αίθουσα, ξεκινούν ε, μπορεί να ξεκινήσουν τώρα και είναι 15 ετών. Και εγώ δεν θέλω να ξεκινήσει το κάμισμα να Τώρα ποιο είναι το κόστος; Από ό,τι μα είπαν, το κάμισμα οφείλεται για 700 θανάτους, δηλαδή 200 την ημέρα, 8 ε, και ένας να περιμένει κάθε δευτερόλεπτο. Επομένω έχουμε 9,94, 517 δις που είναι ζημία, 5,3 όσον αφορά το κόστος στην παραγωγή και 9,94 εκατομμύρια όσον αφορά τα χρόνια ε, των ζώων που χάθηκαν. Τώρα για να δούμε πάλι την αφιόρεση της οδηγίας σε σύγκριση με την μάχη. Δηλαδή όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν πάρα πολύ ισχυρά λόμπι οι κοινοβιομηχανίες. Ξέρετε όμως πόσο ισχυρή είναι στην πραγματικότητα, γιατί το 2010 τα συνδυασμένα κέρδη των 6 κορυφαίων κοινοβιομηχανών ήταν 35 δις δολάρια. Αυτό αντιστοιχεί στο κέρδη της Coca-Cola, της Microsoft και της McDonald's ορευτικά. Και σύμφωνα με κάποιο μητρό διαφάνειας, 97 λομπίστες δρούν εδώ στις Βρυξέλλες για τις και έχουν προβολούν 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Εμείς στο φορέα μας έχουμε μόνο δύο άτομα προσωπικό και στις Βρυξέλλες ε, ε, ασχολούνται τόσο λίγοι όσο τα δάχτυλα ενό χεριού. Και τελικά, ποιο είναι το μήνυμα. Θα πρέπει από την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ να αντιληφθούν τα εξή συμπεράσματα. Πρώτα πρώτα ο Δαβίδ δεν φοβόταν όλοι οι άλλοι φοβόντουσαν γιατί ήξερε ότι θα πολεμήσει αυτόν τον γίγαντα και ελπίζω ότι και εσεί ακριβώ το ίδιο θα σκεφτείτε. Οι Ευρωπαίοι σε εσάς υπολογίζουν. Εσείς να τους προστατεύσετε από τα συμφέροντα των εταιριών. Επίσης, γιατί νίκησε ο Δαβίδ, γιατί είχε πίστη ότι θα νικήσει. Εσείς έχετε το μέρος σας, τον κόσμο. Αυτή η αναθεώρηση του νομοθετήματος είναι μια διαδικασία πάρα πολύ διφορούμενη, επίμαχη, υποφασιστική και έχει σημασία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης γνωρίζουμε τι γίνεται σε εποχές κρίσης και λιτότητας. Είναι μεγάλος πειρασμός μια κυβέρνηση να μην λάβει υπόψη το δημόσιο συμφέρον, αλλά να δώσει σημασία στην οικονομία. Στα οικονομικά μέτρα όμω θα πρέπει μια τέτοια νομοθεσία να, είναι στο επίκεντρο της ε, ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκή οικονομία γιατί έτσι θα ωφεληθούμε και την παραγωγικότητα των Ευρωπαίων, αλλά θα προστατεύσουμε και τους νέους Ευρωπαίους. Πριν δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του, τον, τον Γολιάθ, θα σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και τελειώνω με ένα ερώτημα. Ό,τι και αν σας πούνε τώρα οι οικονομικοί τους πιστεύετε. Mm. Κύριε Γολιάθ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπερτελέτη, αλλά προς το παρόν ακόμα εγώ δίνω το λόγο και ορίζω ποιος ομιλεί. Οπότε, να προετοιμαστείτε, ε, βάλτε και τα ακουστικά σας και όταν είστε έτοιμος ε, μπορείτε να πάρετε και το λόγο κύριε Ρέρινγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, Επίτροπε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι εξ ονόματος της ΚΕΚΕΜ που είναι η ε, Συνομοσπονδία ε, των ε, Κατασκευαστών Σιγαρέτων. Θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω τις θέσεις μας. Λέγομαι Μίχιλ Ρέρινγκ, είναι δύσκολο το όνομά μου, πάντως Γολιάθ δεν λέγομαι. Το τσιγάρο συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε μία ρύθμιση αναλογική δεν θέλουμε τα παιδιά να καπνίζουν, ισορροπημένοι και αποτελεσματικά μέτρα υποστηρίζουμε για να ε, προληφθεί το κάπνισμα στους ανηλίκους. Έχω τρία παιδιά και τον έναν τον έναν και Δαβίδ κατά τύχη και υποστηρίζω πολύ αυτή την πρόταση. Η ΚΕΚΕΜ και τα μέλη της έχουν συμβάλει με περιστατωμένες μελέτες ε, εμπειρογνωμόνων στις 2.000 και πλέον ε, ε, ανταλλαγές απόψεων. Μετά δημοσίευση της πρότασης έχουμε στείλει και νέα σχόλια για διαβούλευση τον Ιανουάριο στην Ιρλανδική Προεδρία στο Υπουργείο Υγείας και σας καλώ αν δεν έχετε ήδη διαβάσει να διαβάσετε τα μέτρα μας και να τα μελετήσετε. Ωστόσο είναι χαμένη ευκαιρία κατά την άποψή μας που έχει προσκληθεί μόνο η ΚΕΚΕΜ, δηλαδή εκπρόσωποι και άλλων κλάδων ε, προϊόντων καπνού και συναφών δεν έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν μαζί σας τις απόψεις τους. Σήμερα θα ε, ασχοληθώ με τους στόχους της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς θα φτάσουμε σε αυτούς, ε, τις ακούσιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τα νομικά ζητήματα και τέλος θα μιλήσω για την ανάγκη διαλόγου και συμμετοχής όσο και διαφάνειας. Όπως σας είπα, εμείς υποστηρίζουμε μία ε, κατάλληλη ανάλογη ρύθμιση βάση στοιχείων. Η πρόταση αυτή όμως αλλιώς δεν θα φτάσει στους δεδηλωμένους στόχους, θα έχει ακούσεις ε, ε, απρόβλεπτες συνέπειες και επιβάρηση και μεγαλύτερο κόστος. Γι' αυτό ανησυχούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το μέγεθος των προειδοποιήσεων στα πακέτα. Δεν έχει επικαλυστεί στοιχεία αξιόπιστα ότι αυτό μειώνει τον αριθμό των καπνιστών ή προλαμβάνει ε, και σταματά, αποτρέπει τα παιδιά από το να αρχίσουν να καπνίζουν. Το ε, ανώτατο ε, εφετείο στις Ηνωμένε Πολιτείε. έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει ούτε ίχνος απόδειξης ότι αυτό συμβάλλει Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να δείχνουν ότι οι γραφικές παραστάσεις, οι οπτικές εικόνες ε, ε, οδηγούν σε μείωση του πνίσματος. Το ίδιο ισχύει και με τη μελέτη σκοπιμότητας που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φαίνεται και να ε, βασίζεται σε αυτή. Σήμερα οι καταναλωτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους κινδύνους που συνδέονται με το κάπνισμα. Το να τους δώσουμε περισσότερες πληροφορίες δεν θα σημαίνει ότι θα αλλάξουν την καπνιστική τους συμπεριφορά και πάλι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της για να ε, απαγορευτούν τα ε, σιγάρα ε, μενθόλης και τα λεγόμενα slim, τα λεπτά. Η πρόταση διατηρεί την απαγόρευση για τους ειδικό νους εκτός της Σουηδίας και ιδιαίτερα βάζει στα φάρμακα κατά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα η πρόταση δεν βελτιώνει την εσωτερική αγορά, ούτε να αρμονίζει, ούτε έρει συγγνώμη, εμπόδια. Αντίθετα, απαγορεύει ολόκληρε κατηγορίε προϊόντων χωρί να βελτιώνει τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Επιβάλλει περιορισμού στο σχέδιο και ε, μειώνει σημαντικά τη δυνατότητά μας να καινοτομούμε και να ανταγωνιζόμαστε. Αυτό βελτιώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το αντίθετο. Ε, στερεί από τους καταναλωτές τη δυνατότητα ε, επιλογής. Δεν είναι ε, ανάλογη. Και μεγάλα μέτρα προστασίας που έχουν μεγάλο κόστος και για μεγάλες αλλά και για μικρές εταιρείες. Και τέλος, δεν αφήνει τα κράτη-μέλη να λάβουν εθνικά μέτρα για τομεί που καλύπτει η οδηγία και τομεί που δεν καλύπτει. Και περαιτέρω έτσι υπονομεύει οποιαδήποτε υποτιθέμενη εναρμόνιση. Οπότε, ε, αντί να καταργεί φραγμούς και εμπόδια στο εμπόριο, η πρόταση εισάγει νέα και θα έχει σημαντικές ανετικές επιπτώσεις. Οι καπνιστές που θα δουν τα προϊόντα του, να απαγορεύονται από τη μια μέρα στην άλλη, είτε θα αλλάξουν προϊόν, είτε θα πάνε στην παρανομή προμήθεια. Και αυτό θα ε, είναι μεγάλο όφελος για τους λαθρεμπόρους και τους ε, όσους παράγουν λαθρέα τσιγάρα. Γιατί εισάγεται αυτή η πρόταση. Μόλις εγκρίθηκε ένα πρωτόκολλο στη συμφωνία, σύμβαση μάλλον πλαίσιο για το λαθρεμπόριο. Επίσης, σημαντικός αριθμός καπνιστών τσιγάρων μεθόλης ε, ε, και slim είναι στην περιφέρεια, στη Φιλανδία, στην ε, Βουλγαρία και σε άλλες περιφερειακές χώρες κοντά στα σύνορα. Και πάλι δεν έχει γίνει ε, μελέτη. Η ε, απαγόρευση της καινοτομίας και περιορισμοί για το πώς θα έχει το πακέτο ε, μας δένει τα χέρια για την πρόθεση των προϊόντων μας και θα είμαστε σε ανταγωνισμό για τα προϊόντα premium και μπορεί να προωθούνται προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας ε, που έχουν και χαμηλότερα εισοδήματα και για τις κυβερνήσεις και για τους λιανοπολιτές και για ε, τις κατασκευάστρες εταιρείε. και αυτό μας κάνει να ανησυχούμε. Όπως σας εξήγησα δεν βελτιώνει η πρόταση λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά εισάγει εμπόδια αντί να καταργεί. Ε, βάζει νέους καθόνες νομική μάλλον ε, καταπολεμά τη βάση της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Και τα ε, στοιχεία που έχει δεν συνάδουν με τις νομικές ε, υποχρεώσεις και μεταξύ αυτών η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του εμπορίου και τελικά η προστασία της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ΠΟΕ και, τη Συμφωνία Τρίψη για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας. Έρχομαι τώρα σε κάποιους ισχυρισμούς που λέγουν ότι η δική μου βιομηχανία, ο κλάδος που εκπροσωπώ, δεν είναι νόμιμος και θεμητός συνομιλητής. Μα ε, συνθήκες ε, ορίζουν ε, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ενδιαφερομένων. Και θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα συμφέροντα. Εμείς εφαρμόζουμε και συμμορφούμαστε προς τους κανόνες και τους κανόνες για τη διαφάνεια και τον κώδικα συμπεριφοράς και δεντρολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα λόμπι. Αλλά πιστεύουμε ότι όλοι οι ενεχόμενοι θα πρέπει να λέγουν τη γνώμη τους για να ακούγονται και να εισακούγονται. Και ως εκπρόσωπο σήμερα της ΚΕΚΕΜ εκπροσωπώ μόνο τις εταιρείε που είναι μέλη μας. Και σας καλούμε να ακούσετε επίσης ε, κάποια στιγμή εν ευθέτω χρόνο τη φωνή των εκπροσώπων των 1,5 εκατομμύριων ε, εργαζομένων που ε, εξαρτώνται εν μέρη πλήρως για το εισόδημά τους από τα προϊόντα καπνού. Θα ήθελα να σας καλέσω τέλος να διαβάσετε σύντομα την διαφάνεια που βλέπετε. Και πάλι να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να συμμετέχουμε σήμερα. Ακούτε σήμερα την ΚΕΚΕΜ και στο μέλλον παρακαλώ τους εκπροσώπους όλων των κλάδων που συνδέονται με τον καπνό γιατί είναι κρίσιμο αυτό και τεράστια σημασία. Εμείς υποστηρίζουμε μία ρύθμιση αναλογική κατάλληλη και βασιζόμενη σε στοιχεία. Η παρούσα πρόταση δεν ανταποκρίνεται σε αυτό. Σας είπα προηγουμένως ότι οι εταιρείε μέλη της ΚΕΚΕΜ προτείνουν λιγότερο περιοριστικά μέτρα, πιο στοχευμένα και ε, αναλογικές εναλλακτικέ λύσεις. Παράδειγμα, μέτρα που πραγματικά θα αποτρέπουν τα παιδιά από την αγορά προϊόντων καπνού. Ε, προϊόντα ε, με μεγάλη αποτελεσματικότητα και είμαι πρόθυμος να συμμετέχω σε επότερο στάδιο. Έχουμε προτείνει 20 μέτρα. Αν έχετε ερωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα ή για τα μέτρα αυτά, ε, με ε, χαρά να σας απαντήσω στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Η κυρία Ρης, δεν βλέπω άλλους. Η κυρία Ρης, παρακαλώ, είστε η μόνη που θέλετε να ρωτήσετε. Okay. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς τον κύριο Ρέρινγκ. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό μαζί του, γιατί εξέφρασε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά ε, το μέγεθος των ε, προειδοποιήσεων ε, που περιλαμβάνονται στα πακέτα. Γι' αυτό και, μίλησα ότι, γι αυτό και είπα προηγουμένως ότι είναι αναγκαίο να οργανώσουμε και ενημερωτικέ εκστρατείε μεγάλη ευέλεια, όπω γίνεται σε άλλε χώρε, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και ούτω καθεξή. Σε ό,τι αφορά τα slim λεπτά σιγαρέτα μενθόλη, έχουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, το πιο δολοφονικό στι περισσότερε χώρε. Γαλλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο. Α, συγγνώμη, διορθώνει η ομιλήτρια. Ε, ο καρκίνο του πνεύμονα είναι πολύ πιο θανατηφόρο πια από τον καρκίνο του μαστού. Δεν ξέρω σε τι έρευνε αναφέρεστε κύριε Ρέρινγκ. Φαίνεται ότι έχουμε διαφορετικέ πηγέ πληροφόρηση. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που μας απασχολούν εδώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να, να, να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την απεξάρτηση, αλλά θα πρέπει η ρύθμιση να ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το κατόφλι. Δεν ξέρω ποιο είναι το κατάλληλο κατόφλι. Ε, είναι μέτρο που πρέπει να βοηθά στην ε, ε, απεξάρτηση. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το σωστό κατόφλι, η σωστή τιμή. Πάντως, δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος της καπνοβιομηχανίας και για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, φαίνεται ότι γίνονται πολλές αγοραπολισίες και μετατοπίσεις. Τι δεν μας βεβαιώνει ότι σε λίγα χρόνια το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα γίνει και αυτό διασκεδαστικό, ελκυστικό, κομψό, για να ελκύει ακόμη περισσότερους ε, που δεν είναι καν μέσα στο κοινό στόχο. Θα πρέπει να ε, εμείνουμε στην αρχική μας προσέγγιση ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα είναι μέσω απεξάρτηση. Ελίνα Μακάβαν. Ευχαριστώ. σε ό,τι αφορά των καλεσμένων από τη ΣΕΣΕΜ, είπατε ότι οι καπνοβιομηχανίες σας θέλουν να αποτρέψουν τους νέους από το κάπνισμα. Ξέρετε την μελέτη της ΠΟΕ για το κάπνισμα σε 14 χώρες μέλη αυξάνεται το κάπνισμα στα αγόρια. Και μάλιστα σε νέα χώρες, ακόμη και στα 15 χρόνια κορίτσια έχει αυξηθεί η τάση, ακόμη και στη Σουηδία ε, έχει αυξηθεί το κάπνισμα στους νέους. Μιλούμε για παιδιά, ούτε καν ε, για νέους. Πρόκειται για παιδιά στα σχολεία. Σε ό,τι αφορά τις διαφημίσεις ε, της καπνοβιομηχανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας είπαν ότι δεν έχουμε αντίστοιχο στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. ή μήπως έχουμε και μπορείτε να μας το πείτε. Αναφερθήκατε στην ομολογία, του ΔΕ, ή μάλλον στην ομολογία των Ηνωμένων Πολιτειών για το κάπνισμα και την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων. Έχουμε όμως μία έκθεση για την, απαγόρευση, για την ε, πρόληψη από το κάπνισμα στους νέους και το συμπέρασμα της μακροσκελούς μελέτης είναι ότι τα πορίσματα ε, μιλούν για την εσκεμμένη χρήση των ε, προϊόντων καπνού για την προσέλκυση νέων στο κάπνισμα. Ε, θα ήθελα, όπως μας είπε και ο Υπουργό ε, προηγουμένως, να πείτε ε, τέτοιου είδους ελκυστικά πακέτα σε ποιον προκατευθύνονται, ποιον προσπαθούν να ελκύσουν. Λοιπόν, είπαμε ένα λεπτό έχετε, μία ερώτηση, δύο οι υπόλοιποι. Και τώρα η κυρία Άντερσον πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα για το λαθρεμπόριο ή το παράνομο εμπόριο και έχω και εγώ μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της ΕΣΕΜ. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι δικηγόροι να σταματούν οποιαδήποτε ε, επιχείρηση. Ε, και ξέρω κύριε Γολιά, αυτό το όνομά σας. Ε, Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το μύθο Δαβίδ και Γολιάθα του Free Trade ε, Partnership και να σας ρωτήσω ε, σε ό,τι αφορά την ε, υποτιθέμενη ανάμειξη στο λαθρεμπόριο εμπόριο. Υπήρχαν κάποιες συμφωνίες συνεργασίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τεσσάρων μεγαλύτερων παραγωγών σιγαρέτων το 2004 από το 2004 με το 2010 και οι συμφωνίες αυτές ζητούσαν την καταβολή 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφευθεί ή να παταχθεί το λαθρεμπόριο σιγαρέτων ως τμήμα της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αποσύρει τις αγωγές της Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των μεγάλων αυτών εταιριών των βιομηχανιών. Κυρία Ζόμερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δυστυχώς άκουσα μόνο το τέλος της παρουσίασής σας γιατί καθυστέρησα αλλά κατανοώ τα επιχειρήματα. Κάτι άκουσα για τα τσιγάρα με με ε, Ότι αγορεύεται το προϊόν αυτό αν απαγορεύσετε τις γεύσεις και τα αρώματα. Αυτό το θεωρείτε σκόπιμο. Και έτσι θα καταστρέψετε και το καπνό ε, που σνιφάρεται και δεν καπνίζεται, που δεν βλάπτει την υγεία. Και στο τέλος η τυποποίηση των πακέτων και τελικά και των τσιγάρων. Ε, αυτό κλειτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προτείνει. Είναι σε θέση η βιομηχανία αυτό να το αποτρέψει, ε, δηλαδή να μπουν λαθρέα τσιγάρα μαζικά στην αγορά. Όταν δεν είναι τυποποιημένα και είναι γενική εικόνα όλων, ακριβώς τότε είναι πιο εύκολο να μπουν λαθρέα τσιγάρα. Και τέλος, ε, ε, πώς εκτιμάτε το κόστος της ε, ανιχνησιμότητας του συστήματος που θέλετε να θεσπίσετε. Ο κύριος Πιέλνερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εγώ έχω κι άλλο πρόβλημα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θεωρώ ότι ρυθμίζει επαρκώς το εθιστικό και επιβλαβές περιεχόμενο των προϊόντων καπνού. Θα προτιμούσα αυτή ήταν η προσέγγιση και όχι το θέμα της γεύσης. Γιατί ακούστηκε η μεθόλη. Ποιος μπορεί να αποδείξει ότι η γεύση κάνει τη διαφορά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια επιστημονικά τεκμήρια. Πολύ δύσκολο νομίζω θα βρούμε κάτι τέτοιο. Όταν ήμουν νεότερος και προσπάθησα να αρχίσω το κάβρισμα ήταν όχι γιατί είχε ωραία γεύση το τσιγάρο, αλλά γιατί ήμουν ηλίθιος και νόμιζα ότι ήταν μαγιά. Δεν ξέρω αν κανένα δοκίμασε σιγαρέτο με θόλης. Δεν νομίζω ότι το προτιμάνε για την γεύση. Ποια είναι λοιπόν τα επιστημονικά κριτήρια που συνηγορούν ε, πέρα αυτή τη ε, προσέγγιση. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρμς a court judgment. I Όχι, κύριο Σλούτερ, συγγνώμη. Για πες μας, δεν κατάλαβα ακριβώς. Τι λένε οι καπνοβιομηχανοί όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτών των προειδοποιήσεων πάνω στο πακέτο. Πού είναι τα στοιχεία. Έχουμε τη, τη μελέτη του 2003, ε, ένα σώρο 12, ένα σώρο μελέτες. Έχουμε αναλύσει, αποστολή από όλο τον κόσμο και από τη Χάμοντ και όλες αυτές λένε ότι πιάνει, πιάνει η προειδοποίηση πάνω στο πακέτο. Ακόμα και αν είναι 100% αποτελεσματικό, δεν κοστίζει τίποτα. Το κόστος χαμηλό, κάποιο αποτελεσματικό, κάτι, κάτι δίνει σαν αποτέλεσμα. Οπότε, τι γίνεται, το, το, το Αμερικανικό δεν μπορεί να ε, ελέγξει, δεν έχει τους πόρους να κάνει όλων, να τα ελέγξει όλα. Εσείς όμως έχετε τόσο κόσμο, τόσο χρήμα, οπότε εσεί μπορείτε να αναλύσετε και να δείτε πόσο ωφελεί αυτή η υποδοχή. Κυρία Χάρμ, έχω μια ερώτηση για ένα πρόβλημα ε, που απασχολεί πολύ το Κοινοβούλιο και την κοινή γνώμη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω πόσοι από τη δική σας οργάνωση και τους άλλους οργανισμούς της καπνοβιομηχανίας ε, εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο προπολογισμό σας ε, για την περασμένη διετία και για το επόμενο έτος ε, για τις δραστηριότητες λόμπι στις Βρυξέλλες και επίσης γιατί δεν θεωρείται αρκετή μια δημόσια ακρόαση τέτοιου τύπου σημερινή στην Επιτροπή μας για να εκπροσωπείτε και, να ακούγονται τα συμφέροντά σας. Γιατί έχετε στρατιά λόμπι και τεράστιο προπολογισμό για να ασκείτε πίεση. Δεν σας φτάνει μια δημόσια ακρόαση για να προβάλλετε τα αιτήματά σας. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, ε, πρώτα ο Επίτροπος γιατί θα φύγει και την Πέμπτη θα ξανάρθει όμως εδώ για ένα άλλο θέμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο θα πρέπει να πάω στο Συμβούλιο Γεωργίας για να μιλήσουμε αργότερα για το θέμα του αλογίσιου κρέατος. Κοιτάξτε τώρα, για να δούμε. Έχουμε την νομική βάση, ναι, έχουμε το άρθρο 114 και η συνθήκη μας επιβάλλει ω υποχρέωση να μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ ψηλά πρότυπα ε, στην ιστορική πολιτική για τη δημοσιογεία. Πρόκειται το άρθρο 114, το οποίο είναι ξεκάθαρο όσον αφορά την προστασία τη δημοσία υγεία για τι πολιτικέ εσωτερική αγορά. Κατά δεύτερον, αυτέ οι αμερικανικέ αποφάσει είναι αποφάσεις ακριβώς ε, ε, όπως ε, είπε ο κύριο Ζέρι, Και έχουμε και άλλα δικαστήρια, και άλλα εξίσου έγκαιρα. Και περιμένουν η Αμερικανία. Τελικά την απόφαση των δικαστήριων. Όμω, καλά δεν θα είναι και καμία τραγωδία αν το ανώτατο δικαστήριο τον είπα κρίνει άλλος, γιατί έχουμε 13 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία έχουν υιοθετήσει την πολιτική αυτών των ε, προειδοποίησεων πάνω στο πακέτο. Μπορεί να αποφασίσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, ότι παραβιάζεται το Αμερικανικό Σύνταγμα. Αλλά αυτό δεν αφορά τις, ε, τις ευρωπαϊκές χώρες, αφορά τους Αμερικανούς. Θα δούμε τι θα κρίνει το δικαστήριο. Και εκείνε οι χώρε που έχουν αυτέ τι φωτογραφίε προειδοποιητικέ ε, δεν έχουν προσαραγεί αποδείξει ότι σαν αποτέλεσμα αυτών των ε, προειδοποιήσεων και για τον άλλον κανόνων για τα πακέτα ότι έχει αυξηθεί το παρεμπόριο, το, το λαθρεμπόριο κλπ. Και έχουμε άλλωστε και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπου θεωρείται ότι το άρθρο 114 είναι η ορθινομική βάση. Και επίσης ότι μπορούμε να στην ιστορική αγορά να θεσπίζουμε τέτοιου είδου διατάξει Πρόεδρος. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και τα θεσμικά όργανα είχαν ε, τόσο εξέχουσα εκπροσώπηση και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απαντήσατε και στις ερωτήσεις και ε, το εκτιμούμε τα μάλα. Ευχαριστώ πολύ για την έλευση και την παρουσίασή σας. Τώρα όμως σας δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, κυρίες πρώτα, για πέντε λεπτά και ε, παρακαλώ να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας υπευλήθησαν. Νομίζω ότι θα είμαι σύντομη γιατί περισσότερες ερωτήσεις δεν αφορούσαν εμένα. Για αυτές τις φωτογραφίες, κάτι ρώτησε η κυρία Οπότε και εγώ να σας αναφέρω μία μελέτη. Μία, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Η Ουρουάη θέσπισε αυτές τις ε, προδοποίησεις, αυτές τις φωτογραφίες και στις δύο πλευρές του πακέτου. Και όταν το έκαναν αυτό, μειώθηκε η κατανόηση των τσιγάρων από τους νέους κατά 8%. Και για το σύνολο του πληθυσμού η μείωση ήταν της τάξης του 4,3% δηλαδή, περισσότερο από το 2%. που εμείς προσδοκούμε να αποδώσουν, να αποφέρουν τα μέτρα. Άρα είναι αποτελεσματικό μέτρο. Μειώνει την κατανάλωση το κάπνισμα τέλο πάντων και των νέων και του πληθυσμού γενικότερα. Και επίσης η, για την έωσα χώρα, η Αργεντινή, είχε αύξηση του καπνίσματος μια που δεν έλαβε σχετικά μέτρα. Αυτό συμπερασματικά. Και ελπίζω ότι η εμπειρογνώμες στο δεύτερο γύρο θα σας πούμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ, ο Πρόεδρος, και δίνει το λόγο στον κύριο Ρίρινγκ. Σας ευχαριστώ. Ναι, όντως οι περισσότεροι ρωτήσαν προς εμένα και θα προσθέσω να απαντήσω με τη σειρά. κυρία ερώτησε κάτι σχετικά με την έλλειψη στοιχείων παρά τις απαντήσεις που έδωσε εδώ η παρακαθημένη. Γιατί έχουμε μια σειρά χωρών που έχουμε ε, ουσιαστικά που δείχνουν ότι οι προειδοποίησεις αυτές δεν επηρέασαν το κάπνισμα ή τέλο πάντων τίποτα σημαντικό. Και έχουμε για κάποιε άλλε χώρε που λένε ότι λειτουργούν, αποδίδουν αυτές οι, οι προειδοποιήσεις. Αλλά αυτό δεν οδηγεί πάντοτε σε, σε μείωση του καπνίσματος. Δεν γνωρίζω τη μελέτη που πρόκειται από την Ουρουάη ή και την Αργεντινή. Αυτό που είπε ο κ. Μπερτελέτη, αλλά μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι τα δεδομένα από τον Καναδά, τα στοιχεία από τον Καναδά που είχαμε αύξηση και πήγαμε στο 25% 50% για τις προδοποίησεις. Ε, αυτό, αυτή η μελέτη, αυτά τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι μακροπρόθεσμα πρόκειται να μειωθεί ο αριθμός των καπνιστών. Για την ερώτηση της ισχύτρης για το κατά πόσον, έχω υπόψη μου μια πρόσφατη ε, μελέτη του ΠΟΗ. Όχι, δεν γνωρίζω τη μελέτη. Παρακαλώ, αν μπορείτε να μου δώσετε τα στοιχεία από τον ΠΟΗ και να το συζητήσουμε ε, με διαφάνεια ε, ευχαρίστως. Δεν έχω στοιχεία σε σχέση με το συνολικό αριθμό των δαπανών των διαφημιστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, εκπροσωπώ όλες τις εταιρείες πάντως. Μπάσχετος και, και, και τα είχα από τις τρεις εταιρείες που εκπροσωπούμε ε, τα, στοιχεία δεν μπορούσαμε να τα αποκαλύψουμε γιατί είναι εμπιστευτικά. Η κυρία Άντερσον ε, ε, κάτι είπε για το παρεμπόριο, το λαθρεμπόριο και ε, αυτό το οποίο κάνουμε εμεί για να μπορέσουμε τις απομιμήσει να τις σταματήσουμε κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μπορούμε και το κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε <laughs> τέλο πάντων. Και τα σήματα μα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και συνεργαζόμαστε με τι διοικητικέ αρχέ σε πολλέ χώρε, ούτω ώστε να προστατεύσουμε αυτά μας τα διακριτικά, τα σήματα τέλο πάντων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι και άλλα θέματα, αλλά εμείς επειδή έχουμε την κυριότητα αυτών των σημάτων προστατεύσουμε. Άρα, προς αυτήν την κατεύθυνση με νομικά μέσα προσπαθούμε να προστατεύσουμε από τις αντιγραφές παρά τις απομιμήσεις. Τώρα, όσον αφορά το λάθρεμπόριο. εμπόριο όπως τονίστηκε, έχουμε συμφωνίες συνεργασίας. Και τρέψω να επεκταθώ στο εξή. Όταν μιλούμε για το άρθρο 14 της προτάσεως, εκεί είπαμε ότι υπάρχει κάποιο σύστημα ε, ανείχνευσης, παρακολούθησης και αυτό αφορά όμως τα προϊόντα που κατασκευάζουμε ε, όχι παντού, αλλά σε Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το σύστημα αυτό της αναζήτησης επισήμενης παρακολούθησης δεν θα ισχύσει για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δυστυχώς εκεί υπάρχει λάθο. εμπόριο. Το πρωτόκολλο αυτό που είπαμε εγκρίθηκε τον Νοέμβριο και πρόκειται στις χώρες που θα το κυρώσουν να ισχύσει. Ελπίζω, ε, κυρία Σόμα σας κάλυψα όταν είπα για τη συσκευασία, κατά πόσο εκεί οι φωτογραφίες δεν κάνουν τον κόσμο να κόψει το καμισμα. Εμεί πιστεύω θα κάνουμε ότι πρέπει από το χέρι μας, ούτως ώστε να μην αρχίζουν το κάπνισμα. To answer Mr. Γι' αυτό που ερώτησε ο κύριος Σλίτερ θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν θέλουμε να λάβουμε υπόψη κάποιες μέτρες που λένε ε, μεγαλύτερες παραστάσεις, μεγαλύτερες φωτογραφίες, κείμενο για φωτογραφίες και αντιθέτως αν αποφασίσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να επιβάλλουν πρωτοπικές φωτογραφίες υποχρεωτικά αυτό είναι άλλο σημείο. Έχουμε τώρα το 30-40% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των καπνιστών, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τους κινδύνους για την υγεία από το κάπνισμα. Το να αυξήσουμε το μέγεθος των γραμμάτων της προειδοποίησης δεν λέει τίποτα. Και έχει αποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ενημέρωσης όσον αφορά τους κινδύνους από το κάπνισμα. Η κυρία Χάρμψα. Αυτέ οι τρει εταιρείε που εγώ εκπροσωπώ, όσους ε, απασχολούμε ως λομπίστες της Υπάρχει κώδικα διοντολογία ε, για του λομπίστε, υπάρχει αυτό το αρχείο, υπάρχει ένα, ένα ιστότοπο. Τέλο πάντων, εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία. Με σχέση με τα όσα είπε ο κύριο Επίτροπο, έχει δίκιο 100% όσον αφορά την προσχήσασα οδηγία την οποία στήριξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμεί όμω πιστεύουμε κατηγορηματικά ότι σε εκείνη την απόφαση έχουμε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία που να λάβουμε υπόψη και τα, ανέλαβα, τα επανέλαβα σήμερα. Αυτά ενισχύουν την απόψη μα. Ότι η τρέχουσα οδηγία δεν έχει σωστή νομική βάση, δεν εναρμονίζει την εσωτερική αγορά, ούτε έχει ω αυθεντικό σκοπό την εναρμόνιση τη εσωτερική αγορά. Και θεωρούμε ότι δημιουργεί περισσότερους φραγμούς στο εμπόριο παρά ότι κάνει καλό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρώτησε αν έχω στοιχεία ότι μεγαλύτερε προειδοποίησει με φωτογραφίες πρόκειται να αυξήσουν το λαθρεμπόριο. Όχι, δεν έχω σημασία στοιχεία μαζί μου, διότι το παράνομο εμπόριο, το, το, το λαθρεμπόριο πρόκειται να το ενισχύσουν οι απαγορεύσει για προϊόντα τα οποία τώρα τα καταναλώνουν πάρα πολλοί καπνιστές. Και για τη μενθόλη, για τα λεπτά, τα τσιγάρα slim. Όταν δεν τα βρίσκουν τα προϊόντα τους, ε, τότε οι καπνιστές αυτών των προϊόντων πρόκειται να στραφούν άλλο Όμως, πολλοί από αυτούς μπορεί να προσθέσουν να βρουν κάπου αλλού ε, αυτά τα προϊόντα. Γιατί καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει απαγορεύσει τα slim τσιγάρα και τα τσιγάρα μενθόλης, όπως προτείνεται. Ευχαριστώ. Ο Γκάχάινς Φλόρεντς έχει συμπληρωματική ερώτηση. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο της καπνοβιομηχανίας. Όταν λέτε ότι η επιρροή της διαφήμιση δεν είναι και τεράστια ή ότι έχει αποδειχθεί ότι είναι σχετικά μικρή, ε, τότε γιατί φοβάστε ε, τι προειδοποιήσει. που δυστυχώς σας πεθαίνουν το χρόνο 700.000 πελάτες ως εταιρεία εγώ θα ήθελα να προσελκύσω καινούριου. Και η διαφήμιση δεν είναι πολύ σημαντικός παράγον εκεί. Κύριε Ρέρινγκ, για πείτε δύο λόγια για τη διαφήμιση παρακαλώ για να κλείσετε. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Ναι. Με χαρά να απαντήσω στην ερώτηση του κύριου Φλόρεντς. Η συσκευασία, λέγω, δεν παίζει ρόλο στο να αρχίσει κάποιος να καπνίζει. Το ίδιο μπορεί κανείς να ισχυριστεί και για τη διαφήμιση. Αλλά η διαφήμιση ουσιαστικά απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο Κοινοβούλιο πριν από 10 χρόνια συζητούσαμε την απαγόρευση διαφήμισης. Εδώ. Η συσκευασία, το πακέτο ενημερώνει τον καταναλωτή για το προϊόν που έχει ή τα προϊόντα για να επιλέξει. Και εμείς χρησιμοποιούμε και τη συσκευασία και την ε, διαφήμιση όπου επιτρέπεται για τα ποια είναι τα προϊόντα μας και να ενημερώνουμε τους καταναλωτές. Σας είπα, δεν θέλουμε να μπαίνουν τα παιδιά στο κάπνισμα. Δεν θέλουμε να αρχίζουν τα παιδιά να καπνίζουν. Αλλά θέλουμε να μπορούμε να πουλάμε τα προϊόντα μας ε, σε ενήλικες καταναλωτές που με τα λόγου γνώσεως αποφασίζουν να καπνίζουν. Και αυτό είναι και θέμα και της συσκευασία και του μάρκετινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε εδώ και αυτή την ενότητα. Ορίστε. Πολύ σύντομα θέλετε να απαντήσετε, όμως πάρα πολύ σύντομα, γιατί έχουμε ήδη καθυστέρηση. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Σε ό,τι αφορά ε, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναφέρθηκε επανειλημμένα από τον παρακαθήμενό μου. Θα ήθελα να σας παραθέσω, το δικαστή Κέσλερ το 2006 είπε ε, ότι ε, παραβιάζουν ομοσπονδιακούς νόμους οι καπνοβιομηχανίες και παραπλανούν το κοινό εμπολής για τους κινδύνους του καπνίσματος και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σχέση που έχουν ε, με την άρνηση ε, της καπνοβιομηχανίας ότι το μάρκετινγκ επηρεάζει τους νέους. Ε, εξακολουθούν να αρνούνται αυτό. Το γεγονός ότι ενέχονται ε, στη συμμετοχή τους και σε διαφήμιση εντύπων με μεγάλη απήχηση σε νεανικό κοινό. Κοιτάξτε παρακαλώ αυτή τη δικαστική απόφαση αν σας ενδιαφέρει να δείτε τι λέγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το θέμα. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε όμως εδώ και το δεύτερο πάνελ και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρέιλι, υπουργό, ε, για να κλείσει, για να φύγει. Ε, τον ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή, για την παρουσίαση και για τη σύνοψη. Έχετε το λόγο τώρα κύριε Υπουργέ και χαιρόμαστε που μας ήρθατε σήμερα. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μερικά σχόλια μου επιτρέπετε Να ευχαριστήσω ε, για την ε, εξαιρετική παρουσίασή της ε, και τα σχόλια την κυρία Περταλέτη. Ευχαριστώ και τον κύριο Ρέρινγκ που ήρθε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από όσα είπε. δεν είναι αξιόπιστα. λέτε ότι αν ενημερώνουμε περισσότερο τον κόσμο θα αλλάξει συμπεριφορά. Μα αν δεν αλλάξει συμπεριφορά τότε γιατί έχετε κατατρομάξει μιλάτε για μη δικαιολογημένη ανάμιξη. Άρα δεν είναι δικαιολογημένο το να σώνουμε ζωές, το να μειώνουμε το κόστος της δημόσιας υγείας, το να μειώνουμε ε, τα βάσανα του κόσμου που υποφέρει και να προστατεύουμε τους πολίτες και τα παιδιά μας. Νομίζω ότι έχουμε τέτοια ευθύνη και μάλιστα είμαστε δικαιολογημένοι να το κάνουμε αυτό. Είπατε ότι θέλετε να βοηθήσετε με ιδέες να σας ακούσω τα μέτρα που προτείνετε ε, σε συνδυασμό και ως προσθήκη των όσων εμείς προτείνουμε. Είναι πολύ ενισχυτικό αυτό που ακούσαμε από τη Λίντα Μακάβαν για την αύξηση των νέων αγοριών κυρίως που καπνίζουν. Τι λέτε λοιπόν στο Κοινοβούλιο ότι δεν έχετε ιδέα για αυτά και η βιομηχανία σας ε, ε, δεν έχει ανάμειξη. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Άντερσον για την υποστήριξή της, ε, για την οδηγία. Και λέει ότι το, ο καπνός σκοτώνει, σε ό,τι αφορά τα πιο εθιστικά στοιχεία και τις ουσίες, νομίζω το περιλαμβάνει η οδηγία. Τα γνωρίζουν αυτά οι, οι παραγωγοί μάλλον και οι μεγάλες μάρκες. Και σε σχέση με τόσο είπε η κυρία Μπαρταλέτη, αναφερθήκατε στον Καναδά. Ήταν τετραπλάσιος ο αριθμός των καπνιστών που δήλωσε πρόθεση να σταματήσει. Ίσως αυτή ήταν καλή αφετηρία από τότε που εφαρμόστηκε το σύστημα στον Καναδά. Επανειλημμένα μιλήσατε για διαφάνεια Μα όταν σας ρώτησε η κυρία Χάνς πόσους ε, λομπίστες απασχολείτε, δεν μας είπατε τίποτα. Ξέρουμε ότι είναι 97 οι λομπίστες εγγεγραμμένοι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρους απασχόληση στις Βρυξέλλες. Και ένας θεός ξέρει πόσα λεφτά ξοδεύετε για να τους πληρώνετε αυτούς και να υποστηρίζετε και άλλες τέτοιες δραστηριότητε. Θα σας πρότεινα το εξή. Μια λογική βιομηχανία που γνωρίζει σήμερα τους κινδύνους, γιατί τους γνωρίζει, θα πρέπει να ανακυκλωθεί και να επενδύσει σε άλλους κλάδους και άλλα προϊόντα που δεν έχουν τόσες ολέθριες συνέπειες. Οι προειδοποίησεις βοηθούν. Ξέρετε, εγώ ήμουν γιατρός ε, και ε, τους είπα όσοι ήταν διαβητικοί τύπου 1 ή τύπου 2 να γράψουν κάτι ε, ε, στο πακέτο των τσιγάρων για να το θυμούνται. Δηλαδή, ε, κάπνισμα συν διαβήτης ίσον θάνατος και κάθε φορά που πήγαινα πάνω ένα τσιγάρο να το βλέπαν. Και, και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγιακές παθήσεις ο διαβήτης και σε ακροτηριασμό. Λέτε ότι δαιμονοποιούμε τη βιομηχανία. Μα θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Και πώς τη λέτε μια βιομηχανία που παράγει ένα προϊόν που επίτηδες ε, δημιουργεί εσκεμένα εθισμό και τελικά ε, προσελκύει νέους και θα χάσει τη ζωή τους ο ένας στους δύο. Ορισμένοι σταματούν το κάπνισμα, αλλά άλλοι πεθαίνουν. 700.000 Ευρωπαίοι το χρόνο για να είμαι ακριβής. Και εσείς θέλετε να τους αντικαταστήσετε αυτούς, γιατί ε, από αυτό ζει, από τις ζωές τους η βιομηχανία σας. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί πραγματικά είναι θέμα ζωή και θανάτου για 700.000 Ευρωπαίους πολίτες το χρόνο. Και πάλι θα απευθύνω έκκληση προς του Ευρωβουλευτές. Χρησιμοποιήστε την εξουσία που έχετε για το καλό και για την υγεία των λαών μας. Ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, Βλέπετε ότι έχετε την υποστήριξή μας, είμαστε στο πλευρό σας. Θα χρησιμοποιήσουμε την εξουσία που έχουμε. Ελπίζω και εσείς να χρησιμοποιήσετε τη δική σας εξουσία στο Συμβούλιο για να περάσει αυτή η νομοθεσία και να έρθει σε αίσιο πέρας. Ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε στην ακρόασή μας σήμερα το απόγευμα. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στη δόκτωρα Μαρτίνα Πέτσχελάνγκε, που είναι ε, τμήματάρχη ε, στο τμήμα πρόληψης του καρκίνου στο Γερμανικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, θα ήθελα να προβάλλετε την πρώτη μου διαφάνεια. Υπάρχει πρόβλημα? Όχι. Καλησπέρα σας, καταρχήν, αγαπητά μέλη. Εκπροσωπώ το, Τμήμα Πρόληψης και Έρευνας για τον Καρκίνο και θα σχολιάσω την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προϊόντα καπνού και τη σχετική οδηγία. Θα ήθελα να σας προτρέψω να δείξετε όσο μεγαλύτερη φιλοδοξία γίνεται και παρακαλώ να λάβετε άμεση δράση. Έχουμε δημοσιεύσει αρκετές μελέτες και άρθρα σε έγκυρα περιοδικά και σε εφημερίδες για τα πρόσθετα και αυτό είναι και το αντικείμενο της σημερινής μου παρουσίασης. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την Διεθνή Συνένεση ε, για την απαγόρευση ή τη ρυθμίση όλων των προσθέτων του καπνού. Αυτό περιλάμβαναν οι μερικέ κατευθυντήριε γραμμέ για την εφαρμογή του άρθρου 9 και 10 τη ε, σύμβαση τη πλαίσιο της ΠΟΗ για τον έλεγχο του καπνού. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιήθηκε έντονα και προσπάθησε να αναπτύξει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του ΣΠΕΚ, τη σύμβαση της ΠΟΗ. Και γιατί ενεργοποιήθηκε τόσο δραστήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας περάσουμε παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια. Γιατί λοιπόν τα πρόσθετα, οι προσθετικές ουσίες θα πρέπει να απαγορευτούν από τα προϊόντα καπνού. Υπάρχουν επιστημονικά πορίσματα, υπάρχουν τεκμήρια, αλλά και δηλώσεις ε, της καπνοβιομηχανίας. Για παράδειγμα, ο Πίτερ Σμάρκιν ε, του Μπόρτα, Το British, η ε, ο Συνεγός για το Καπνού, είπε ότι προσπάθησα να κάνω πιο εύπεπτο τον καπνό και να περιορίσω την τραχύτητα και την ε, αερεθισμό. Γι' αυτό ακριβώ χρησιμοποιεί η καπνοβιομηχανία τα προσθετικά. Και μάλιστα ε, μάθαμε και από έρευνα και από άρθρα ότι τα πρόσθετα στον ε, καπνό μπορούν να βελτιώσουν την καλή γεύση, την, την ελκυστικότητα του καπνού και μια ήπια γεύση και, και να οδηγήσουν σε αύξηση της κατανάλωσης του καπνού και άρα να αυξήσουν το κίνδυνο της υγείας, να αυξήσουν την νοσηρότητα και την θνησιμότητα. Επιτρέψτε μου να σας δείξω τρεις διαφάνειες για τα επιστημονικά πορίσματα. Η πρώτη διαφάνεια αφορά τα σάκχαρα, η, τη ζάχαρη ή συναφή προϊόντα, όπως τη γλυκόζη, τη φρουκτόζη, το μέλι και άλλα τέτοια προϊόντα γλυκαντικά τέτοιου είδου γλυκαντικές ουσίες βελτιώνουν τη γεύση του καπνού, μειώνουν την τραχύτητα και αυξάνουν ε, την ε, καλή γεύση και μάλιστα σε ό,τι αφορά το, τον τρόπο καύσης είναι εξίσου καρ, καρκινογόνες αυτές οι ουσίες. Και μάλιστα αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Και να επιστρέψω στην ζάχαρη. Γιατί επιτρέπουμε την γλύκαρση του δηλητηρίου, της δηλητηριώδης αυτής της ουσίας που είναι ο καπνός. Γιατί επιτρέπουμε τέτοια διαδικασία. Επόμενο θέμα, επόμενη διαφάνεια, μεθόλη. Έχουμε πολλές καλές έρευνες που μας λέει ότι απλώς συγκαλύπτει την τραχύτητα του καπνού η μεθόλη. Και μπορώ να σας δώσω και στοιχεία. Γνωρίζουμε ότι αυτό το, φρε... το φρεσκαριστικό αποτέλεσμα που έχει είναι παυσίπονο και ε, ναρκώνει κατά κάποιο τρόπο τον ε, το ουρανίσκο. Το χρησιμοποιούμε μάλιστα τη μενθόλη σε προϊόντα κατά πολέμηση του βήχα. Βελτιώνει επίση την εισπνοή. Μπορεί κανεί να εισπνεύσει πολύ πιο βαθιά όταν το προϊόν που εισπνέει έχει μενθόλη. Γνωρίζουμε τα αποτελέσματα τη μενθόλη και τι προκαλεί. Και γνωρίζουμε ότι τα σιγαρέτα με μενθόλη μέχρι στιγμής είναι μικρό μερίδιο της αγοράς στην Ευρώπη, αλλά η καπνοβιομηχανία προτίθεται να επεκτείνει αυτό το μερίδιο της αγοράς. Το γνωρίζουμε αυτό από τα έγγραφα της ε, καπνοβιομηχανίας και από τις ε, ομιλίες και τα πρακτικά συνεδριάσεων. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ετοιμαστούμε για μια αύξηση της αγοράς, της αγοράς τέτοιων προϊόντων. Άλλωστε, μην ξεχνούμε ότι ε, ο συνδυασμό μεθόλη με άλλε ουσίε προσθετικέ ε, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το προϊόν του καπνού. Και το χρησιμοποιούν ήδη πολλέ βιομηχανίε. Δεύτερο, τρίτο στοιχείο, η γλυκόριζα επίση αυξάνει τη γεύση, βελτιώνει τη γεύση, την κάνει πιο εύγευστο το καπνό, το δηλητήριο ουσιαστικά, βελτιώνει τη γεύση και υπάρχουν και για τη γλυκόριζα αρκετά στοιχεία που δείχνουν το καρκινογόνο της αποτέλεσμα σε περίπτωση καύσης της γλυκόριζας. Και μάλιστα όταν γίνεται η σπνοή του καπνού. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε πρόσθετα χωρίς γεύσεις ή αρώματα. Κάποιες δεσμευτικές ουσίες, κάποιες εγραντικές, χρωστικές, που επίσης είναι καρκινογόνες ουσίες και έχουμε επίσης επιστημονικά τεκμήρια που το αποδεικνύουν. Ακόμη και πρόσθετα που δεν έχουν ιδιαίτερη γεύση αυξάνουν την, ε, τον χαρακτήρα του προϊόντος. Και τώρα ερχόμαστε σε μια αγορά που αποτελεί και το αντικείμενο της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ζητά απαγόρευση τη εμπορία προϊόντων καπνού με χαρακτηριστικέ γεύσει. Φυσικά θα πρέπει να απαγορευτεί η εμπορία τέτοιων προϊόντων. Φυσικά είναι απαράδεκτο μενθόλη, ε, βανίλια ή γεύσεις μάγκο ή άλλων εξωτικών φρούτων να συμπεριλαμβάνονται σε τσιγάρα, αυξάνοντας ε, την ε, ελκυστικότητά τους ενώ αυτή τη στιγμή η αγορά αυτών των προϊόντων έχει μικρές διαστάσεις, ε, αυξάνεται όλο και περισσότερο. Υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί η έναρξη καπνίσματος από νέους εξαιτίας της ε, θεκτικότητας αυτών των προϊόντων. Βέβαια η μεγάλη αγορά προϊόντων είναι άλλη, είναι αλλού. Και αυτή η μεγάλη αγορά προϊόντων καπνού θα πρέπει να ρυθμιστεί. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ποιες είναι οι κυρίαρχες μάρκες στην αγορά προϊόντων καπνού και όλες αυτές οι ουσίες. Όλα αυτά τα μείγματα προσθέτων, προσθετικών ουσιών προσθέτων επιτρέπουν την καπνοβιομηχανία να τα συμπεριλάβει στο προϊόν προκειμένου να γίνει πιο εύγευστο, να μειωθεί η ε, διέγερση που προκαλεί, να μειωθεί ο ρυθμός που προκαλεί και η τραχύτητά του και άρα να, να αυξηθεί το κάπνισμα. Επίσης, ε, η, η αλληλεπίδραση των διαφόρων προσθέτων είναι επικίνδυνη. Ακόμη και το μείγμα μικρών ποσοτήτων διαφόρων προσθέτων έχει τα ίδια αποτελέσματα με χρήση μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός και μόνο προσθέτου. Οπότε, το, ε, το μείγμα προσθέτων έχει ακόμη μεγαλύτερη καρκινογόνο δράση. Ενώ ακριβώς επειδή το μείγμα αποτελείται από μικρές ποσότητες των επιμέρους προσθέτων, δεν πληρούνται τα κατώ, κατόφλια. Ενώ το αποτέλεσμα μετά την καύση είναι εξίσου επιβλαβές και καρκινογόνο. Και περνάμε τώρα στις νέες τεχνολογίες που υιοθετήθηκαν προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των τσιγάρων και να, να προσελκυστούν περισσότεροι εμ, καταναλωτές. Πρόκειται για, τις, ε, για τα πιπάκια που υποτίθεται ότι φιλτράρουν ε, την νοικοτήνη ή τα πρόσθετα. Που μπορούν μάλλον να ε, ε γεμίσουν πρόσθετα και να φιλτράρουν την νοικοτήνη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πρόσθετα που μπορούν να βελτιώσουν την ε, καλή γεύση και να μειώσουν τον ερεθισμό από τον ε, καπνό για να περιοριστεί η έναρξη του καπνίσματος αλλά και να βοηθήσουμε όσους καπνιστές θέλουν να απεξαρτητοποιηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να απαγορεύσουμε όλα τα πρόσθετα που είναι καρκινογόνα είτε πριν είτε μετά την καύση για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές και να περιορίσουμε την οσιρότητα και την θνησιμότητα. Επίσης κάτι που δεν θα πρέπει να γίνει είναι να τεθούν ανώτατα όρια για, για τα πρόσθετα. Γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αξιόπιστες μεθόδους για να επιλέξουμε την κατάλληλη οριακή τιμή για τα διάφορα πρόσθετα, τις διάφορες γεύσεις. Και υπάρχουν και οι αλληλεπιδράσεις ε, και η συνέργεια του, ε, από το μείγμα των προσθέτων. Ε, είτε γίνεται εισαγωγή από το στόμα είτε από την ε, μύτη. Οπότε οποιαδήποτε πρόσθετο βελτιώνει την γεύση και περιορίζει τον ρυθμό, θα πρέπει να απαγορευτεί. Επίσης να απαγορευτούν τα πρόσθετα που είναι ε, καρκινογόνα είτε πριν είτε μετά την καύση και οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι οποιοδήποτε πρόσθετο χρησιμοποιούν είναι πραγματικά ακίνδυνο, τελείως αυλαβές και θα πρέπει να χορηγούν τα επιστημονικά κριτήρια και να προτείνουν ε, κατάλογο για την απαγόρευση των προσθέτων ή την, τον αποκλεισμό ορισμένων προσθέτων από την απαγόρευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάγκερ. Τώρα το λόγο έχει ο Λίκ ε, από την Ένωση των Αντικαρκυνικών ε, Ενώσεων των Κρατών Μελών. Ε, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ ε, θα αναφερθώ στο θέμα του λαθρεμπορίου. Το έχω ερευνήσει από το 1992 έχω δημοσιεύσει αντίστοιχα άρθρα. Γιατί το αναφέρω αυτό. Διότι κάνουν κάποιους ισχυρισμούς οι βιομηχανίες που δεν ε, ελέγχονται σε επιστημονικά έντυπα. Πριν από 20 χρόνια μας έλεγε η βιομηχανία ότι ήταν πολύ εύκολο το πρόβλημα του λαθρεμπορίου και είχε να κάνει με το ύψος φορολόγησης. Όταν ήταν υψηλή η φόρη ήταν μεγάλο το λαθρεμπόριο, όταν χαμηλή η φόρη, ειδική φόρη κατανάλωσης μειώνεται. Η ε, ε, πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Η Δανία έχει υψηλού φόρους και χαμηλό λαθρεμπόριο και η Ισπανία που είχε τους χαμηλότερους ειδικού φόρους είχε τεράστιο λαθρεμπόριο. Ενώ η Ιταλία ε, είχε και ε, χαμηλούς φόρους και μεγάλο λαθρεμπόριο. Για ποιο λόγο. Διότι ε, η ίδια βιομηχανία οργάνωνε το λαθρεμπόριο. Αυτό δεν ήταν μόνο δική μου ε, άποψη, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1997 στην Αρμόδια Επιτροπή και αυτό έλεγε και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε για την βιομηχανία καπνού. Αποτέλεσμα το 2004 η Φίλιπ Μόρις κατέληξε σε ένα συμβιβασμό και πλήρωσε ε, εκατομμύρια και στον Καναδά 1,7 ε, δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια αντίστοιχε εταιρείε. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν και δεν ε, έχουν υποτροπιάσει. Η JTI όμως τον Νοέμβριο του 2011 ε, επανήλθε. Ε, ποιος είναι ο λόγος που οδηγεί ε, στο λαθρεμπόριο. Είναι περίπλοκα τα πράγματα. Είναι θέμα ζήτησης και αγοράς και προσφοράς. Και οι εταιρείε και νόμιμες και παράνομες θέλουν να αυξήσουν το κέρδος τους και με τη διαφορά φθορά μπορούν να προάγουν εγκληματικά δίκτυα γιατί και οι χώρες έχουν χαμηλή δυνατότητα. Δεν είναι μόνο η τιμή λοιπόν που ορίζει αυτές τις καταστάσεις, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες και η προσφορά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη ζήτηση και η επιρροή της. Έχουμε κάνει μια μελέτη εμείς σε 18 ευρωπαϊκές χώρες ε, που ε, δημοσιεύθηκε σε μια επιστημονική ε, επιθεώρηση. Και μελετήσαμε λοιπόν το λαθρεμπόριο σε 18 χώρες και δείχνουν τα στοιχεία ότι το λαθρεμπόριο δεν συνδέεται άμεσα με την τιμή των προϊόντων καπνού και είναι πιο ευρέα ε, διαδεδομένων σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Μολδαβία ή τη Λευκορωσία. Λετωνία, Λιθουανία δηλαδή και ε, λοιπές χώρες που συνορεύουν ε, προς τις προηγούμενες. Τι ισχυρίζεται λοιπόν η βιομηχανία. Έχει λανσάνει μια καμπάνια που λέει ότι θα αυξηθεί το παράνομο εμπόριο εάν είναι λευκό το πακέτο ή ε, ενιαίο. Αυτό είναι από την ιστοσελίδα της Φίλιπ Μόρις και λέει ότι διάφοροι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι αν είναι ενιαίο το πακέτο θα αυξηθεί το λαθρεμπόριο και θα είναι πιο εύκολο να αντιγραφούν τα τσιγάρα. Πιο εύκολο και πιο φτηνό μάλιστα. Κοιτάξτε εδώ ε, το πακέτο. Η JTI στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης ε, έχουν ε, λευκή συσκευασία για να ε, δείξουν το ενιαίο πακέτο. Μα δεν θα είναι λευκό. Θα έχουν φωτογραφίες με προειδοποίηση. Αυτό θα είναι το ενιαίο πακέτο. Δεν θα είναι λευκό. Ε, και τώρα λέγουν ότι βεβαίως αυτές οι φωτογραφίες για τις προειδοποίησεις υγείας μπορεί να βοήθησαν, μπορεί να μην βοήθησαν. Και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι, και δύσκολο να αντιγραφεί, είναι η μάρκα και αυτά ανοησίες είναι. Γιατί, τι εννοώ. Τι λέει η καπνοβιομηχανία. Κάθε προϊόν είναι εύκολο να αντιγραφεί. Οτιδήποτε σχεδιάζεται μπορεί να, ε, να αντιγραφεί. Και αυτό το γνωρίζει και η Φίλιπ Μόρις. Ε, για ένα σύστημα ανείχνευσης και εντοπισμού και ε, κωδικό. Οτιδήποτε σχεδιάζεται, και ακόμα και το πιο ο δύσκολο και τα πιο δύσκολα γραμματώσιμα ή οτιδήποτε, τρει εβδομάδε αρκούν για να αντιγραφούν. Οτιδήποτε μπορεί κανείς να δει με το γυμνό μάτι αντιγράφεται. Ε, και είναι και πιο ε, φτηνό, λέει η βιομηχανία. Δεν ισχύει αυτό. 10 με 12 cents κοστίζει η αντιγραφή. Μάλλον το κόστος παραγωγής, συγγνώμη. Ακόμα και γίνουν από εκεί οικονομίε, οικονομίες. Τι οικονομίες θα είναι, ένα σέντ, δύο σέντς ε, σε ένα πακέτο που κάνει από 4 μέχρι 10 ευρώ. Και πάλι ε, εγώ σας παραπέμπω σε έγγραφα της Φίλιπ Μόρι, που δείχνει ότι το κόστος παραγωγής και συμφωνεί η εταιρεία είναι πολύ χαμηλό. Τώρα, πια η μελέτη σκοπιμότητας και αντικτύπου που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε στη σελίδα 93 στο ίδιο συμπέρασμα. Ε, ισχυρίζεται η βιομηχανία ότι το ενιαίο πακέτο θα αυξήσει το λαθρεμπόριο. Ωστόσο δεν ε, έχουν υποβληθεί πιστικά στοιχεία. Έχει αναφερθεί αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο τι λέγουν στη σελίδα 20 της αντίστοιχης έρευνας ότι τα τυποποιημένα ε, πακέτα θα πρέπει να έχουν φωτογραφίες και έγχρωμες ε, προειδοποίηση ε, και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν θα είναι λευκά τα πακέτα. Και επίσης ήδη από σήμερα είναι σε θέση οι παραχαράκτες, οι εκείνοι που κάνουν τι απομίσεις να τα αντιγράφουν. Οπότε ας μην λέμε νοησίες για το ενιαίο πακέτο και το τυποποιημένο, ότι θα αυξηθεί το λαθρεμπόριο. Ε, και επίσης η απαγόρευση ε, προβολής θα οδηγήσει σε μείωση. Η διαφήμιση έχει απαγορευτεί και επίσης στον Καναδά από τον Ιούλιο του 2010 απαγορεύονται οι πρόσθετες αρωματικές ουσίες. Και έχει μειωθεί σημαντικά και το λαθρεμπόριο που και πάλι δείχνει ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν είναι άσπρο μαύρο όπως ισχυρίζεται η βιομηχανία. Έρχομαι και πάλι στο πρωτόκολλο λαθρεμπορίου που εγκρίθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 2012 στην Νότια Κορέα. Για να είμαστε σαφείς, περί τίνος πρόκειται. Έχει εγκριθεί αυτό, δεν έχει εφαρμοστεί. Θα πρέπει να κυρωθεί από 40 χώρες. Μέχρι τώρα 13 έχουν υπογράψει αυτό το πρωτόκολλο, αλλά χρειάζονται 40 κυρώσεις για να τεθεί σε ισχύ. Το πρωτόκολλο λοιπόν για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου είναι μια διεθνή σύμβαση και ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, μοναδικά ασφαλή και μη αφαιρούμενα χαρακτηριστικά σε όλα τα πακέτα και σε όλες τις συσκευασίες ε, και στις κούτες ε, ε, τσιγάρων, όχι μόνο στα πακέτα ή γενικότερα στις μεγαλύτερες συσκευασίες. Θα πρέπει λοιπόν να επιβληθεί μια υποχρέωση και για την εξωτερική συσκευασία, όχι μόνο το πακέτο αυτό καθ' αυτό. Και ποια είναι μία από τις σαφείς λοιπόν υποχρεώσεις στο πρωτόκολλο αυτό είναι το άρθρο 8 για τις υποχρεώσεις και το ρόλο της βιομηχανίας. 8.2. το 8-12 μάλλον. Ε, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ένα υπογράφο ε, μέλος δεν θα πρέπει να ε, ανατίθενται στη βιομηχανία καπνού. Είναι μεγάλη ιστορία λοιπόν ε, της συνενοχής της βιομηχανίας και πάλι παραμένει να κατηγορείται μια μεγάλη εταιρεία ότι οργανώνει το λαθρεμπόριο ίδια. θα πρέπει να έχουμε στοιχεία λοιπόν ανιχνησιμότητας ε, και μια εταιρεία να επιλέξουν τα κράτη-μέλη που θα αποθηκεύει τα στοιχεία αυτά ε, με βάση και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα πρέπει να φυλάσσονται στα στοιχεία σε επίπεδο κράτους και Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ένα εταιρεία όπως ορίζουν οι σημερινές προτάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα πολύ σημαντικό επίσης, αν θέλετε να έχετε ανευσιμότητα ή χνηλασιμότητα θα πρέπει να συνδέεται ε, η εξωτερική συσκευασία με τα μοναδικά ε, χαρακτηριστικά και ταυτοποίησης του πακέτου. Γιατί αν είναι μόνο στο πακέτο πρέπει να ανοίξει κανείς την παλέτα, ε, τις κούτες, ε, τα χαρτόκουτα για να φτάσει στο τελικό πακέτο, να βγάλει ένα πακέτο και να δει το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει η εξωτερική συσκευασία να φέρει ε, διακριτικά. Συμπέρασμα. Δεν θα αυξηθεί το λαθρεμπόριο όπως ισχυρίζεται με το ενιαίο πακέτο, όπως ισχυρίζεται η βιομηχανία. Ε, κάθε πακέτο μπορεί να αντιγραφεί και μάλιστα εύκολα και κάθε συσκευασία. Και η επιλογή της εταιρεία ε, που θα διατηρεί τα στοιχεία θα πρέπει να είναι απόφαση των κρατών μελών και η υποχρέωση ανιχνευσιμότητας δεν θα πρέπει να ανατίθεται ή να υλοποιείται από την ίδια την καπνοβιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Γιώσενς. Επόμενος ομιλητής είναι ο Δόκτωρ Ντέιβιτ Χάμοντ, ε, αναπληρωτής καθηγητής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Συστημάτων Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Βατερλού στον Καναδά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ με μεγάλη μου χαρά. Απευθύνω το λόγο σήμερα και μου ζητήσατε να συζητήσουμε τα στοιχεία που υπάρχουν όσον αφορά τη συσκευασία, την ειδικατοθεσία σε σχέση με την διατάξη της νέα οδηγία και άλλωστε τα συζητήσαμε ε, ε, και ο Ντέβιτ, πριν τέλο πάντων, ε, και εγώ Ντέβιτ, αλλά είναι απλώ αυτό μια σε μια σύμπτωση έχουμε επομένως ε, μια ομάδα που αφορά ε, το, το, το πακέτο χωρίς διακριτικά, χωρίς φωτογραφίες και έχουμε επίσης και άλλα στοιχεία που θα σας δείξω και έχουμε επομένω ε, το, μάρκετινγκ και την διαφήμιση που έχει παίξει πάρα πολύ σημαντική, σημαντικό ρόλο όσον αφορά το τι έχει γίνει, πώς έχουν υποθεί συμπεριφορές των καταλωτών για το τσιγάρο. Που, τώρα πολύ πρόσφατα χάσαμε κάποιους διάβλους λόγω της ε, της νομοθεσίας, οπότε ακριβώς επειδή απαγορεύονται οι διαφημίσεις είναι σημαντικό το πώς γίνεται η συσκευασία και οπότε θα πρέπει όσο γίνεται πιο νωρίς να τους αγγίξει τους, ε, τους ενδυνάμει καπνιστές και ε, ναι, δεν είναι θέμα να προβάλλει το τσιγάρο το ίδιο, αλλά το, το lifestyle, τον τρόπο ζήτηση σχετίζεται με το τσιγάρο και επομένω βλέπουμε ότι αυτή η διαφήμιση έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια καπνιστές και χιλιάδες φορέ τη, τη, βλέπει ο καπνιστής το πακέτο και επίσης προβάλλονται πάρα πολύ τα πακέτα. Τα βλέπουν και οι μη καπνιστές, τα βλέπουν και οι νέοι, εκεί που πουλιούνται λιανικά και σε άλλους χώρους. Τώρα δεν θα συζητήσω τώρα. Ε, να δούμε τώρα τι θα γίνει με, με, με τρία-τρία σημεία. Να δούμε αυτό το, το κλασικό ή τέλο πάντων το, το, την, την απλή συσκευασία. Να πω είναι το, το πακέτο. Ε, αυτό είναι τυποποιημένο ε, και βάσει τη νομοθεσίας έχουμε αυτές τις ε, προειδοποίησεις και επειδή έχουμε ε, πολλές παραλλαγές ε, σε, κάθε τσιγάρο έχουμε και αντίστοιχε προειδοποίησεις εδώ έχουμε το 2012 και η Νέα Ζηλανδία είπε θα ακολουθήσει αυτόν τον, τον τρόπο επισήμανσης στην Αυστραλία έχουν γίνει διάφορες προσφυγές σε σχέση με αυτού του είδους την, την, τη συσκευασία και το αστυνομικό δικαστήριο τελικά πέριψε την προσφυγή για λόγους δημοσίας υγείας, οπότε ακόμα νωρίς να αποτιμήσουμε ποια, ποιος είναι, ποια είναι η επιπτώση στην Αυστραλία, γιατί αυτό έχει μόλις ε, πολύ πρόσφατα. Και έχουμε εδώ πέρα επομένως διάφορες άλλες ε, μελέτες, ε, άλλα στοιχεία, κυβερνητικέ έρευνε στην Αυστραλία. Πάντω τα πιο αξιόλογα στοιχεία προέρχονται από την μηχανία. Και εδώ έχουμε να κάνουμε κάποια εμπιστευτικά έγγραφα που με δικαστική απόφαση υποχρεώθηκαν να δημοσιεύσουν για τη στρατηγική τους οι και οπότε υπάρχουν επομένω αδιάστα στοιχεία ότι η συμπεριφορά του καπνιστή, του καταναλωτή επηρεάζεται από το, το τσιγάρο. Όταν ξεκίνησε επομένω αυτό το πακέτο το ασημένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυξήθηκε η πώληση αυτών των τσιγάρων σε σχέση με άλλε διαφημίσει Επίσης ε, υπάρχουν κάποιο είδους ε, ε, ψευδείς πεπιθήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στην υγεία. Μπορεί να θεωρηθούν ότι κάποια τσιγάρα, ότι είναι mild, δηλαδή πιο ήπια, βλάπτουν λιγότερο από άλλα. Και επίσης υπάρχουν διάστα στοιχεία ότι ιδίω μεταξύ των νέων πιάνουν το από αυτού του είδους τα τα πακέτα και βλέπουμε ότι εάν δεν, ε, είναι, δεν προβάλλεται, δεν είναι, είναι το πακέτο, δεν το προτιμάει ο νέος. Επομένως θα δούμε ε, κατά πόσον θα έχουμε μείωση στους νέους ή στους ε, ενήλικες καπνιστές. Εμεί πάντως θεωρούμε δεν θα έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις αυτή η αλλαγή στην, στο, στο, στο πακέτο, στην συσκευασία. Από την άλλη μεριά όμως ε, θεωρούμε ότι για τους νέους θα υπάρχει, θα υπάρχει μείωση γιατί μέσω των νομίμων προϊόντων θα υπάρξει κάποια, κάποια ωφέλεια. Και στον Βασίλειο θεωρούμε ότι θα έχουμε και 1% να είναι επιπτώσεις, σημαίνει τα εκατομμύρια καμιστών κάποιες χιλιάδες. Επίσης, μειώθηκε το μέγεθος των πακέτων στην Αυστραλία. Ε, να τώρα ποιο είναι το νόημα πακέτο των λεπτών slim τσιγάρων σε σχέση τώρα με τη ρύθμιση της μιας οδηγίας. Τα slim και τα super slim είναι η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο κομμάτι της αγοράς των τσιγάρων. Ο τρόπος ανοίγματος του πακέτο, το σχήμα του κλπ. έχουν σημασία και έχει γίνει επομένως έρευνα που καταδεικνύει ότι θεωρούν ε, ο κόσμος ότι τα, τσιγάρα έχει λιγότερη πίσα που δεν έχει και ότι ε, τα slim ε, βοηθούν περισσότερο να αδυνατήσει κανείς να μην παχύνει τέλο πάντων. Έχουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες από την Επιτροπή Οικονομικής Έρευνας της Ευρωπαϊκής ότι 46% και 30% των των, των κοριτσιών, 30% των αγοριών καπνίζουν για να ελέγξουν το βάρος τους και 80-90% ε, ξεκινά, των καπνιστών αρχίζουν να καπνίζουν όταν είναι ανήλικοι. Επίσης ε, τα slim κυρίως πουλούνται σε νέες γυναίκες. Εδώ έχετε ε, αυτό το έγγραφο της Φίλιπ Μόρις του 1986 που σας δείχνει ποια ηλικία στοχεύει. Τώρα έχουμε άλλες συνέπειες του, του σχήματος. Αυτά τα καινούργια super slim ε, διαστρεβλώνουν τις προειδοποίησεις για την υγεία. Να βλέπετε εδώ πέρα από τον Καναδά ένα πακέτο, δύο πακέτα και βλέπετε ότι στα αριστερά είναι τόσο μικρή η φωτογραφία που σχεδόν ε, δεν μπορεί να διαβάσει κανείς και έτσι αλλοιώνεται και το κυβερνητικό μήνυμα και επίσης ε, άρα έχει λιγότερες επιπτώσεις η προειδοποίηση στο SLIM παρά στο παραδοσιακό πακέτο. Τέλος, για αυτές τις προειδοποίησεις σχέση με την υγεία θα πρέπει να πούμε ότι ε, γίνεται επικοινωνία μέσω του πακέτου και από την κυβέρνηση και βλέπουμε εδώ ότι έχουν πάνω από 100 δημοσιευμένες μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά. Και μέσω διαφόρων μέσων ανείχνευσης έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και όπως είπαμε προηγουμένως έχουμε και τις αποφάσεις των δικαστηρίων και δεν αποδείχθηκε ε, ότι τα δικαστήρια ε, απορρίπτουν τις προσφυγές κατά των ε, πρωτοποίησεων. Υπάρχουν αποφάσεις υπέρ και άλλες κατά. Ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. Έχουμε διάφορες αποφάσεις και δεν ξέρω πάντως εγώ καμία υπόθεση όπου το δικαστήριο να καταδίκασε τις ε, επισημάνσεις, τις ειδοποίησεις σε σχέση με τα τσιγάρα. Άρα, πού καταλήγουμε ότι οι μεγάλες φωτογραφίες που προδοποιούν ε, βοηθούν αυτούς που να κόψουν το κάπνισμα. Πάντως, ο βασικός στόχος δεν είναι αυτός, αλλά πριν την ηλικία που κανείς τίνει να αρχίσει το τσιγάρο, να τον έχει προειδοποιήσει, τον έχει αποτρέψει. Και έχουμε το 16% των μη καπνιστών που θυμούνται αυτά τα μηνύματα από τα πακέτα. Και 4 στους 10 ε, Άγγλους που δεν καπνίζουν είπαν ότι ε, δεν έξανε ποτέ ακριβώ λόγω αυτών των ε, μηνυμάτων. Και έχουμε επίσης δημοσιευμένες έρευνες ότι δηλαδή ε, αυτές οι φωτογραφίες είχαν σημαντική, σημαντικό αποτέλεσμα τελικά. Και από τον Καναδά και θα πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ ότι μόλις οι ειδοποιήσεις αυτές είχαμε ρεκόρ ε, μειωμένης από τα, το, το, το, το καλύτερη επίδοση τα τελευταία 16 χρόνια. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω του διεθνού μέσου όρου, γιατί έχουμε είπαμε 50 χώρε διεθνώ που έχουν τέτοιε. Επίση, βλέπετε εδώ κάποιε χώρε που έχουν τέτοιε ε, φωτογραφίε που δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπετε εδώ πέρα το μέγεθο σε με το πακέτο αναχώρα και ενώ στα ευρωπαϊκά πακέτα είναι στη μία πλευρά του πακέτου, αλλού είναι και στις δύο. Και έτσι προβάλλονται καλύτερα στο σημείο πωλήσεως ε, αυτές οι προειδοποίησεις. Πάντως, ε, τίνει να τονίσει το μήνυμα όσο περνάει ο χρόνος και ας, πολλές χώρες ανανεώνουν το μήνυμα στα 10 χρόνια. Επίσης για το περιεχόμενο είναι το ότι θα πρέπει κανείς να, είναι, να έχει αξιοπιστία να γίνει πιο δυνατό μήνυμα, να, είναι πιστικό, να, χρησιμοποιεί φωτογραφίες από πραγματικά πρόσωπα. Να υπάρχουν επομένως πληροφορίες εκτός από το σοκ και για αυτούς που θέλουν να κόψουν το τσιγάρο. Πάντως θέλω να σας πω ότι πέραν όσων είπαμε είναι πάρα πολύ άμεσο το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Βλέπετε αριστερά ένα πακέτο ε, που για το 2000 και ε, περιγράφει το τι γίνεται στα δεξιά όμως κάτι το οποίο πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά ε, διεθνίζει το τσιγάρο, δεν το δεν, δεν, αποθαρρύνει το κανονισμό. Ε, νομίζω αυτό πέραν των, των στοιχείων το λέει και η κοινή λογική και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, ε, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για την παρέμβαση της καπνοβιομηχανίας σε πολιτικές ελέγχου του καπνού και τι πρέπει να κάνουμε. Είμαστε μια ερευνητική οργάνωση με το, το μεγαλύτερη έρευνα από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και κυρίως ε, ερευνούμε για την πρόληψη του καρκίνου. Και φυσικά ασχολούμαστε με τον καπνό, γιατί ένα τέταρτο όλων των θανάτων εξαιτία καρκίνου οφείλονται σε... έχουν σχέση με το κάπνισμα. Οπότε οτιδήποτε λέμε για το θέμα αυτό στηρίζεται σε αδιάστα επιστημονικά κριτήρια. Παρά τις εσφαλμένες, από εσφαλμένους χειρισμούς ότι δεν έχουμε επιστημονικά κριτήρια. Λοιπόν, γιατί είμαστε κατά τη καπνοβιομηχανία. Τι έκανα η καπνοβιομηχανία για να εμποδίσει την αρχική οδηγία προϊόντο καπνού του 2001. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από τη σύμβαση πλαίσιο τη ΠΟΕ για τον έλεγχο του καπνού. Τι λέει το 5.3. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τηρήσουμε τις υποσχέσει μα από τη Συμφωνία Πλαίσιο. Γιατί είμαστε ε, κατά της καπνοβιομηχανίας. δεν έχουμε ακούσει πολλά για το πώς προσπάθησε να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προστασία των πολιτών. Γιατί έχουμε αποδείξεις που, που δείχνουν ότι κάποια βιομηχανία έχει διαστρεβλώσει τα επιστημονικά κριτήρια, προσπάθησε να, να αποσιωπήσει ε, επιστημονικές μελέτες, χρησιμοποιήσει μεροληπτικές μελέτες και μάλιστα χρησιμοποίησε κάποια κριτήρια που κάποιες ε, ομάδες που συνδέονται και με τα δικά της συμφέροντα ε, και μάλιστα διευκόλυνε το λαθρεμπόριο, χρησιμοποίησε πρόσθετα για να αυξήσει την ελκυστικότητα και την εθιστικότητα των προϊόντων καπνού ε, προς τα παιδιά και στοχεύει κυρίως η βιομηχανία στα φτωχούς γυναίκες και παιδιά. Και μάλιστα βλέπουμε ότι εκατοντάδες μνήες υπάρχουν για τέτοια στοιχεία και αδειάστε επαναλαμβάνω κριτήρια και αποδείξεις και επιστημονικά πορίσματα. Δεν έχουμε ένα συνηθισμένο καταναλωτικό περιόν καταναλωτικών προϊόντων. Ε, μακροπρόθεσμα θανατώνει ένα στους δύο χρήστες. Οπότε, όπως δείχνουν και οι έρευνες, η καμπροβιομηχανία αρνείται το, τον επιβλαβή χαρακτήρα των προϊόντων και χρησιμοποιεί ε, τα πρόσθετα για να προσελκύσει παιδιά. Δεν είναι επιλογή ενήλικα, είναι ένα εθισμό που ξεκινάει στην παιδική ηλικία. 150.000 μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 11 με 15 χρόνια, ξεκινούν κάθε χρόνο το κάπνισμα. Φανταστείτε πόσα παιδιά ξεκινά να καπνίζουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Πώς λοιπόν προσπαθεί η καπνοβιομηχανία να εμποδίσει την έγκριση της οδηγίας ε, για τα προϊόντα καπνού, όταν πρώτο υποβλήθηκε το 2001. Ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, εξαιτίας κάποιων αντιδικιών, εκατομμύρια σελίδες στο ίντερνετ και επιστημονικές μελέτες ενέκυψε σε αυτό το θέμα και έχουμε μια μακροσκελή έρευνα στην ιστοσελίδα του Smoke Free Partnership και έχουμε τρία βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις οδηγίες. Ότι βρισκόταν εκτός το πεδίο αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αντέβαινε σε υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες και θα έχει δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα. Ε, είναι τα γνωστά επιχειρήματα που ακούσαμε και σήμερα. Και μάλιστα πολύ συχνά η καπνοβιομηχανία χρησιμοποιεί ανεδαφικά επιχειρήματα. Γιατί το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να καθυστερήσει τα πράγματα, όχι όμως με δαπανηρές δικαστικές ε, προσπάθειες και διαδικασίες. Και αντίστοιχη προσπάθεια είχαμε και στην ε, οδηγία για τα προϊόντα του καπνού. Περνάμε λοιπόν στο άρθρο 5.3 τη σύμβαση πλαίσιο της ΠΟΗ για τον έλεγχο του καπνού που θέλει να προστατεύσει τους ε, πολίτες από τον καπνό με διάφορα μέτρα. Είναι σαφές ότι η ΠΟΗ και 176 χώρε που έχουν κυρώσει αυτή τη σύμβαση πλαίσιο γνωρίζουν ότι η καρβιομηχανία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά όχι ο συνηθισμένος αντισυμβαλόμενο ή ενδιαφερόμενο. Το 5.3 λέει ότι υπάρχει ασυμφιλίωτη και θεμελιώδης ε, σύγκρουση ξεπέριστη μεταξύ των συμφερόντων της καπνομηχανίας και των συμφερόντων δημόσιας υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα για τον έλεγχο του καπνού και οι κυβερνήσει θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για να περιορίσουν τι αλληλεπιδράσει τη καπνοβιομηχανία και να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια αυτών των αλληλεπιδράσεων όταν υπάρχουν. Και οι κατευθυντήριες γραμμές ε, μιλούν στη συνέχεια για το γεγονό ότι τα μέρη θα πρέπει να έχουν σχέση με την καπνοβιομηχανία μόνο στο απολύτως απαραίτητο βαθμό προκειμένου να ρυθμιστεί ε, αποτελεσματικά η καπροβιομηχανία και τα προϊόντα καπνού. Είναι σαφέστατες λοιπόν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές. Και όποτε χρειάζονται κάποιες αλληλεπιδράσεις με την καπνοβιομηχανία θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε διαφανείς. Να γίνονται δημοσίως, ε, οι διαβουλευσει και να δημοσιεύονται και τα πρακτικά. Επίσης, ε, τα μέρη θα πρέπει να εφαρμόσουν ε, δεντολογικό κώδικα για τους υπαλλήλου με τι συγκεκριμένε προδιαγραφές θα πρέπει και τι προποθέσει που θα πρέπει να πληρεί κάποια μηχανία. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν αυτέ οι βέλτιστε πρακτικέ. και να δώσουμε εμεί το παράδειγμα προ μίμηση και στον υπόλοιπο κόσμο. Ποιε είναι λοιπόν αυτέ οι βέλτιστες πρακτικέ και τα διεθνή πρότυπα. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή ισχύουν κάποια μέτρα που εισήγαγαν το, Συμβούλιο και, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι ανεπαρκή για να τηρηθούν οι υποχρεώσει που απορρέουν από το άρθρο 5, παράγραφο 3 και μάλιστα είχαν θεσπιστεί πριν τη σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού. Χρειαζόμαστε ένα διδολογικό κώδικα α, για να διέπον, που θα διέπει τη σχέση με την καπνομηχανία, να ενημερωθούν οι διδολογικοί κανόνε και ε, να έχουμε σχέση ε, να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα κάποιων ε, ε, επιχειρήσεων συμβουλών και δημοσίων σχέσεων και επίσης να μην χρησιμοποιούνται μέλη της καπνοβιομηχανίας σε συμβουλευτικές επιτροπές για τον έλεγχο του καπνού. Επίσης, θα πρέπει πληροφορίες για την καταγραφή των λόμπι να είναι διαθέσιμες. Θα πρέπει να δημοσιεύονται επίσης ε, οι σχέσεις τέτοιου λόμπι με ε, ευρωβουλευτές και να τις δημοσιεύουν. Ε, οι πράσινοι έχουν δημοσιεύσει το σχετικό μητρό, για παράδειγμα. Επίσης, με βάση το άρθρο 5.3, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταγράφουν τις συναντήσεις τους με εκπροσώπους της καπνομηχανίας και μάλιστα όπου είναι δυνατό θα πρέπει να δημοσιεύονται και τα πρακτικά τέτοιων συναντήσεων για να εξασφαλίζεται διαφάνεια. Θεωρούμε ότι η καπνοβιομηχανία μπορεί να υποβάλει και γραπτό στι αιτήσει ε, στους αρμοδίους, ε, να ακούγεται φυσικά η φωνή τους, αλλά οι διμερείς επαφές θα πρέπει να πληρούν τη σύμβαση πλαίσιο της ΠΟΗ, δηλαδή να γίνονται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η σωστή ρύθμιση Τη καπνοβιομηχανίας και των προϊόντων καπνού. Αν υιοθετηθούν σαφείς κατευθυντήρες γραμμέ ε, για να τηρηθούν υποχρεώσει μα από την σύμβαση πλαίσιο τη ΠΟΗ, θα δείσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ε, υγεία των συμπολιτών και τη θεωρούμε ω υπέρτερο αγαθό σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα τη καπνοβιομηχανίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στη συζήτηση με τους συναδέλφους, ε, κυρίες και κυρίους. Η κυρία Παρβάνοβα πρώτη, παρακαλώ. Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας τα πω στη γλώσσα μου. Οπότε παρακαλώ βάλτε όλοι τα ακουστικά σας. Κύριε Πρόεδρε. τα κά сякаш индустрията има по-добри предложения как да бъдат ограничени съответно въздействието. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μεταφράστηκε η ομιλήτρια. Δεν μας είπε κανείς ότι δεν έχουμε ερμηνεία από τα βουλγαρικά. Μπορείτε να μιλήσετε βουλγαρικά, παρακαλώ. Shall I... Repeat from Να σας το επαναλάβω. Παρακαλώ, ναι, και δεν θα μετρήσουμε το χρόνο σας. Ξαναρχίστε παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους εμπειρογνώμονες, λέει η κυρία Παρβάνοβα, για τις παρουσιάσεις τους. Τι διαπιστώνουμε λοιπόν εμείς τελικώς. Έχουμε ένα πακέτο μέτρων το οποίο προσφέρουμε, το οποίο μάλλον είναι αναποτελεσματικό. Και από ό,τι φαίνεται η οικονομία, ο κλάδος ε, έχει καλύτερες μεθόδους και μέτρα να μας προτείνει. Υπάρχουν αποδείξεις ότι το κάπνισμα σκοτώνει. Και όχι μόνο σκοτώνει, θράψη κάνει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο πεθαίνουν χιλιάδες. <laughs> Θυμάστε τον καουμπόι του Μάλμπορο. Ε, έτσι, ε, πόσο κάπριζε και πέθανε μετά από 20 χρόνια. Και μόλις το 2002 η Φίλιπ Μόρις αναγνώρισε γιατί υποχρεώθηκε ότι πέθανε κάποιος λόγω των τσιγάρων που του πουλούσαν και μάλιστα υποχρεώθηκαν να καταβάλουν και ένα πρόστιμο αποζημίωση 280.000 ε, δολάρια. Ακούσαμε επίση ότι σε περιόδο οικονομική κρίσης είναι ένα περιττό έξοδο για τον καπνιστή, ε, ε, το κάπνισμα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ακούσουμε διάφορα μέτρα. Δεν ξέρω αν θα αρέσουν και στη βιομηχανία. Λοιπόν, να υποχρεθεί η βιομηχανία να καλύψει ένα τμήμα του κόστου των ιατρικών δαπανών ε, των καπνιστών για να δούμε πώς θα αντιδράσει ή γενικότερα του κόστους για τη δημόσια υγεία, για τα ασφαλιστικά ταμεία ή για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Ε, στη συνέχεια για τις προειδοποιήσεις. Είναι δυνατόν να υπάρχει, ορισμένοι προτείνουν να υπάρχει προειδοποίηση σε κάθε τσιγάρο, όχι στο πακέτο και να τα πληρώνει αυτά η βιομηχανία, όχι μόνο τη διαφήμιση. Ε, ακούστηκε λόγο, ε, έγινε λόγο συγγνώμη για αυτούς που χάνουν τη δουλειά τους. Μπορούν να μετεκπαιδευτούν και να εργάζονται αλλού και να τα πληρώσει η καπνοβιομηχανία. Επίσης, το κόστος ε, παραγωγής των προϊόντων καπνού θα πρέπει να το επομίζεται η ε, καπνοβιομηχανία και ε, σε περίπτωση που αλλάζουν προϊόντα επίσης. Ευχαριστώ κύριος Λίζε. Θα ήθελα να πω ξανά ότι υποστηρίζω την ουσία της πρότασης αλλά παρακαλώ η διαδικασία να είναι δίκαιη Ε, κάποια στιγμή ακούσαμε χειροκροτήματα. Ε, ε, λέμε συνήθως, Πρόεδρε, όμως ότι το κοινό απαγορεύεται να εκδηλώνεται. Θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία ανεξάρτητα με ποιον χειροκροτούν. Για το παθητικό κάπνισμα έχω να πω το εξή. Από πλευρά τη καπνοβιομηχανίας αμφισβητούνται τα στοιχεία για το παθητικό κάπνισμα. Ότι μπορούμε να μιλούμε και για κρούσματα θανάτου. Προσωπικά συμμετείχα σε μια μελέτη για τον ευνίδιο θάνατο των νεογνών. Και είναι σαφής η κατάσταση ότι ε, συνδέεται ο ευνίδιος θάνατος του νεογνού με το παθητικό κάπνισμα. Γιατί είμαι γιατρός και συμμετείχα σε τέτοιες έρευνες πριν ε, έρθω στο κοινοβούλιο. Κατά την άποψή μου υπάρχουν μερικά στοιχεία και θέλω να επαναλάβω την πρότασή μου για να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και ουσία στο παθητικό κάπνισμα. Δηλαδή, να μην μιλάμε για, ε, κατά 90% για την υγεία του καπνιστού, αλλά και για την υγεία των παιδιών και άλλων που εισπνέουν τον καπνό ανεξαρτήτως της ελίσεως τους. Και τα ξέρουμε τις προειδοποίησεις και τις ε, εικονογραφικές λεγόμενες και το κείμενο. Να ρωτήσω κάτι για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Να το ξεκαθαρίσω, το είπε και ο Πρόεδρος. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα προάγουν την υγεία. Αλλά άκουσα από πολλούς και πήρα και γράμματα που λέγουν ότι για μένα ήταν ο δρόμος να φύγω από το κάπνισμα, να το κόψω. Και ε, επιβαρύνω τουλάχιστον το περιβάλλον μου λιγότερο και τους παθητικούς καπνιστές. Ε, ε, και στην ηρωίνη, εγώ ήμουν, ήμουν διαφωνών, αλλά ε, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την έννοια της μείωσης του κινδύνου, harm reduction. Ας πούμε για την ηρωίνη μοιράζει σύριγγες, μοιράζει υποκατάστατα κτλ. Η κυρία Ζόμερ. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ για το ηλεκτρονικό τσιγάρο ακριβώ με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχω και άλλες ερωτήσεις, μην νομίζετε. Ε, η πρώτη ομιλήτρια, δεν θυμάμαι το όνομά σας, η κυρία Ποιτσκελάνγκε, ε, ε, μιλούσε συνέχεια για το δηλητήριο καπνό και τα άλλα δηλητήρια. Μα αν είναι δηλητήριο ο καπνός, είναι αλήθεια αυτό, είναι τόσο δηλητηριώδες. Και το, ρωτώ και τον κύριο από τον Καναδά, αν είναι τέτοιο δηλητήριο, γιατί δεν απαγορεύονται όλα τα προϊόντα καπνού. Τα πάντα. Και στον Καναδά. Αυτό δεν θα ήταν η συνέπεια αν είναι δηλητήριο καπνός. Ε, τότε μην κυκλοφορεί καθόλου στην αγορά αφού είναι τέτοιο δηλητήριο. Κυκλοφορεί όμως. Και ακόμα και σε που έχουν τις ε, πιο ισχυρές ε, ε, ρυθμίσει ως προς τι προειδοποιήσει και τα χαρακτηριστικά, υπάρχουν και κυκλοφορούν ακόμα προϊόντα καπνού. Μπορείτε να με διαφωτίσετε σχετικά. Ξέρω εγώ μήπως να το ξανασκεφτούμε. Και κάτι ακόμα. Έχω να ρωτήσω δεν θυμάμαι ποιος το είπε, νομίζω ο δεύτερος ομιλητής είπε ότι επηρεάζει οπωσδήποτε το πακέτο τη συμπεριφορά του καπνιστού και υπάρχουν ε, επαρκείς μελέτες που το στοιχειοθετούν. Μπορείτε να μας κάνετε ένα κατάλογο ποιες είναι αυτές οι μελέτες. Γιατί όλο μας λένε διάφοροι ότι έχουν γίνει μελέτες, έρευνες και δεν ξέρω ή κάποιος κάποτε κάτι. Μπορείτε να μου τα τεκμηριώσετε πολύ συγκεκριμένα και με τις μελέτες αυτές. Αλλιώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Και εγώ δεν συμφωνώ καταρχήν να χειροκροτούν οι θεατές, ε, το κοινό. Ναι, απαγορεύεται λέει ο πρόεδρος. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ της διαφάνειας. Ναι, ναι αλλά δεν το θεωρώ σωστό. Να το επιπλήτεται συγκεκριμένες συμπεριφορές. Είπα και εγώ ότι απαγορεύεται καταρχήν οποιαδήποτε εκδήλωση του κοινού έτσι μου το υπέδειξαν και εμένα και αυτή τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Εντάξει, ωραία. Επόμενος, ο κύριος Κουμουτσάκος, παρακαλώ. Ένα μισή λεπτό αν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο σημεία θέλω να θίξω τα οποία και τα δύο τα παίρνω από την εισηγητική έκθεση. Το πρώτο σημείο λέει το εξή η εισηγητική έκθεση. Ο γενικό στόχο αναθεώρηση τη οδηγία είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και βεβαίως να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Όλες οι ρυθμίσεις που βρίσκονται στην πρόταση βοηθούν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τη βελτιώνουν ή της δημιουργούν προβλήματα. Αυτό το λέει η συγκεκριτική έκθεση. Ο σκοπός είναι να βελτιωθεί η λειτουργία συγκεκριτική εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται σε αυτόν τον στρατηγικό στόχο της οδηγίας. Δημιουργούν προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Ξαναλέω λοιπόν ότι ψάχνουμε ένα μείγμα μεταξύ προστασίας της δημόσιας υγείας και της προστασίας της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Και είμαστε σε θέση, πιστεύω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς θρησκευτικού φανατισμούς, να βρει αυτή τη λύση. Δεύτερο σημείο. Πάλι από την εισηγητική έκθεση και τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση, λέει η εισηγητική έκθεση, εξαιρεί από ορισμένε διατάξει, όπω παραδείγματο χάρη την απαγόρευση προϊόντων με χαρακτηριστικά αρώματα, γεύσει, τα προϊόντα καπνού, που είναι διαφορετικά από τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά τσιγάρα και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, δηλαδή πουρα, πουράγια κλπ. Και αυτή την εξαίρεση την θεμελιώνει στο γεγονός ότι αυτή η χρήση γίνεται από συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών και ουσιαστικά δεν αφορά τους νέους. Γι' αυτό τα επιτρέπουμε ως εξαίρεση. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε, να ρωτήσω όλους τους συναδέλφους. Έχουμε δει νέα παιδιά να καπνίζουν slim τσιγάρα στις χώρες σας έχετε δει και ποιες είναι οι έρευνες που το επιβεβαιώνουν αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Oh, one and a half please. Thank you, Chairman. κύριε um, Πρόεδρε, σίγουρα θέλουμε να μειωθούν οι καπνιστές. Είναι κάτι πολύ κακό για την υγεία και το επιβεβαιώνω γιατί εγώ κάπνιζα και δεν είναι εύκολο να το κόψει κανείς, αλλά όταν το κόψει κανείς τότε είναι κανείς σαν να κάπου φυλακισμένος και να είναι ξαφνικά ελεύθερος. Επομένως, 100% συμφωνώ και σήμερα η συζήτηση ε, μου άφησε δύο ερωτήματα. Δεν θέλω να κάνουμε κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε αποτελέσματα που δεν τα θέλουμε. Θέλω να κάνουμε το σωστό. Ακόμα. Δεν έχω καταλάβει τι ισχύει, τι γίνεται με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Να δούμε. Σε σχέση με αυτά που στο τέλος ακούσαμε, γιατί ας πούμε ναι, τι έγινε, πώς, μπορεί να ληφθεί υπόψη η καναδική εμπειρία για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Επομένως, εάν συμβάλλουν στο να κόψουν στο κάπνισμα, μην κάνουμε κάτι που δεν το οδηγήσει δεν τα αποτελέσματα, δεν είμαι σίγουρη. Τώρα όσον αφορά τη συσκευασία, το πακέτο, το αποτέλεσμα στο λαθρεμπόριο, η διαφήμιση πώς επηρεάζει τους νέους και εάν χρειάζεται τότε να υπάρχει χώρος πάνω στο πακέτο που να έχει μήνυμα να προοδοποιεί για το ελάθρο εμπόριο γιατί τελικά είναι σίγουρο ότι τα δηλητρία τσιγάρα είναι πολύ πιο βλαβερά από αυτά που είναι νόμιμα. Σας παρακαλώ, μία ερώτηση να κάνετε, όχι τοποθετήσεις, δεν θα έχουν το χρόνο να απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες στις ερωτήσεις. Chris Davis, η κυρία Κονή. Uh, just When... Ένα μικρό μάθημα ιστορίας. Όταν έσπεσε κατά πρώτη, πρώτη φορά πριν από μια δεκαετία που αυτή την νομοθεσία, δεν υπήρχε πρόταση για φωτογραφίες προειδοποιητικές. Αυτό προήλθε από το Κοινοβούλιο, που σε συνάδελφους άλλους και από τον ομιλούντα, απερίφθη από το Κοινοβούλιο τελικά και τελικά υπήρχε διακομιτική συμφωνία που λέγανε όλες οι παρατάξεις ότι μπορούν να το κάνουν τα κράτη-μέλη και πέρασε τελικά εκείνη η πρόταση στι 3 η ώρα το, το, το ξημόραμα. ξημέρωμα. Την τελευταία συνάντηση τη της, ε, ε, και είπαμε ότι δίνονται τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν σχετική νομοθεσία. Επομένω, συμφωνήσαμε, παρακάμψαμε την Κομισιόν και είχαμε μια συνέντευξη τύπου και τα τρία όργανα ε, μίλησαν στον τύπο και είπε τελικά, αφού έξι μήνες είχε στυλώσει τα πόδια, η Κομισιόν είπε ότι συμφωνεί. Και το ερώτημα τώρα είναι, όσον αφορά τα στοιχεία, τι αποδείξει που υπάρχουν, εγώ κατέβασα ε, πρώτα για αυτά τα μέτρα, οπότε βεβαίω και θέλουν να έχουν αποτέλεσμα και κυρίω για να μην, ε, για να αποτρέπουν τους νέους να αρχίζουν το κάπνισμα και ε, λέει η καπνοβιομηχανία ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτού του είδου προειδοποίησει έχουν αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά μα λένε το αντίθετο. Μπορεί κάποιο να απαντήσει. Έχουν ή δεν έχουν αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, Κρίς, λέει ο πρόεδρο. Και κύριε Όκονη έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε για αυτή την ε, ακρόαση που είναι τόσο ενδιαφέρουσα. Και Προσωπικά μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα τέτοιο νομοθέτημα να δείξει τόλμη. Να δείξει τόλμη διότι όλοι γνωρίζουμε, όπως και επανειλημμένα ακούστηκε σήμερα, ότι έχουμε ότι 750 θανάτους ετησίως, 5 εκατομμύρια, χιλιάδες, εκατομμύρια στον κόσμο, 50.000 στην Ευρώπη που δεν καπνούν, δεν καπνίζουν και πεθαίνουν από το παθητικό κάπνισμα και Πρόκειται για κάποια αριθμητικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Θεωρώ ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα θαραλέο νομοθέτημα πρόκειται να προβληθεί, να έχει να προβληθεί μια θετική εικόνα της και επομένως θα πρέπει αυτό να προσέξουμε. Οι ανήλικοι με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε θα πρέπει να προειδοποιηθούν. Εγώ έχω τέσσερα παιδιά και δύο από αυτά καπνίζουν. Και πάω στο σχολείο όταν μπορώ να βλέπω όλα αυτά τα παιδιά που καπνίζουν και δηλητηριάζονται. Γιατί θέλουν να μιμηθούν το γκολιτό τους. Οπότε όλα αυτά τα οποία βάζουμε πάνω στη συσκευασία, όλα αυτά τα μηνύματα δεν αρκούν. Ποιο είναι το κρίσιμο, ποιο είναι το αποφασιστικό, ούτως ώστε τα παιδιά να μην συνηθίζουν το καπνίσμα. Θα πρέπει να αυξήσουμε το, το μέγεθος, να υπάρχει διαπαιδαγώγηση, να έχουμε αυτά τα πάτσο, αυτά τα αυτοκόλλητα νοικοτήνης, που βοηθούν πάρα πολύ να κόψει κανείς το κάπνισμα. Ο κύριος Φλόρενς. Ναι. Η ενημέρωση για το θέμα του καπνίσματος είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Είπατε ε, και θέσατε ως σημαντικό επιχείρημα την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τα λοιπά, το νόμιμο εμπόριο. Εγώ διάβασα τώρα πολύ σοβαρές μελέτες που λέγουν ότι τα λαθρέα τσιγάρα κατά 50% και πλέον προέρχονται από νόμιμους παραγωγούς, από την ε, ουδέτερη ε, πόλη της Αγίας Πετρούπολης και βρίσκουν το δρόμο ε, της παρανομίας μέσω της νομιμότητας. Δηλαδή αν παράγονται νόμιμα τα τσιγάρα σε εσά και μετά κυκλοφορούν λαθρέα, αυτό είναι κόλαφος για οποιοδήποτε πολιτικό ε, ασχολείται με τη δημόσια υγεία. Καρσούτερ, σύντομη ερώτηση μου. Προς τον David Hammond θα ήθελα να υποβάλω την ερώτηση. είπατε ότι ήσασταν και σύμβουλος κυβερνήσεων. Η καπνοβιομηχανία ισχυρίζεται ότι να χρησιμοποιεί κανεί ένα λιτό πακέτο χωρίς το εμπορικό σήμα είναι παράνομο, παραβιάζει τα δικαιώματα τέτοιων καπνοβιομηχανιών. Με ποιο επιχείρημα θα καταρρύψετε αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ. Απευθύνθηκε άμεσα ερώτηση στον εκπρόσωπο της βιομηχανίας. Ε, σύντομα να μας απαντήσει και μετά οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Εννοείται την ερώτηση του κυρίου Φλόρενς, λέει ο κύριος Ρέρινγκ. Ε, μπορώ να είμαι πολύ σύντομος. Το λαθρεμπόριο εμάς μας πλήττει. Έχουμε συμφωνία, τα μέλη μας δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει αυτών των όρων της συμφωνίας Εάν το προϊόν μας που πωλείται στη Ρωσία, όπως είπε ο κύριος Φρόνης, κατασχεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς πληρώνουμε πρόστιμα. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί πέντε ως πρόστιμο. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ σαφές κίνητρο πέρα από το εμπορικό και επιπλέον το εμπορικό να ε, προλάβουμε αυτές και να αποτρέψουμε αυτές τις πρακτικές. Και το εμπορικό κίνητρο είναι οτιδήποτε ε, πολύ λαθρέα δεν πάει στη δική μας τσέπη καταρχήν. Ευχαριστώ. Λέω ο Πρόεδρος. Με τη σειρά τώρα απαντήσετε. Παρακαλώ. Yes. Ευχαριστώ. Έχω πολλά σχόλια. Θα προσπαθήσω να τα αναφέρω επιγραμματικά για να αφήσω και τους άλλους καλεσμένους. Ο κύριος Λίζε μίλησε για το παθητικό κάπνισμα. Φυσικά εκεί είναι που προσπάθησε η καπνοβιομηχανία να στρεβλώσει τα επιστημονικά απορίσματα και να εμποδίσει τι ε, κυβερνήσει που ήθελαν να υιοθετήσουν πιο αυστηρά μέτρα. Αλλά πολλέ χώρε ήδη έχουν ε, ε, μέτρα απαγόρευση του καπνίσματο. και θα πρέπει να το γενικεύσουμε αυτό για να προστατεύσουμε και τα παιδιά. Γιατί αυτά είναι τα πρώτα θύματα του παθητικού καπνίσματο. Βέβαια, η οδηγία για τα προϊόντα καπνού δεν ασχολείται κυρίως με το θέμα αυτό, αλλά επίση είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, φαντάζομαι θα το σχολιάσω και οι συνάδελφοι, αναγνωρίζουμε ότι πολλοί κόσμος λέει ότι τους βοηθάνε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα για να περιορίσουν ή να σταματήσουν το κάπνισμα. Αλλά τέτοια ε, προϊόντα με νοικοτήνη χωρί καπνό να εμπίπτουν στην οδηγία για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Στην, Ηνωμένε ΗΠΑ προβλέπονται δύο διαβουλεύσει για το θέμα αυτό και με ενδιαφέρον περιμένουμε την έκβασή του. Πάντω, το, ο μα μας προβληματισμός είναι να είναι μπροστά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε αυτού που τα επιθυμούν, αλλά να μην κυκλοφορούν στην αγορά ελεύθερα για να προσελκύσουν και νέου ή να αποτρέπουν το σταμάτημα του καπνίσματο. Ε, είναι σημαντικό θέμα των ηλεκτρονικών τσιγάρων, αλλά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτήν την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Και η ΠΟΗ ζήτησε περισσότερε μελέτε και έρευνε για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τα τσιγάρα slim, τα πολύ λεπτά, υπάρχουν αποδείξει, ρώτησε κανεί κάποιο. Ναι, φυσικά υπάρχουν αδιάσπαστα, στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λένε μερικά κορίτσια ότι θεωρούν τα πακετάκια αυτά πολύ πιο δελαστικά γιατί μοιάζουν ε, ότι δεν είναι πακέτα τσιγάρο μοιάζουν με συσκευασίε ε, καλλιντικών ε, ή ε, αρώματος. Μερικές φορές έχουν και λουλουδάκια πάνω. Έχουν ως κοινό στόχο τα νερά κορίτσια. Όντως πιάνει αυτή η παραπλάνηση. Γι' αυτό θέλουμε να απαγορευτούν πλήρω αυτά τα πολύ λεπτά τσιγάρα. Κάποιος μίλησε για τα παραπημένα τσιγάρα και ότι θεωρού, θεωρείται ότι είναι πιο επιβλαβή από τα αγνήσια, τα αυθεντικά. Τα αγνήσια τσιγάρα, τα αυθεντικά, έχουν γύρω στου 70 καρκινογόνους παράγοντες και σκοτώνουν ένα στου δύο χρήστε, ένα στου δύο καπνιστέ μακροπρόθεσμα. Και δεν νομίζω ότι ένα παραποιημένο τσιγάρο θα ε, είναι πιο επιβλαβές, θα σκοτώσει με ταχύτερο ρυθμό από ένα γνήσιο αυθεντικό τσιγάρο. Ευχαριστώ να απαντήσω στα, ε, σχόλια στις ερωτήσει όσον αφορά το παθητικό κάπνισμα. Εδώ υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει συνειδητοποίηση, αλλά όχι τόσο πολύ και οι ρυθμικές αρχές, προσπαθούν να δουν πώς θα προειδοποιήσουν τον κόσμο και έχουμε περίπου 12 στήρες που συνδέονται με το κάπνισμα και υπάρχει συνένεση από τι αρχέ τη υγεία και τι δημιουργικές αρχέ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα το παθητικό κάπνισμα σε σχέση επίση με τα SLIM. Πώ ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα στοιχεία. Αυτά που μου λέει η καπνοβιομηχανία όσον αφορά την αύξηση των πωλήσεων είναι γεγονό. Αυξήθηκε η πωλήση των, των SLIM για την καναδική αγορά. Έχουμε ένα πολύ διάζων νομοθετικό πλαίσιο, οπότε έχουμε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νοικοτήνη απαγορεύονται. Έχουμε, πολλούνται τέλο πάντων και αυξάνονται οι, οι προτίμηση του κοινού σε αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά χωρί νοικοτήνη. Ακόμα πάντω ε, θα τελειοποιήσουμε περισσότερο ε, την ε, μαθησία μα τώρα όσον αφορά τι απομιμήσει και το λαθρεμπόριο. Από ό,τι γνωρίζω η καπνομηχανία έχει αυτό το επιχείρημα για να μην υπάρχουν οι προδοποίησεις και οι φωτογραφίες λέγοντας ότι με αυτές τις προδοποίησεις αυξάνεται το λαθρεμπόριο. Εγώ δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Εμείς τα έχουμε πάνω από μία δεκαετία. Ε, αυτού του είδου τα, τα πακέτα προειδοποίηση. Και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό που λένε οι καμπνοδομήχανοι. Επίση, υπάρχει ε, μια, μια λίστα από όλε αυτέ τι μελέτε που σα ανέφερα. Ναι, έχω ένα κατάλογο και να διαβιβάσω το κατάλογο σε όποιον θέλει. Αυτό το οποίο είπατε ε, μα οδηγεί σε κάτι σημαντικό, ότι θα πρέπει να είναι τα στοιχεία ε, δημόσια, θα πρέπει να είναι αξιοποιημένα αξιόπιστα και θα πρέπει να ελέγχονται από τους ε, επιστήμονες και γι' αυτό και θα σας δώσω ό,τι στοιχεία έχω. Επίσης, άλλη ερώτηση. Υπάρχει κάποια διαφορά ε, για την, αποτελεσμα... για την αποτελεσματικότητα των προεδοποιήσεων και τελικά ό,τι σας είπα σήμερα το στήριξα με δημοσιεύσεις και επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Η καπνοβιομηχανία, ό,τι στοιχεία είχε, τα είχε από κάποιους που μάλιστα τα στοιχεία που παρουσίασαν, αφού τους πλήρωσε η ίδια καπνοβιομηχανία. Άρα, ευχαριστούμε κύριε Γιώσενς. Θα πρέπει να απαντήσω σε τρία ζητήματα. Πρώτον, το θέμα του λαθρεμπόριου, της απομίμησης. Ε, ανησυχία που ακούσαμε σχετικά. Σε σχέση με αυτό, Έχουμε ένα ε, χαρακτηριστικό ασφαλείας ορατό, αλλά είναι εύκολο αυτό να παραποιηθεί και θα σας συμβούλευα να υπάρχουν και αόρατα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Δηλαδή, ε, Αυτό θα ήταν ένας τρόπος να γίνει πιο δύσκολη ακόμα η ε, απομίμηση. Η χαρακτηριστικά όρατα, λοιπόν, ό,τι φαίνεται αντιγράφεται. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των προειδοποίησεων υγεία, να σα πω κάτι για το Βέλγιο. Ήταν η πρώτη χώρα που εισήγαγε αυτό το θέμα, το 2007, φωτογραφίες δηλαδή, εικονογραφικές προειδοποίησεις. Έχουμε τα στοιχεία επιπολασμού για 10.000 πρόσωπα από το Επιστημονικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και το 1997 ήταν 30%, στη συνέχεια το 2029 το 2004-28 οι φωτογραφίες ε, εισήχθησαν το 2007 και ο πυπολασμός έπεσε στο 25% το 2008. Τι σημαίνει αυτό. Σε τέσσερα χρόνια μείωση κατά 3% και στο ποσοστό των καπνιστών 10%. Τα στοιχεία λοιπόν ε, δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικά στο Βέλγιο το τελευταίο για το πώς συμμετέχει η JTI στο λαθρεμπόριο. Το 2001 έγινε μια μεγάλη καταγγελία με διάφορα email και για τη συμμόρφωση δεν ε, ευθυγραμμίστηκαν με την πολιτική της μηδενικής ανοχής λαθρεμπορίου. Επανειλημμένα και ειδικά παραβιάζει τις υποχρεώσεις ε, με, ε, της συμφωνίας που συνήψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος της παράθεσης. Η δόκτωρ Μαρτίνα Πέτσχε παρακαλώ. Επειδή ερώτηση έγιναν από δύο Γερμανούς ευρωβουλευτές, ε, θα ήθελα να απαντήσω στα γερμανικά. Η κυρία Ζόμερ ρώτησε για τα στοιχεία για το παθητικό κάπνισμα. Μπορώ να σας καθησυχάσω. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο που δείχνουν ε, ε, πώς απειλείται η υγεία των παθητικών καπνιστών. Ε, την περιγράφουν πάρα πολύ καλά και τεκμηριώνουν και με στοιχεία και είναι στη διάθεσή σας και εμείς έχουμε εκδώσει αντίστοιχη έκθεση. Τη δεύτερη ερώτηση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Νομίζω και οι δύο βουλευτές ρώτησαν τι έχω να πω γι' αυτό. Δημοσιεύσαμε στο περιοδικό των Γερμανών ιατρών ε, μία μελέτη ε, που ε, χαρακτηρίζουμε ομιχλώδες αυτό το, νεφελώδες αυτό το προϊόν, γιατί πραγματικά εκπέμπει κάτι σύννεφα ατμού και είναι νεφελώδες γιατί δεν ξέρουμε τι έχει μέσα αυτό το προϊόν. Δεν είναι ένα προϊόν που έχει οριμάσει, δεν υπάρχουν στάνταρ και προδιαγραφές οριμότητας. Υπάρχουν δοδε... Κάδες, ε, ε, εφαρμογών με διάφορα φιαλίδια που τα περισσότερα έχουν νικοτίνη ε, από ανεύθυνα υψηλές ε, σε μεγάλο βαθμό ε, συγκεντρώσεις και ο κάθε καταναλωτής μπορεί να διαλέξει το φιαλίδιο νικοτίνης και να το αναμίξει και έρχεται στην κουζίνα και μπαίνει κάποιο στοιχεία και το παίρνει και το ανακατεύει με το φαγητό. Μα η νοικοτήνη είναι φωνικό όπλο. Όλα αυτά που λέγουν οι κατασκευαστές του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι πάρα πολύ επικίνδυνα σε ό,τι αφορά το ίδιο το προϊόν για τι επιπτώσεις στην υγεία αυτή καθ' αυτή. Ε, αλλεργίες, ενοχλήσεις στο αναπνευστικό, το λέγουν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, αλλά και δηλητηρίαση από την οικοτίνη όταν οι καταναλωτές ε, ρουφούν πάρα πολύ έντονα αυτό το τσιγάρο, γιατί δεν έχουν έλεγχο στο ηλεκτρονικό τσιγάρο ε, και κάποια στιγμή υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση από νοικοτήνη του οργανισμού και μπορεί κανείς να καταρρεύσει με πραγματικά δηλητηρίαση από νοικοτήνη. Αυτά. Ναι, γιατί θα μας φύγουν οι διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Ε, να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, τη Λίντα Μακάβαν, ε, για να συνοψίσει και να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. thank you, Ευχαριστώ. Δεν έχω να πω και πολλά γιατί είχαμε πραγματικά ένα πολύ μεστό απόγευμα ε, πλήρες ε, ομιλιών και παρεμβάσεων. Σας ευχαριστώ, τα σημείωσα προσεκτικά όλα και έχουμε πολύ τροφή για σκέψη και συζήτηση, αποδείξεις, ε, ανταποδείξεις. Ακούσαμε και για τη σύμβαση πλαίσιο της ΠΟΗ. Εγώ θα συναντήσω συγγήτρια εκπροσώπους του κλάδου θα σας δημοσιεύσουμε τις ημερομηνίες των διαβουλεύσεων. Θα γίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα γνωρίζετε πότε ακριβώς θα γίνουν. Ακούσαμε λοιπόν τις ανησυχίες σας ως προς την ανάγκη εφαρμογής της Σύμβασης Πλαισίου. Άκουσα πολύ προσεκτικά και τα σχόλια των συναδέλφων και θεωρώ ότι είναι πολύ υπεύθυνη η στάση των συναδέλφων και υπέβαλαν πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Φαντάζομαι ότι όλοι οι συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν μια νομοθεσία που θα βελτιώνει τη δημόσια ηχεία και θα αποτρέπει τους νέους από το κάπνισμα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία, για τη συζήτηση και είμαι βέβαια ότι θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Γιατί έχουμε χρόνο για μια κανονική, ομαλή ε, κοινοβουλευτική διαδικασία, προκειμένου κατά τη διάρκεια της δική μα κοινοβουλευτική θητεία να εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα. Ευχαριστώ όλους του συμμετέχοντες, όλους τους εμπειρογνώμονε που μας έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε και να κάνουμε τις ερωτήσεις μας κυρίως ε, και να πάρουμε απαντήσεις. Πολύ ε, χρήσιμα όλα αυτά, πολύ ωφέλιμα για μας. Τώρα εναπόκειται σε μας να περάσουμε αυτή την νομοθεσία από το Κοινοβούλιο, αλλά και το Συμβούλιο καλείται να δράσει. Ε, δεσμεύτηκε σήμερα ο υπουργό ότι αυτή η νομοθεσία ε, θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις ευρωεκλογέ και θα θέσει και ένα ορόσημο στην πολιτική δημόσια υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαραίτητο αυτό το ορόσημο κατά τα άλλα, χρειάζονται πιο αυστηροί κανόνες για να αρχίζουν να καπνίζουν όσο γίνεται λιγότεροι ε, αυτή είναι η δουλειά μας. Έχουμε μια εισηγήτρια η οποία ακούει πάρα πολύ προσεκτικά και είναι σε θέση να φέρει σε αίσιο πέρα σε αυτή την νομοθεσία. Ευχαριστώ όλους τους παρόντες και σας εύχομαι καλή επάνωδο και καλό σας βράδυ. Αύριο 9.30 ώρα συνεχίζεται η Επιτροπή μας για τους συναδέλφους. Γιατί ψηφίζουμε.